Σί, Καλησπέρα σα. Κυρίσω την επανάληψη των εργασιών τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τη Ολομέλεια που ε, διεκόπη στι 19 Ιουνίου. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να καλωσορίσω την ε, Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγγελα Μέρκελ, και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Ούρσουλα Φόντερ Λάιον, που βρίσκονται μαζί μας σήμερα εδώ στην αίθουσα της Ολομέλειας. Τα πρακτικά των συνόδων 17ης, 18ης και 19 η Ιουνίου 2020 έχουν εγκριθεί και μοιραστεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί έχουν μοιραστεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι, οπότε και τα πρακτικά εγκρίνονται. Δύο ανακοινώσεις. Διάφορες επιτροπές αποφάσισαν να ε, ε, με βάση το άρθρο 171 του στερικού κανονισμού να αναβάλουν ε, την, την έναρξη των διαπραγματεύσεων και οι εκθέσεις που περιέχουν την εντολή για την έναρξη των διαπραγματεύσεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης με τους τίτλους τους. Ένας αριθμός ευρωβουλευτών ή περισσότερες κοινοβουλευτικές ομάδες ε, με το ελάχιστο κατόφλι μπορούν ε, μέχρι την πέμπτη ε, με τις 12 τα μεσάνυχτα να αποφασίσουν, να ζητήσουν την ψηφοφορία στο Κοινοβούλιο για την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αν δεν υποβληθούν εγκαίρως τέτοια αιτήματα θα θεωρηθούν συγκεκριμένε οι αιτήσει αυτές. Επίσης δεν έχουμε λάβει αντιρρήσει ό,τι αφορά τη σύσταση τη επιτροπή ΕΚΟΝ να μην αντιταχθεί σε μια κατεξοδότηση πράξη δυνάμει το άρθρο 111 παράγραφος 6 του εσωτερικού κανονισμού. Η σύσταση αυτή περιέχεται στη, στην ιστοσελίδα της Ολομέλειας. Αν μέχρι τα μεσάνυχτα καμία πολιτική ομάδα ή ελάχιστος αριθμός ευρωβουλευτών ε, ε όπως προβλέπετε στο κατόφλι δεν ε, ψηφοφορία θα θεωρηθεί εγκεκριμένη η σύσταση αυτή. Δεν θα διεξαχθεί ψηφοφορία. Περνάμε στην ημερήσια διάταξη. Το τελικό σχέδιο ημερήσια διάταξη που εθετήθηκε από τη διάσκεψη των Προέδρων στι 2 ε, του Ιουλίου με βάση το άρθρο 157 έχει μοιραστεί. Και επίσης θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχω λάβει δύο αιτήματα κατεπίγουσας διαδικασίας με βάση το άρθρο 123 του εσωτερικού κανονισμού για να προσθέσουμε τα εξή νομοθετικά κείμενα στην, στη Σύνοδο μας. Καταρχήν, μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο αντίκτυπος ε, της ε, κρίσης COVID-19 κατόπιν ε, η διεξαγωγή κλινικών δοκιμών σε ό,τι αφορά τις, τους γενετικώς τροπημένους οργανισμούς για τα φάρμακα και επίσης η παροχή ε, θεραπείας ιατρικής για το COVID. Και αυτά τα, αυτές οι συστάσεις θα, θα υποβληθούν σήμερα για ψηφοφορία. Μπορούμε να ακούσουμε τους ε, ε, ετούντες ή μια, έναν ευρωβουλευτή κατά του αιτήματο αυτού. Θέλει κανείς το λόγο για τις μεταβατικές διατάξεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19. Δεν βλέπω να ζητά κανείς το λόγο. Θέλει κανείς το λόγο για την κατεπήγουσα διαδικασία σε ό,τι αφορά τη διεξαγωγή κλινικών δοκιμών με φάρμακα. Η κυρία Κόνετσνα είναι κατά του αιτήματο αυτού κατεπήγοντος. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η QNGL. Ε, θεωρούμε ότι ε, δυνάμει της κρίσης μπορούμε να κάνουμε μια εξαίρεση από την αυστηρή προσέγγιση που έχουμε για τους ε, γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Αλλά η ε, ευελιξία αυτή δεν είναι απεριόρεξη και για να αποφύγουμε κατάχρηση των παρεκκλήσεων στις, στην νομοθεσία για τους γενετικώς ιστοποιημένους οργανισμούς θα πρέπει αυτή η παρέκκληση να περιορίζεται μόνο στα εμβόλια και η προτινόμενη παρέκκληση θα πρέπει να είναι χρονικά οριοθετημένη και περιορισμένη. Επίσης, μπορεί να καθυστερήσει η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για χρόνια ολόκληρα. Οπότε, στο μεταξύ, οι δυνητικοί κίνδυνοι για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία θα εξακολουθούν να υπάρχουν. Επίση, ε, το κοινό θα πρέπει να ενημερώνεται ότι χρησιμοποιούνται γενετικώ τροπημένοι οργανισμοί στι δοκιμέ. Επίση, ε, Ζητείται παρέκκληση από την νομοθεσία για του γενετικώ τροπημένου οργανισμού και την αδειοδότηση για αυτού, χωρί προηγούμενη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το αίτημα αυτό είναι ανεύθυνο και δυσανάλογο. Οπότε θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους να καταψηφίσουν ε, την αίτηση αυτή για τη χρήση της κατεπίγουσας διαδικασίας για τις ε, κλινικές αυτές δοκιμές με φάρμακα που περιέχουν και γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Τώρα, σε σχέση με την πρόταση αυτή ε, και τις προτάσεις για την τροποποίηση ημερήσεις διάταξης, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των που έχουν υποβληθεί για ξεχωριστές και κατατμήματα ψηφοφορίες θα έχουμε ε, πολλούς γύρους ε, ψηφοφοριών. Σε ό,τι αφορά τι διάφορε ψηφοφορίε, έχετε τι σχετικέ πληροφορίε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για το δεύτερο γύρο την Παρασκευή θα γίνει, 14, ε, γίνει στις 2 και 4 με 3,5. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της δεύτερης αυτής ψηφοφορίας θα λάβει χώρα στις 6 το απόγευμα. Η τρίτη ψηφοφορία της Παρασκευής ακυρώνεται. Υπάρχουν αντιρρήσεις, όχι. Οπότε εγκρίνονται οι αλλαγές αυτές. Τώρα σε ό,τι αφορά τις ε, ηλεκτρονικές πληροφορίες για τη μεταφορά εμπορευμάτων, πρόταση του Συμβουλίου. Δεν έχει υποβληθεί πρόταση απόρριψης της πρότασης του Συμβουλίου, ούτε έχουν κατατεθεί τροπολογίες δυνάμει των άρθρων 67 και 68 του εσωτερικού κανονισμού. Οπότε η προτινόμενη αυτή πράξη εγκρίνεται. Τώρα, η μερίσια διάταξη προβλέπει δήλωση του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, με θέμα την παρουσίαση του προγράμματος της Γερμανικής Προεδρίας. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι δεν προβλέπεται διαδικασία ούτε catch the eye, ούτε υποβολή ερωτήσεων με την μπλε κάρτα. Θα δώσω το λόγο στην καγκελάριο Μέρκελ, παρακαλώ. Αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι, ε, ευρωβουλευτές, ε, κυρίες και κύριοι. Είναι χαρά για μένα η ευκαιρία που έχω να μιλώ ε, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην αρχή της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Όπως οι περισσότεροι από εσά, έτσι και εγώ νιώθω ότι μου λείπει η επαφή με κόσμο, έτσι κατηδίαν και αυτοπρόσωπη παρουσία. Και έρχομαι ε, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας ε, σε αυτούς τους καιρούς όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να ξεπεράσει την κρίση ενισχυμένη και χρειάζεται για αυτό το σκοπό το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι τεράστιες οι αποστολές ε, που έχουμε και χρειάζονται τεράστιες προσπάθειες. Με κοινοβουλευτική αντιπαράθεση, με πολιτική διαμεσολάβηση, με πολιτιστική μετάφραση στις διάφορες χώρες και περιφέρειες. Και γι' αυτό χρειάζεστε εσείς και σας χρειάζεται η Ευρώπη. Και για μένα είναι ιδιαίτερη τιμή η ευκαιρία που έχω σήμερα να σας παρουσιάσω τις βασικές προτεραιότητες της Γερμανικής Προεδρίας. Για μένα είναι πέντε τα σημαντικότερα θέματα. Τα θεμελιώδη μας δικαιώματα, η συνοχή μας, η προστασία του κλίματος, η ψηφιοποίηση και η ευθύνη της Ευρώπης στην Ιφίλιο. Αυτά τα πέντε θέματα είναι σημαντικά διότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε την Ευρώπη με βιωσιμότητα, αν θέλουμε να την προστατεύσουμε και να τη διαφυλάξουμε. Μόνο τότε η Ευρώπη ε, σε ένα παγκόσμιο ε, σύστημα και μια τάξη που αλλάζει ραχδαία θα μπορεί να είναι κυρίαρχη και υπεύθυνα να αναλάβει το ρόλο που της αναλογεί. Γνωρίζω ότι σήμερα η επίσκεψή μου συμπίπτει με την μεγαλύτερη πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πανδημία, παγκόσμια πανδημία κορονοϊού ε, χτύπησε σφοδρά και ανελαίητα ε, τους ανθρώπους και στην Ευρώπη. Και μόνο στην Ευρώπη έχουμε 100.000 και πλέον νεκρούς που θρυνούμε και πολλοί πολίτες, άνδρες και γυναίκες, δεν μπόρεσαν ούτε καν να αποχαιρετήσουν τους δικούς τους όταν έφευγαν από τη ζωή τις τελευταίες ώρες λόγω των αυστηρών μέτρων και της καραντίνας. Αυτό δεν θα πρέπει να το λησμονούμε. Είμαστε βέβαια ε, υπέρ της ανάκαμψης και της οικονομικής, αλλά δεν θα πρέπει να ξεχνάμε το πένθος για τους νεκρούς, το θρήνο ε, θα εξακολουθήσει να μας συνοδεύει για πολύ καιρό ακόμα αυτή η εικόνα των ανθρώπων που δεν μπόρεσαν να αποχαιρετήσουν τους ε, δικούς τους και η οικονομία επέστη σφοδρή επίθεση και συντριβή. Κατομμύρια έχασαν τις ε, δουλειές τους. Ανησυχούν εκτός από την υγεία τους και την υγεία των οικογένειών τους και τώρα περισσότερο ανησυχούν και για την ίδια τους την οικονομική επιβίωση. Όλοι αυτοί χρειάζονται τώρα την δική μας κοινή υποστήριξη. Για να σπάσουν οι αλυσίδες μετάδοσης χρειάστηκε προσωρινά να περιοριστούν και τα πιο βασικά θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό ήταν πολύ μεγάλο τίμημα, γιατί για αυτά τα θεμελιώδη δικαιώματα αγωνίστηκαν σκληρά γενιές ολόκληρες στην Ευρώπη. Οι άνθρωποι και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι το πιο πολύτιμο αγαθό που έχουμε στην Ευρώπη. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα ε, πολιτικά δικαιώματα θα πρέπει να περιορίζονται πάντα με αυστηρά κριτήρια και η πανδημία να μην είναι ποτέ πρόφαση για εξουδετερώση της δημοκρατίας. Κάθε χώρα της Ευρώπης έχει διαφορετικές ιστορικές εμπειρίες. Έχει διαφορετικούς αγώνες δώσει για το κράτος δικαίου και την ελευθερία. Ταυτόχρονα όμως αυτή η κατάκτηση των θεμελιδών δικαιωμάτων μας ενώνει στην Ευρώπη. Προσωπικά έχω περάσει 35 χρόνια από τη ζωή μου σε ένα σύστημα ανελευθερίας. Ο περιορισμός αυτών των δικαιωμάτων στην πανδημία λοιπόν για μένα ήταν μια απόφαση την οποία δυσκολεύτηκα απίστευτα να πάρω. Σε αυτή την ιστορική φάση λοιπόν αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης η Γερμανία με γεμίζει σεβασμό και με πολύ πάθος ε, αυτή η αποστολή μου και το καθήκον, γιατί εγώ πιστεύω στην Ευρώπη. Είμαι ε, πεπισμένη Ευρωπαία, όχι μόνο ε, ως ανάμνηση στο παρελθόν αλλά και ως ελπίδα για το μέλλον. Η Ευρώπη δεν είναι μια κληρονομιά, ε, κάτι μοιραίο το οποίο μας υποχρεώνει για κάτι. Όχι, η Ευρώπη είναι κάτι το ζωντανό που μπορούμε να διαμορφώνουμε και να αλλάζουμε. Η Ευρώπη δεν μας αφαιρεί δυνατότητες δράσης, αλλά σε μια παγκοσμιοποιημένη πραγματικότητα μας δίνει, κάνει η Ευρώπη τη δυνατότητα της δράσης δεν γίνεται χωρίς την Ευρώπη, αλλά μόνο με την Ευρώπη να διατηρήσουμε τις πεπιθήσεις και τις ελευθερίες μας. Και γι' αυτό χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ να προσανατολιζόμαστε στα θεμελιώδη δικαιώματα, αλλά και να υποστηριζόμαστε και να έχουμε κοινή αλληλεγγύη και συνοχή. Γιατί η Ευρώπη θα παραμείνει Ευρώπη μόνο εάν βάσει αυτών θα βρούμε καινοτόμε ε, απαντήσεις για την κλιματική αλλαγή και την ψηφιοποίηση και θα αναλάβουμε τις ευθύνες μας παγκοσμίω. Αυτά είναι τα μεγάλα καθήκοντα που έχουμε. Είμαι όμως αισιόδοξη. Σκεφτείτε πόσες δοκιμασίες και πόσες συγκρούσεις έχει ξεπεράσει η Ευρώπη. Σκεφτείτε πριν από 15 χρόνια την αποτυχία του Ευρωπαϊκού Συντάγματος ή τις οικονομικές και χρηματοπιστωτικές ε, κρίσεις ε, στις οποίες συγκρουστήκαμε ε, σφοδρά ή το μεταναστευτικό πριν από 5 χρόνια. Αυτό δεν ήταν ποτέ εύκολο και πάντα οδήγησε και σε πληγές. Αλλά Ακόμα και πιο πικρές κρίσεις μας βοήθησαν να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες και τη σκέψη των άλλων. Μάθαμε από κοινού. Η Ευρώπη ξεπέρασε όλες αυτές τις κρίσεις γιατί στο τέλος όλοι κατάλαβαν ότι η Ευρώπη ε, έχει κάτι το αδιαπραγμάτευτο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη συνοχή της. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι αναπαλωτρίωτη ε, κοινωνική, πολιτική, οικονομική ανάπτυξη, η προστασία από τις διακρίσεις και ε, ε, τέλος, χωρίς αυτό είναι λιγότερο σημαντικό, η ισότητα, όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη, εκεί είναι τα θεμέλια στα οποία βασίζεται η Ευρώπη και είναι δικαιώματα που ισχύουν για όλους. Δεν ισχύουν περισσότερο για κάποιους και λιγότερο για λίγους. Δεν ισχύουν για κάποιους πάντοτε, για κάποιους άλλους καμιά φορά. Ισχύουν. Αυτό είναι η υπόσχεση της Ευρώπης που θα πρέπει εμείς να εγγυηθούμε. Ότι οι πολίτες, άντρες και γυναίκες θα μπορούν να είναι ελεύθεροι, ε, να ε, ε, ασκούν την, και να βιώνουν την πίστη τους, τις πολιτικές τους πεπιθήσεις και να έχουν την ιδέα για τη ζωή τους και για την ευτυχία τους, εκείνοι που νομίζουν η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία ζει από ε, την ανοιχτή ε, συζήτηση με κριτικό πνεύμα. Μια δημοκρατία που είναι ανεπιθύμητη η αντιπολίτευση, οι αντιπολιτευτικές φωνές ή ε, είναι ανεπιθύμητη η πολυμορφία, η πολιτιστική, η θρησκευτική, η καλλιτεχνική δεν είναι δημοκρατία. Η πανδημία μας έδειξε πόσο πολύτιμα είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα και πόσο ουσιαστικές οι ελευθερίες που εγγυώνται για την προστασία των θεμελιδών δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση επαγρυπνούν ισχυροί θεσμοί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα θεμελιώδη δικαιώματα είναι το πρώτο ε, το οποίο πραγματικά μου είναι προσφυλέ σε αυτή την Προεδρία. Αυτό θα έρθει να υποστηριχθεί και από τη δεύτερη αρχή ε, που συνιστά την Ευρώπη, που είναι η συνοχή μας, διότι για να βγει ενωμένη από την κρίση αυτή η Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε πρόθυμοι, όσες διαφορές και αν έχουμε, να βρούμε κοινέ λύσεις. Αν είμαστε πρόθυμοι να δούμε τον κόσμο και μέσα από τα μάτια του διπλανού για να έχουμε κατανόηση για την προοπτική του άλλου. Η Ευρώπη μετά την κρίση θα είναι πιο ισχυρή από ό,τι πριν εάν ενισχύσουμε αυτή την κοινή αντίληψη που έχουμε. Κανένας δεν πρόκειται μόνος του να βγει από την κρίση αυτή. Είμαστε όλοι ευάλωτοι. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη δεν είναι απλώς ένα δείγμα ανθρωπισμού, μια χειρονομία. Είναι μια ε, βιώσιμη επένδυση. Δεν είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται πολιτικά, αλλά κάτι το οποίο πραγματικά αξίζει και θα πιάσει τόπο. Αυτό είναι και το light motif της Προεδρίας μας. Από κοινού κάνουμε και πάλι την Ευρώπη ισχυρή αυτό ε, είναι κάτι για το οποίο θα αγωνιστώ με όλο μου το πάθος με τη γερμανική κυβέρνηση. Αλλά σας χρειάζομαι και εσά γι' αυτό για να ισχύσουμε αυτή την κοινή αντίληψη στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε το Κοινοβούλιο γιατί εσείς πραγματικά μεταφέρετε την αλληλοκατανόηση που χρειαζόμαστε για να προχωρούμε σε συμβιβασμούς. Εκπροσωπείτε σχεδόν 450 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε 27 κράτη-μέλη. Εσείς μεταφράζετε τις ευρωπαϊκές αρχές. Εσείς εξηγείτε ε, ε, στους πολίτες την Ευρώπη Ευρώπη και έχετε ένα είδος διαμεσολαβητή ανάμεσα στο Στρασβούργο, τις Βρυξέλλε και τι περιφέρειες και τι πατρίδε σας. Δεν επικοινωνείτε απλώς σε 24 γλώσσες, αλλά ζείτε με αυτή την εμπειρία. Ποιο άλλο θα μπορούσε καλύτερα να εξηγήσει την Ευρώπη στα κράτη-μέλη, πιο πολύ από εσά. Γι' αυτό σα παρακαλώ ε, να μεσολαβήσετε ε, για αυτή τη συνοχή και θέλω την υποστήριξή σας σε αυτούς τους δύσκολους ε, καιρούς. Βοηθήστε μας να εμβαθύνουμε την αλληλοκατανόηση και να ενισχύσουμε τη συνοχή στην Ευρώπη. Η ύψιστη προτεραιότητα της Γερμανικής Προεδρίας είναι η Ευρώπη να βγει από την κρίση ισχυρή και ενωμένη. Αλλά δεν θέλουμε απλώ να σταθεροποιήσουμε βραχυπρόθεσμα την Ευρώπη. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ λίγο. Θέλουμε μια Ευρώπη που να δίνει ελπίδα, που να ε, έχει αυτοπεποίθηση και θάρρος απέναντι στις προκλήσεις και τα καθήκοντα. Μια Ευρώπη που να μπορεί να δράσει στο μέλλον με καινοτομία και με βιωσιμότητα, να διεκδικεί και να καταλαμβάνει τη θέση της στον κόσμο. Θέλουμε μια άνοιξη για την Ευρώπη. Ε, εδώ εγγράφεται και η γαλλογερμανική ε, πρωτοβουλία των μέσων Μαΐου. Μαζί με τον Γάλλο πρόεδρο Μανουέλ Μακρόν πρότεινα ένα ταμείο ανάκαμψης 500 δισεκατομμυρίων. Χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλά από τα στοιχεία αυτή τη γαλλογερμανική πρωτοβουλία θα έχει συμπεριλάβει στην πρότασή τη για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο και για το Ταμείο Ανάκαμψη. Αυτό τον καιρό το θέμα αυτό το συζητεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο από την ηγεσία του Σαλ Μισελ. Κοινό μα στόχο είναι να βρεθεί μια συμφωνία ε, ή δυνατόν νωρίτερα. Γιατί ε, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Θα πρέπει να δράσουμε γρήγορα, γιατί εκείνοι που θα υποφέρουν θα είναι οι πιο ασθενείς. Ελπίζω ε, μέσα στο θέρος να επιτύχουμε συμφωνία. Θα χρειαστεί μεγάλη προθυμία για συμβιβασμό από όλες τις πλευρές και από εσάς. Είναι έκτακτη η κατάσταση, μοναδική μάλιστα στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό η Γερμανία και για αυτή την έκτακτη περίσταση ε, προτείνει τα 500 δισεκατομμύρια που είναι επίσης ένα εξαιρετικό έκτακτο ποσό. Τώρα θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Είμαι πεπισμένη ότι η κοινωνική διάσταση είναι εξίσου σημαντική με την οικονομική. Μια Ευρώπη δίκαιη οικονομικά και κοινωνικά είναι αποφασιστική για τη δημοκρατική συνοχή. Είναι η καλύτερη συνταγή απέναντι σε εκείνους που αποδυναμώνουν τις δημοκρατίες μας και θέλουν να αμφισβητήσουν και τα κοινά μας για το λόγο αυτό και για αυτό το λόγο κατά την Προεδρία μας θα αφιερώσουμε ιδιαίτερη προσοχή ε, στα δικαιώματα των νέων και των παιδιών ε, στους νέους και τα παιδιά γενικότερα γιατί είναι το μέλλον της Ευρώπης και θέλουμε ε, να προωθήσουμε την εγγύηση για την νεολαία και την εγγύηση για την είσοδο των νέων στον χώρο εργασίας και δεν θα πρέπει να είμαστε αφελείς. Σε πολλά κράτη-μέλη οι αντίπαλοι της Ευρώπης περιμένουν να καταχραστούν την κρίση ε, με ιδιωτελή κίνητρα. Ε, ε, θα πρέπει να εντείνουμε τη συνεργασία μας και να δείξουμε πού βρίσκεται η προστιθέμενη αξία στην Ευρώπη. Πρέπει να δείξουμε ότι η επιστροφή στον εθνικισμό δεν σημαίνει περισσότερο έλεγχο, αλλά λιγότερο. Μόνο από κοινού μας προστατεύει και μας ενισχύει η Ευρώπη. Γι' αυτό είναι σημαντικό και σωστό οι ε, περιοχές που επλήγησαν ιδιαίτερα από την κρίση να μπορούν να υπολογίζουν στην αλληλεγγύη μας και κυρίως οι κάτοικοι των περιοχών αυτών. Είναι και προς το ίδιο μας το συμφέρον. Ταυτόχρονα όμως στο αποτέλεσμα αυτό σημαίνει πάντα ότι η προσπάθεια που θα πρέπει τώρα να καταβληθεί από όλους δεν θα πρέπει να επιβαρύνει οικονομικά μόνο τα ισχυρά οικονομικά κράτη στην Ευρώπη. Ε, καλούνται όλοι να ε, βγουν στη θέση του άλλου. Ας σκεφτούμε λοιπόν τι μπορούν να δώσουν τα κράτη-μέλη και τι δεν μπορούν να δώσουν οικονομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Και σας παρακαλώ σε όλα αυτά ε, να με υποστηρίξετε ως Ευρωβουλευτές. Είμαι πεπισμένη ότι ο καθένας ε, στην κρίση αυτή είναι πρόθυμος να δείξει εξαιρετική ελεγγύη. Η Γερμανία είναι πρόθυμη. Η καταπολέμηση ε, της ε, πανδημίας και των επιπτώσεών της φραγίζει την Προεδρία μας. Ταυτόχρονα όμως θα πρέπει να ασχοληθούμε και με τις άλλες μεγάλες προκλήσεις που έχουμε είναι τα θέματα 3, 4 και 5 ε, για την Ευρώπη, όπου σας ανέφερα προηγουμένω. Το πρώτο είναι η κλιματική αλλαγή. Πριν από ένα εξάμεινο περίπου, η πρόεδρος τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, παρουσίασε το πρόγραμμά της για την προστασία του κλίματος. Ήταν τα λόγια της πραγματικά σήμαντα και σας είπε ότι τώρα θα πρέπει να δράσουμε η Ευρώπη αν θέλουμε ο πλανήτης να παραμείνει βιώσιμος. Είμαι πεπισμένη ότι μια παγκόσμια λύση τη κλιματική αλλαγή είναι δυνατή μόνο εφόσον η Ευρώπη είναι πρωτοπόρος στο ρόλο της. Η στρατηγική για την Πράσινη Συμφωνία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι γι' αυτό για μας ε, σημαντική πηξίδα. Θέλουμε ε, να προχωρήσουμε προς μια κοινωνία και οικονομία ουδέτερη ως προς το διοξίδιο του άνθρακα με ισχυρές επιχειρήσεις και νοτόμες. Ε, μια οικονομία που να σέβεται το περιβάλλον, τη φύση ε, και να προστατεύει ε, και την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και να την ενισχύει. Γι' αυτό είναι σημαντικό η ιδιαιτερότητα της Ευρώπης προς το κλίμα μέχρι το 2050 να κατοχυρωθεί νομοθετικά. Γι' αυτό καλωσορίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, μέχρι το 2030 να μειωθεί το διοξείδιο του άνθρακα κατά 50 με 55% σε σχέση με το έτος αναφοράς 1990. Και θα τα δούμε αυτά και νομοθετικά. Άλλη μεγάλη πρόκληση, τέταρτο σημείο, το οποίο θα μας απασχολήσει ιδιαίτερα στην Προεδρία μας, είναι η ψηφιοποίηση. Η ψηφιακή αλλαγή και αυτή όπως και η κλιματική αλλαγή και η προστασία του κλίματος απαιτεί να αλλάξει βιώσιμα ο τρόπος με τον οποίο ε, ζούμε και παράγουμε. Αυτό δημιουργεί άγχος σε πολύ κόσμο γιατί ε, φοβάται μήπως χάσει το γνώριμο περιβάλλον, φοβάται τις ταχύτητες ε, με τις οποίες επέρχεται η αλλαγή. Είναι κατανοητό αυτό. Αλλά η δέσμευση για την ψηφιοποίηση όπως και για την προστασία του κλίματος δεν σημαίνει ότι θα απεμπολίσουμε ό,τι γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και ό,τι έχει κατοχυρωθεί και θα ρηψοκινδυνεύσουμε ε, τις θέσεις εργασίας εκατομμύριων ε, Ευρωπαίων. Το αντίθετο, είναι απαραίτητη αυτή η αλλαγή και ε, στο Δινεκές θα παρέχει μεγαλύτερη προστασία και μεγαλύτερες εγγύησεις γιατί είδαμε ακριβώς τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες πόσο εξαρτάται ψηφιακά η Ευρώπη από τρίτες χώρες. Αυτό το είδαμε πολλοί από εμά, ε, χωρίς καμία αμφιβολία, καθημερινά στις επικοινωνίες μας, στην τεχνολογία ή στην παροχή υπηρεσιών. Είναι σημαντικό η Ευρώπη ψηφιακά να γίνει κυρίαρχη. Ιδιαίτερα σε τομείς κλειδιά όπως είναι η κβαντική υπολογιστική και η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και μια ασφαλής ψηφιακή υποδομή. Αυτά είναι θέματα που θέλουμε να προχωρήσουμε. Αποφασιστική επίσης είναι η αποτελεσματική προστασία των δημοκρατιών μας από εκστρατείες παραπληροφόρησης και επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Γιατί η δημοκρατία χρειάζεται μια κοινή όπου να μπορεί ε, κανείς να ενημερώνεται ε, και η γνώση και η άποψη να κυκλοφορεί και οι πολίτες να συνεννοούνται και να ε, ενημερώνονται για το πώς θέλουν να ζήσουν. Σήμερα βλέπουμε ψεύδι και παραπληροφόρηση, τα οποία όμως δεν μπορούν να καταπολεμήσουν την πανδημία και εξίσου λίγο βοηθούν το μίσος και η υποδάβλησή του. Σε μια δημοκρατία λοιπόν χρειάζεται αλήθεια, χρειάζεται διαφάνεια. Και αυτό διακρίνει την Ευρώπη και γι' αυτό θα αγωνιστεί η Γερμανία με την Προεδρία. Και κατά πέμπτον, για την ευθύνη της Ευρώπης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Αν δούμε τι γίνεται στο χάρτη, θα δούμε ότι πέρα από την Μεγάλη Βρετανία και τα Δυτικά Βαλκάνια, η Ευρώπη και τα εξωτερικά της σύνορας έχουν να κάνουν με την Τουρκία, την Συρία, την Ρωσία, την Λευκορωσία, την Λίβανο, την, ε, την Αίγυπτο, την Τινησία, την Αλγερία, το Μαρόκο. Περιτριγυρίζεται λοιπόν από όλε αυτέ τι χώρε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, ζούμε και σε μια εποχή παγκόσμιων αλλαγών. Υπάρχουν μετατοπίσει εξουσία και η Ευρώπη με όλα τα, κρατικά, τα κράτη-μέλη και τι διατλαντικέ σχέσει, πρέπει να επιδροθεί στον εαυτό τη. Εμείς μπορούμε και πρέπει να αποφασίσουμε μαζί πώς ε, θα διαμορφωθεί η Ευρώπη και ποια θέλει να είναι η Ευρώπη σε αυτή την ε, ταχαίως μεταβαλλόμενη κατάσταση. Είμαστε σοβαροί για την Ευρώπη. Θέλουμε μια Ευρώπη για την ελευθερία και για την ταυτότητά της, η οποία θα αγωνιστεί για τις αξίες αυτές. Υπάρχει η ανάγκη λοιπόν να ανισχύουν όλα αυτά, να υπάρξει μια ισχυρή πολιτική εξωτερική και πολιτική άμυνας σε ό,τι αφορά τι μελλοντικέ μα σχέσει με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα μα απασχολήσει πολύ το επόμενο εξάμεινο και η πρόοδο των διαπραγματεύσεων ω τώρα είναι ακόμα σε δύσκολο επίπεδο. Θέλουμε να επιταχύνουμε λοιπόν τι διαπραγματεύσει αυτέ προκειμένου να συνάψουμε μια συμφωνία το φθινόπωρο η οποία θα επικυρωθεί στα τέλη του χρόνου. Θα ταχθώ υπέρ μια καλή λύση, ε, αλλά θα πρέπει κυρίως να φροντίσουμε να προβλέψουμε για την περίπτωση που δεν θα υπάρξει συμφωνία. Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας μας λοιπόν θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και θα επικεντρωθούμε σε τρει ε, άλλου ε, τομεί εξωτερική πολιτική. Καταρχά, σε ό,τι αφορά την διάσκεψη προσχώρησης τη Μακεδονία, τη Βορείας Μακεδονίας, της Αλβανίας επίσης και και στην παροχή μια διάσταση προσχώρηση στι υπόλοιπε χώρε της Δυτικών Βαλκανίων και κατά δεύτερον σε ό,τι αφορά την Αφρική και την Αφρικανική Ένωση έχουμε τη διάσκεψη η οποία επέκειται. Και εδώ πέρα θα πρέπει να κοιτάξουμε και θέματα συνεργασίας για τη μετανάστευση. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο, πιο πολύ κόσμο από ποτέ που βρίσκεται σε καθεστώς δίωξης. Και θα πρέπει να επικεντρωθούμε και να κάνουμε προσπάθειες περαιτέρω σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου και πολιτική μετανάστευση στην Ευρώπη. Αυτό απαιτεί ω ερώτημα και ω θέμα μεγάλη πολιτική ευαισθησία. Δεν μπορούμε να το αμελήσουμε. Θα πρέπει να αναλάβουμε την πολιτική αυτή ευθύνη, την ανθρωπιστική αυτή ευθύνη. Και τέλος. Οι στρατηγικέ μας ε, σχέσεις με την Κίνα θα μας απασχολήσουν επίσης. Έχουμε στενέ ε, εμπορικές ε, σχέσεις, αλλά από την άλλη έχουμε και διαφορετικές κοινωνικές και οικονομικές οράματα. Και παρά το γεγονός ότι δεν θα γίνει διάσκεψη με την Κίνα, θέλουμε να συνεχίσουμε τον ανοιχτό διάλογο με την Κίνα κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Προεδρίας. Θα θέλουμε επίσης να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε κατά πόσο σε θέματα πολιτικής άμυνας και πολιτικής ασφάλειας θέλουμε να διατηρήσουμε το κοινό μας όραμα και το ποια θα είναι τα διδάγματα τα οποία θα έχει η Ευρώπη από την κρίση του κορονοϊού και πώς μπορούμε έτσι να ενισχύσουμε τον οικονομικό κλάδο αυτή η συζήτηση θα πρέπει να γίνει και στο πλαίσιο μια διάσκεψης για το μέλλον τη Ευρώπη, Το είναι την προηγούμενη χρονιά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το αναπτύξετε κι εσεί με τα πολλαπλά ψηφίσματά σα. Θέλω μια διάσκεψη η οποία θα επικεντρωθεί σε λίγα θέματα για να έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα προκειμένου να προσφέρει στους πολίτε από τα διάφορα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να συζητήσουν. Και σήμερα συζήτησε το θέμα αυτό με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον κύριο Ντάβιτ Σασόλη. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, κυρίε και κύριοι, θέλουμε την Ευρώπη. Αν την θέλουμε, χρειαζόμαστε αυτά που σα ανέφερα. Θεμελιωδή δικαιώματα, συνοχή, απαντήσει για την αλλαγή του κλίματο και την ψηφιοποίηση και μια ευρωπαϊκή ευθύνη σε όλη την φίλιο. Θα πρέπει να διαμορφώσουμε την Ευρώπη με πράσινο τρόπο με πιο ψηφιακό τρόπο για να είναι πιο ανταγωνιστική και πιο κοινοτόμα. Γιατί η Ευρώπη σε διεθνές επίπεδο θα πρέπει να εκπροσωπεί την κοινοτομία και την βιωσιμότητα. Αυτό είναι το όραμα για την Ευρώπη. Θα ήθελα να κλείσουμε μια προσωπική σκέψη. Αγαπώ τη μουσική. Και είναι μεγάλη μου χαρά που στην Προεδρία μας έχουμε μια ιδιαίτερη ημερομηνία τον ε, Δεκέμβριο του 2020 ο συνθέτης ε, Μπετόβεν θα έχει κλείσει τα 250 χρόνια του. Αυτή είναι ενάτη συμφωνία. Πάντα ε, με γεμίζει χαρά. Κάθε φορά που την ακούω ανακαλύπτω κάτι καινούριο στην μουσική και αυτό πραγματικά με συγκινεί. Όπως και με την Ευρώπη. Πάντα έχει κάτι καινούριο να ανακαλύψει κανείς. Και αυτό πάντα με εντυπωσιάζει. Θα ήθελα λοιπόν να κλείσω με την επιθυμία το μήνυμα της μουσικής αυτής να είναι η ιδέα της αλληλεγγύης και της ομόνοιας. Αυτό να αποτελέσει το κοινό μας όραμα στην Ευρώπη. Ποιο μήνυμα θα ήταν άλλωστε πιο κατάλληλο ότι η Ευρώπη είναι ικανή να κάνει τα πάντα αν ε, έχουμε αλληλεγγύη και βοηθάμε ένα τον άλλον. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε κυρία Μέρκελ. Και τώρα το λόγο έχει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Καγκελάριε. Χαιρόμαστε που έχει έρθει η Γερμανική Προεδρία οι προεδρίες δεν είναι κάτι που επιλέγει κανείς ε, και σίγουρα ε, ακολουθούν ένα προδιαγραμμένο πρόγραμμα και η Γερμανία έπεσε σε μια φάση η οποία θα μπορούσε να είναι πιο γεμάτη με προκλήσεις. Οι προσδοκίες από τη Γερμανική Προεδρία είναι υψηλέ και ξέρω ότι αυτό αποτελεί παράγοντα πίεση, αλλά είναι και κάτι όμορφο γιατί δείχνει ε, ότι σας εμπιστευόμαστε με αυτό το μεγάλο έργο. Κυρίες και κύριοι, η κρίση του κρονοϊού θέτει πολλά υπό αμφισβήτηση σε κοινωνικό επίπεδο, σε οικονομικό επίπεδο. Ακόμα και τα αυτονόητα. Ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίζουμε οι τους δε που βλέπουμε τον εαυτό μας και οι σχέσεις που έχουμε μεταξύ μας. Όλα αυτά λοιπόν σε ένα παγκόσμιο σκηνικό όπου οι τρέχουσες δομές διαλύονται και υποχωρούν. Μέσω της ε, κρίσης του κορονοϊού έχουμε κάτι και έχουμε σκεφτεί την αξία της αλληλεγγύης, της κοινότητας και όλα αυτά έχουν αποκτήσει μια νέα διάσταση. Σκεφτόμαστε με διαφορετικό τρόπο πλέον λοιπόν την κοινή αξία της Ευρώπης η οποία διαμορφώνεται με νέο τρόπο κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα. Και ναι, όντως στην αρχή πολύ κοιτάξαμε στο τοπικό επίπεδο, στο μικρό επίπεδο αν θέλετε, ένδοθεν αλλά σταδιακά γυρίσαμε το βλέμμα μας στα ευρωπαϊκά και τα βλέπουμε όλα αυτά πλέον με μάτια ευρωπαϊκά, με μια καρδιά ευρωπαϊκή. Κυρία Καγκελάρη. Τις τελευταίες εβδομάδες η Γερμανική Προεδρία διακατέχεται από αυτό το πνεύμα της ευθύνης για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ακούμε από όλες τις πλευρές της Υπήρου ε, εν το μέσο της κρίσης ε, διάφορες φωνές οι οποίες μας κάνουν να απελπιζόμαστε και να μην πιστεύουμε ότι θα υπάρξει κοινή λύση. Αυτό που είναι καλό για την Ευρώπη είναι καλό και για μας. Όταν τα ακούω όμως αυτά, ξέρω ότι αυτός είναι ο ήχος της Ευρώπης τον οποίο θέλω να ακούω. Και αυτό λοιπόν το πνεύμα δεν είναι κακός ε, σύμβουλος για μια τέτοια προεδρία η οποία θα είναι καθοριστική για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Γερμανική Προεδρία και όλοι μας το επόμενο εξάμεινο. Αυτές οι προκλήσεις πραγματικά είναι άνευ προηγουμένου, πρωτοφανείς. Και το τελευταίο εξάμεινο πάνω από 100.000 ε, ζωές χάθηκαν στην Ευρώπη λόγω της πανδημίας COVID-19 και εισήλθαμε στη χειρότερη ύφεση τα τελευταία περίπου 100 χρόνια, τον τελευταίο αιώνα. Και μάλιστα οι χθεσινέ προβλέψει για το καλοκαίρι δείχνουν μια συρρήκνωση πάνω από 8% φέτος με μερική μόνο ανάκαμψη του χρόνου. Η τρέχουσα κρίση είναι βαθύτερη και πολύ ευρύτερη από αυτή που βιώσαμε πριν από μια δεκαετία. Η προηγούμενη όμως κρίση της προηγούμενης δεκαετίας είναι ακόμη παρούσα, πολύ ζωντανά στη μνήμη μας. Και μερικά κράτη-μέλη στη διάρκεια της κρίσης ε, της οικονομικής ε, είδαν την ε, ανεργία να εκτινάσεται στα ύψη. Είδαν ε, τους νέους τους να αποδημούν, αναζητώντας ε, ευκαιρίες απασχόλησης στην Αλαδαπή. Είδαν πρωτοφανή μείωση των ε, κρατικών επενδύσεων που έφτασαν σε ιστορικού επίπεδο χαμηλά επίπεδα. Κάτι που κατέστρεψε τα δημόσια προγράμματα και ε, έπληξε τις ε, κρατικές υποδομές. Για, πολλούς, για πολλά κρατημέλη η οικονομική κρίση ήταν μια τραυματική εμπειρία. Δεν θα πρέπει όμως να βιώσουμε και δεν θα βιώσουμε κατά ανάγκη το ίδιο και σε αυτή την οικονομία. Σε πολλά μέρη της Ένωσης ε, στηρίχθηκε η οικονομία από ισχυρές οικονομικές κρατικές επενδύσεις από την αρχή της κρίσης. Πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να παραμείνουν στις θέσεις απασχόλησης. Και μάλιστα τότε ε, υιοθετήσαμε τη μερική απασχόληση σε ευρύτερο επίπεδο με περιορισμένο ε, ωράριο. Και μάλιστα έτσι μερικοί θα ε, βγούμε δυνατότεροι από την κρίση και θα πρέπει να αντλήσουμε κάποια διδάγματα από την τρέχουσα κρίση και αυτή τη, στιγμή, αυτή τη φορά να συνεργαστούμε, να εξέλθουμε από κοινού από την κρίση. Αν το επιχειρήσουμε, ίσως βγούμε ισχυρότερη από την κρίση αυτή χάρη στον κοινό ευρωπαϊκό στόχο και χάρη στο, στην Ευρώπη της επόμενης γενιάς, στο πρόγραμμα Next Generation EU. Και μάλιστα η Προεδρία αυτή διάλεξε μία λέξη και την έφερε στο επίκεντρο του προγράμματος. Το μαζί, το gemeinsam. Όλοι μαζί. Και αυτή είναι η κινητήριος δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σταθώ σε δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αλληλεγγύη σημαίνει ότι αυτοί που το χρειάζονται θα λάβουν περισσότερη ενίσχυση. Αυτό όμως ε, που δεν ε, σημαίνει είναι αδράνεια, έλλειψη δράσης. Γι' αυτό και το πρόγραμμα Next Generation EU συνδέει τις επενδύσεις με τις ε, μεταρρυθμίσεις με βάση τις ειδικές ένα χώρα και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Κάθε κράτος μέλος πρέπει να κάνει το καθήκον του. Για όλα τα κρατη υπάρχουν ειδικέ συστάσεις αναχώρας που θα πρέπει να συνδέονται με τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις. Και αν πραγματικά εξέλθουμε ισχυρότεροι από την κρίση αυτή, θα πρέπει όλοι να αλλάξουμε προς το καλύτερο. Και καμία χώρα μέλο δεν εξαιρείται από αυτό. Όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε προ το καλύτερο. Όλοι έχουμε δρόμο μπροστά μα να κάνουμε. Και αυτό περιμένει από εμά και ο ευρωπαϊκό λαό, η Ευρωπαϊκή λαοί. Και Σίγουρα κάθε λαός είναι διαφορετικός ε, ως προς τις προσδοκίες του, αλλά όλοι οι λαοί είναι απόλυτα ενωμένοι γιατί όλοι θέλουν να πίνουν καθαρό πόσιμο είδωρ, να αναπνέουν καθαρό αέρα, να βλέπουν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν στη φύση και σίγουρα αυτό που δεν θέλουν οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι να συμβάλλει η πολιτική στις αυξανόμενες ε, πλημμύρες, στις ανοβρίες, στους καύσονες και αυτό είναι ένα πραγματικά ε, πιθανό σενάριο αν δρανήσουμε, αν δεν λάβουμε δράση. Οπότε η οικονομική ανάκαμψη είναι αναπόσπαστα δεμένη με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη ε, και με την ψηφιοποίηση και αδιαχώριστη και από την ανθεκτικότητά μας. Και το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι δεν θα πρέπει να αμελήσουμε ε, για το πολιτέ δημοσιονομικό μα πλαίσιο, τον, επόμενό μας, τον επόμενό μας επταετή προπολογισμό. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Το Next Generation EU θα αντιμετωπίσει την οξία κρίση. Το πολιτέ όμω δημοσιονομικό πλαίσιο είναι εκεί και θα παραμείνει. Είναι το σημαντικότερο εργαλείο που έχουμε για να υλοποιήσουμε τους μακροπρόθεσμους στόχους μας. Την ε, καινοτομία, την έρευνα, την μετανάστευση, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια. Ενδεικτικά αναφέρω μερικούς στόχους. Και όλες οι πολιτικές αυτές χρειάζονται την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και χρειάζονται έναν ισχυρό επταετή προπολογισμό για να μπορέσουν να υλοποιηθούν. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, όλα αυτά θα πρέπει να τα συμφωνήσουμε τώρα στο εγγύς μέλλον, τις επόμενες εβδομάδες, για να χαράξουμε το δρόμο και για τα υπόλοιπα θέματα που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε. Μέχρι τα τέλη του έτους θα πρέπει να ανοίξουμε το δρόμο ε, προς το στόχο της κλιματικά ουδέτερης Ευρώπης. Το Σεπτέμβριο θα προτείνουμε τους νέους κλιματικούς στόχους μας για το 2030 φυσικά με μια εύρωστη μελέτη επιπτώσεων και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά. Η συνεργασία μας είναι ζωτική σημασία στα θέματα αυτά. Επίσης, θέλουμε να περάσουμε σε μεγαλύτερη ταχύτητα σε ό,τι αφορά την ψηφιακή μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, στα γαλλικά, η κυρία Φοντερ Λάιεν, στη διάρκεια της Προεδρίας θα κάνουμε το παν δυνατό για να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις νέες μας σχέσεις με σεβασμό φυσικά των αρχών μας και με διαφύλαξη της ευρωπαϊκής μας ενότητας. Το ίδιο ισχύει και είναι σημαντικό να κρατήσουμε μια ισχυρή διατλαντική σχέση παρά τα προβλήματα, τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Εταιρική σχέση με την Αφρική επίσης βρίσκεται στην καρδιά του προγράμματος της Γερμανικής Προεδρίας αλλά βρίσκεται στο επίκεντρο και του προγράμματος Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αντιμετωπίζοντας την πανδημία και τον ιό COVID, θα πρέπει να δείξουμε ότι η εταιρική σχέση με την Αφρική δεν υπάρχει μόνο για τις εύκολες για την εύκολη περίοδο, για τον ε, καλό καιρό, αλλά ότι είμαστε αλληλέγγυοι και όταν αρχίζουν και διαφαίνονται κάποια σύννεφα. Επίσης θέλουμε μια πιο ισορροπημένη εταιρική σχέση και με την Κίνα. Και τέλος και κυρίως ήγηκε η ώρα για να κηρύξουμε την έναρξη της ε, διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Όλοι θέλουμε να δώσουμε το εναρκτήριο λάκτισμα από τη στιγμή που θα μας το επιτρέψει φυσικά η υγειονομική κατάσταση. Για όλα αυτά τα θέματα είμαι ευτυχής που μπορούμε να υπολογίζουμε στην γερμανική εμπειρία ξεκινώντας με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας. Γιατί τώρα είναι η στιγμή να δράσουμε από κοινού και να υιοθετήσουμε το σύνθημά σας. Μαζί για την ανάκαμψη της Ευρώπης. Όλοι μαζί για να οδηγηθούμε στην ανάκαμψη της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την πρόεδρο Φόντερ Λάιεν και τώρα ακούμε τους ε, αρχηγούς των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Μάνφρετ Βέμπερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Παρακαλώ. Καγκελάρια Μέρκελ, πρόεδρε Φόντερ Λάιεν, πρόεδρε σα όλοι αγαπητοί συνάδελφοι. Φραντσέσκο ονομάζεται. Και είναι γιατρό των Περγαμών και έρχεται αντιμέτωπο με μια κατάσταση την οποία κανένα γιατρό δεν ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπο. Ήθελε να σώσει ζωέ, αλλά δεν είχε πλέον κλίνε στο νοσοκομείο του και ε, αναγκάστηκε να πάρει αποφάσει ζωή και θανάτου. Και εκ παραλίλου, σε γειτονικέ χώρε στην Ευρώπη υπήρχε μπλοκάρισμα τη εξαγωγή ε, για τι μάσκε. και τελικά ε, επεκράτησαν οι εθνικισμοί και τελικά ο Φραντσέσκο απελπίστηκε και δεν είναι μόνος του ο Φραντσέσκο πολλοί είναι οι άνθρωποι εκείνοι ε, που αναρωτιούνται τι έγινε με την αλληλεγγύη πού είναι η Ευρώπη όταν τη χρειαζόμαστε πιο πολύ παραποτέ και έτσι λοιπόν υψηλέ είναι οι προσδοκίες τι οποίε έχει όλος ο κόσμος από τη Γερμανική Προεδρία, αγαπητή Άγγελα Μέρκελ. Η Ευρώπη σα εμπιστεύεται όπου επικρατούν δυνάμεις απόσχησης, ε, εσείς θεωρείστε δύναμη ενωτική και αυτό θα είναι σημαντικό για την ανάκαμψη της Ευρώπης μετά την κρίση του COVID-19. Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει, να είναι αυτή η Προεδρία μια υποσημείωση και μόνο στην ιστορία. Χρειαζόμαστε λοιπόν συνοχή στην Ευρώπη και το κατά πόσο θα καθορίσει κατά πόσον το 2020 και μετά η δεκαετία αυτή θα είναι καλή ή όχι. Και κοιτάμε προ τα πίσω. Διαπιστώνουμε ότι υπήρξε η κρίση του ευρώ, είχαμε την κρίση τη μεταναστευτική και τώρα έχουμε την κρίση του COVID-19. Περνάμε λοιπόν από κρίση σε κρίση. Και γιατί, γιατί συχνά φοβόμαστε, φοβόμαστε την αλληλεγγύη. Ο φόβο είναι ο εχθρό τη ελευθερία μα. Α ξαναδούμε τον Φραντσέσκο. Ο φόβο δεν ήταν αυτό που τον ε, καθοδήγησε, το κουράγιο, η τόλμη. Τόλμη χρειαζόμαστε για να δείξουμε λοιπόν αλληλεγγύη και χρειαζόμαστε καταρχά το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρώτο βήμα είναι αυτό. Θα πρέπει να λεφτούν αποφάσει αυτό το μήνα. Τόλμη και στο μέλλον χρειάζεται. Δεν μπορούμε να δαπανίσουμε του πόρου αυτού, τα οποία τα έχουμε δανειστεί από τα παιδιά μα για το παρελθόν. Πρέπει να χτίσουμε το μέλλον, το κλίμα, την ψηφιοποίηση, τη βιομηχανία. Μια υπερσύγχρονη ήπειρο. Τον τόλμη να είμαστε δίκαιοι. Όποιο δανείζεται χρήματα θα πρέπει να μα πει αυτό που δανείζεται τα χρήματα πώ θα τα επιστρέψει. Πιστεύει κανεί εδώ σε αυτή την αίθουσα ότι μπορεί να ξεπληρώσει τα χρέη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ε, να βάλει το χέρι στη τσέπη στους ιδίους πόρους. Δεν νομίζω. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει το 2020. Και τόλμη για να είμαστε ελεύθεροι επίσης. Γιατί η Ευρώπη δεν είναι ταμείο. Είναι μια ένωση κοινών αξιών. Θα πρέπει να γίνεται σεβαστό στο κράτο δικαίου και αναφερθήκατε και σε άλλα θέματα στην ε, παρέμβασή σα σε ό,τι αφορά την παρουσίαση τη γερμανική Προεδρία. Θα πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένε λύσει και απαντήσει για την μετανάστευση, το Brexit, το εμπόριο και σε πολλού άλλου τομεί. Συνάδελφοι, όμω αυτό που φοβάμαι είναι το εξή ότι όλα αυτά πολύ απλά δεν θα αρκέσουν. Δεν φτάνουν. 70 χρόνια μετά το Σούμαν είμαστε αντιμέτωποι με ακόμα πιο μεγάλες προκλήσεις. Τότε η Ευρώπη ήταν ε, σε ρήπια, ο κόσμος ε, πεινούσε, ήταν ε, χωρίς σπίτι. Ο Σούμαν όμως είχε την τόλμη το κουράγιο να κοιτάξει πέρα από τα καθημερινά. Είχε πίστη, στην Ευρώπη. Και σήμερα έχουμε ένα τεράστιο καθήκον. Έχουμε την ψηφιακή επανάσταση, μια εχθρική Ρωσία, την ε, Αμερική που υποχωρεί, την Κίνα η οποία ε, επιμένει, η Αυστραλία καίγεται. Μια φιλεύθερη δημοκρατία στην οποία όλοι πιστεύουμε δέχεται καθημερινές επιθέσεις. Ναι, και σήμερα λοιπόν έχουμε καθημερινές επιθέσεις. Το θέμα λοιπόν είναι θα έχουμε την τόλμη να κοιτάξουμε πέρα από τα καθημερινά. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο θέτω. Αν θέλουμε λοιπόν να τοποθετηθούμε πάνω από τα καθημερινά, θα πρέπει να κοιτάξουμε την ταυτότητά μα. Σήμερα δικαιολογούμε την Ευρώπη με τι μικρέ καθημερινέ επιτυχίε. Τα τέλη το ότι δεν έχουμε ελέγχου στα σύνορα. Και άλλα τέτοια καθημερινά. Αγαπητοί συνάδελφοι, όμω αυτή η προπτική είναι μάλλον εγωιστική. Αυτό τι σημαίνει ότι αν με βολεύει η Ευρώπη, καλή είναι η Ευρώπη. Αν δεν με βολεύει, δεν είναι καλή αυτό δεν αρκεί πλέον. Αυτή η θεώρηση της Ευρώπης και πάλι αφήνει τον Φραντσέσκο μόνο του στη μονάδα αν έκανα και ανήμπορο. Δεν υπάρχει δηλαδή κλίμα ε, και ατμόσφαιρα ταυτότητας κοινωτικής. Για να το πω με όρους ΕΛΚ, είναι ο ευρωπαϊκός τρόπος ζωής. Ε, όπως τον περιγράψατε εσείς κυρία Καγκελαρία, είναι η ε, κοινωνική, κοινωνία, κοινωνική α, οικονομία, η κατάργηση της αντικής ποινής. Στη ΣΥΠΑ έχουν ακόμα τα αντική ποινή, δεν έχουν σύστημα υγειονομική περιθάλψη στην Κίνα, δεν έχουν καθόλου ελευθερίε και α, τέτοια θεμελιώδη δικαιώματα. Ο, ο τρόπο αυτό, ο ευρωπαϊκό τη ζωή, είναι μοναδικό και είμαι περήφανο που μπορώ να πω ότι είμαι Ευρωπαίο. Θα πρέπει να ανακαλύψουμε εκ νέου λοιπόν το το θάρρο, την τόλμη για το μέλλον, να κάνουμε το επόμενο βήμα. Η αλληλεγγύη θα διαρκέσει μόνο και οι αξίε μα θα επικρατήσουν σε παγκόσμιο επίπεδο μόνο αν υπάρχει ένα κοινό πνεύμα κοινότητα αλληλεγγύη. Και χρειάζεται λοιπόν μια ευρωπαϊκή δημοκρατία με την οποία θα συνδεθεί ο κόσμο. Εκεί θα πρέπει να σκεφτούμε σε μεγάλο ε, επίπεδο, όπω έκανε ο Χέλμουντ Κόλ, ο Λαχιβαλέσα και πολλοί άλλοι. Αγαπητή κυρία Καγκελάρια, υπολογίζω και σε εσά και στην Γερμανική Προεδρία ότι θα καταφέρετε να πετύχετε όλα αυτά. Όχι μόνο δηλαδή να τα απεξέλθετε στα καθημερινά, αλλά να κάνετε και το επόμενο βήμα στην Ευρωπαϊκή Ενωποίηση, να, χρησιμοποιη... να ιδρυθεί μια ζωντανή Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Ναι, λοιπόν, στην Ευρωπαϊκή Ταυτότητα, ναι, στον Ευρωπαϊκό Τρόπο Ζωή. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο έχει τώρα η Πρόεδρο Γκαρσία Πέρες η πρόεδρος τη της ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Σας ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αξιότιμοι καγκελάρια. Καλώ ήρθατε στον οίκο αυτό που είναι ο οίκο τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Υπάρχουν κάποιε στιγμέ στην ιστορία που απαιτούν όραμα και θάρρο. Και αυτή είναι μία από τι στιγμέ αυτέ. Και γι' αυτό μπορούμε να βασιστούμε, πιστεύω, στην εμπειρία σας και στην γερμανική σας ιδιότητα και ποιότητα για να αναζητήσετε συνενέσεις πέραν των ιδιαίτερων και ατομικών συμφερόντων ή εθνικών συμφερόντων. Ε, έχουμε μπροστά μα ένα εξάμεινο που θα χαράξουν την πορεία τη Ευρώπη και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτό το εξάμεινο για να αντιμετωπίσουμε ε, εμφανεί αδυναμίε. Θα πρέπει να αντιδράσουμε πιο άμεσα, ταχύτερα και πιο ενωμένα απέναντι στι κρίσει και θα πρέπει να ενισχύσουμε του στρατηγικού μα κλάδου και την ανθεκτικότητά μα ω κοινωνία. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για να συμφωνήσει για το Ταμείο Ανάκαμψης και τον επόμενο προλογισμό θα έχει ε, μεγάλη σημασία. Και σίγουρα αυτές τις μέρες μιλάμε πολύ για χρήματα, αλλά η συζήτηση αυτή δεν περιορίζεται μόνο στα ποσά και στους αριθμούς. Είναι μια συζήτηση για το πολιτικό σχέδιο. Όταν ο Ρόμπερτ Σούμαρ πρότεινε στον Κόνερα Τεντενάουερ την κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, Εκείνος αντιλήφθηκε αμέσω την ιστορική του διάσταση. Δεν επρόκειτο για ένα τεχνικό υλικό σχέδιο. Πρόκειται για μια ηθική ευθύνη απέναντι στους λαούς της Ευρώπης. Το μέλλον της ε, Γερμανίας σήμερα συνεχίζει να εξαρτάται από το μέλλον της Ευρώπης και τον άπαλιν. Θα ήθελα το επόμενο εξάμεινο λοιπόν να συνεργαστούμε στενά για να ξεπεράσουμε τις διαφορές και τις διαστάσεις μεταξύ Βορράς και Νότου, Ανατολής και Δύσης και να ενισχύσουμε την ένωσή μας προς το συμφέρον και το καλό των Ευρωπαίων πολιτών. Ας δείξουμε στον κόσμο ότι είναι δυνατό να δημιουργήσουμε μια πιο δίκαιη, πιο αηφόρο κοινωνία που θα σκέφτεται και το περιβάλλον και τις επερχόμενες γενιές. Μια κοινωνία ισότιμη, με γυναίκες σε υψηλόβαθμες θέσεις, ε, σε, όλες, ε, σε όλα τα θεσμικά όργανα, που θα αξιοποιεί τις δημόσιες πολιτικές, της υγείας, της παιδείας, που θα προστατεύει τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες, που θα απαιτεί δίκαιους μισθούς, που θα αξιοποιεί τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία και θα διαχειρίζεται τις μεταναστευτικές με αλληλεγγύη. Όλα αυτά θα είναι στο πρόγραμμά σα και μπορείτε να στηριχτείτε και στη δική μα συνεργασία. Είδαμε ότι τα μοτίβα του παρελθόντων και οι μέθοδοι του παρελθόντος δεν λειτουργήσαν. Και μαζί με τους ε, συναδέλφους του S5 ε, χαράξαμε έναν οδικό χάρτη για μια Ευρώπη που θα είναι πιο κοντά στους πολίτες και πιο δίκαιη. Και γι' αυτό δύο είναι τα ζητούμενα. Ήδη οι πόροι πρώτα απ' όλα για να, για να λύσουμε διασυνοριακά προβλήματα και επίσης με τη διάσκεψη της Ευρώπης να ξαναδημιουργήσουμε δεσμούς με τους Ευρωπαίους πολίτες. Κυρία Καγκελάρια, έχουμε κοινέ ευρωπαϊκές αξίες. Ας έχουμε λοιπόν και κοινή δέσμευση να τις προστατεύσουμε και να συνεργαστούμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος Τσόλος ε, της ομάδας Renew Europe. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κυρία Κακελάρη, ακούγοντας την παρέμβασή σας συγκινήθηκα πολύ έντονα και οι δυο μας ε, καταγόμαστε από την ίδια γωνιά της Ευρώπης ε, που συχνά ορισμένοι ονομάζουν Ανατολική Ευρώπη όπου επί δεκαετίες ε, είχε συνθλιβεί από αυταρχικά καθεστώτα και δικτατορίες και είναι πολλοί οι συνάδελφοι που είναι από αυτή την περιφέρεια της Ευρώπης. Σήμερα όμως θέλουμε όλοι το ίδιο, μια ισχυρή Ευρώπη, ελεύθερη και ευημερούσα. Θα πρέπει όμως γι' αυτό να αγωνιστούμε απέναντι στην αποθάρρυνση και ε, την ε, ε, μείωση της ε, ευρωπαϊκής ιδέας που φθήνει. Θα πρέπει να δώσουμε νέα πνοή ε, στα ευρωπαϊκά εγχειρήματα, γιατί μόνο η ελπίδα, όπως είπατε, θα θριαβεύσει απέναντι στην απογοήτευση. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι κάτι στο οποίο αναφερθήκατε. Τώρα θα πρέπει να εγκριθεί το σχέδιο ανάκαψης και το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την οικονομία, ε, βλέπουμε για άλλη μια φορά ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή. Διακυβεύεται το ίδιο το μέλλον των Ευρωπαίων. Το να υποχωρήσουμε σήμερα στις ε, διχόνοιες θα ήταν ε, βαρύ ιστορικό σφάλμα. Συμφωνήσετε την άλλη εβδομάδα και θα βοηθήσει αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου. Ε, σας είπα για την έντονη συνήγησή μου, αλλά δεν θέλω να σας κρύψω και την ανησυχία μου. Είπατε ότι θα πρέπει πρώτα να βρούμε τα χρήματα πριν μιλήσουμε για κράτος δικαίου. Επιτρέψτε μου να διαφωνήσω σε αυτό, διότι δεν μπορούμε να χτίσουμε την Ευρώπη με μία αμυγός λογιστική αντίληψη, αλλά όπως πολύ ωραία είπατε γύρω από ένα εγχείρημα, ε, ένα σχέδιο, ένα όραμα και ε, ισχυρές αξίες. Σήμερα είναι πάρα πολλοί ακόμα οι Ευρωπαίοι ηγέτες που εξακολουθούν να τορπιλίζουν αυτό το ευρωπαϊκό ε, ιδεώδες. Τρανό παράδειγμα ο κύριος Όρμπαν που είναι και μέλος του πολιτικού σας κόμματος, Ευρωπαϊκού Κόμματος, μόνο Θα πρέπει λοιπόν να διαψεύσουμε εκείνους που θέλουν να αλλάξουν την ιστορία. Θα πρέπει να αρχίσουμε να συνδέουμε την εκταμείευση των ευρωπαϊκών πόρων με το σεβασμό του κράτους δικαίου. Η πολιτική ευκαιρία είναι πρόδειλη. Αυτό ε, το πακέτο ε, του 1,83 θα πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε ως μοχλό για να μπορέσουν όλοι οι Ευρωπαίοι να ζουν σε ένα δίκαιο, ελεύθερο και ευημερούντα κόσμο. Έχετε ε, τη δύναμη να το κάνετε αυτό κυρία Καγκελάρη, μην απογοητεύσετε τους πολίτες. Ευχαριστώ. Για την ομάδα Ελευθερία και Δημοκρατία, ταυτότητα συγγνώμη και Δημοκρατία, ο κύριος Μόιτεν, παρακαλώ. Κυρία Καγκελάρη, κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Πολλοί άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουν από τη Γερμανική Προεδρία του Συμβουλίου πολιτική ευφυΐα και ε, ευρύτητα πνεύματος. Αυτό είναι απαραίτητο περισσότερο από ποτέ στην Ευρώπη. Αλλά ε, όλα αυτά που είπατε δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που σας είπα, αλλά με ιδεολογία, με άγνοια ε, και δυστυχώς εσείς δεν είστε ή ε, ευγενής ε, θεματοφύλαξ της Ευρώπης. Μάλλον νεκροθάφτης της Ευρώπης είστε. Τα ιδεώδη της Ευρώπης βασίζονται στην πολιτιστική ταυτότητα, στο αυτόβουλο και την ελευθερία του ατόμου. Όλα αυτά εσείς τα, καταπατάτε. Η πολιτιστική ταυτότητα της Ευρώπης, οι χριστιανοϊουδαϊκές της ρίζες, η πολυμορφία ε, ε, είναι κάτι που θέλετε εσείς να αντικαταστήσετε με ένα θολό πολυπολιτισμικό. Αυτό που οδηγεί, ε, το είδαμε με τα θλιβερά συμβάντα στη Διζόν και τη Σουτκάρδη. Ποια είναι τα συμφέροντα των ανθρώπων. Οι άνθρωποι πρώτα απ' όλα αισθάνονται Γάλλοι, Ιταλοί, Πόλοι, Ορονοί, Ούγγροι, Γερμανοί πρώτα και μετά μόνο Ευρωπαίοι ο διαφωτισμός οδήγησε σε μια λογική ε, που απαιτεί πολιτική με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και το σεβασμό του δικαίου. Εσείς έχετε μια χαόδη και ε, ε, άφρονα πολιτική και δημοσιονομική και νομισματική και έχετε ε, πάρει τις αποστάσεις σας οριστικά από τη λογική με όλα αυτά το χορό των δισεκατομμυρίων και περιορίζεται την ελευθερία των ανθρώπων, να αμεβιοποίηση χρέους, πράσινη συμφωνία ε, με άφρονη σπατάλη. Αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο των όσων πρεσβεύεται για να κάνει το χατήρι ε, του κυρίου Μακρόν και άλλων μεσογειακών ε, δίνει 500 δισεκατομμύρια η ε, κυρία Μέρκελ και έρχεται η κυρία Φόντερ Λάιν να προτείνει και άλλα να προσθέσει. Δεν είναι δικά σας τα λεφτά, είναι των φορολογουμένων που καλούνται τώρα να πληρώσουν τα σπαγμένα. Είναι ιδεολογία και μάλιστα καμία ελευθερία, βιασμό τη ελευθερία. Και μετά λέτε κυρία Μέρκελ ότι επιβάλλεται η Γερμανία να μην σκέφτεται μόνο τον εαυτό τη, αλλά να δείξει ένα δείγμα έκτακτη εξαιρετική αλληλεγγύη. Έχετε καταλάβει ότι κατά μέσο όρο οι Γερμανοί έχουν χαμηλότερο ε, εισόδημα από ότι οι Ιταλοί, ε, οι ε, Ισπανοί και οι Γάλλοι, ότι δεν έχουν σπίτια δικά τους, ιδιοκατοίκηση που υπάρχει σε χώρες της Μεσογείου. Μα τι παράλογη αντίληψη έχετε για την αλληλεγγύη. Και εσείς κυρία Μέρκε και η κυρία Φόντερ Λάιεν και η κυρία ε, Λαγκάρτ είναι μία τριάδα ε, ε, της φρίκης. Επιταχύνεται ε, αυτή την τρελή κούρσα την οποία έχετε αρχίσει. Γι' αυτό ε, δεν είναι απλώς κακή υπηρεσία στην Ευρώπη, αλλά είναι προδοσία στην ίδια την ευρωπαϊκή ιδέα και επίσης διακυβεύεται και υπονομεύεται ε, το μέλλον των μελλοντικών γενναιών. Η κυρία Κέλλερ από τους Πρασίνους, παρακαλώ. Uh, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μέρκελ, νομίζω ότι μπορώ να σας πω εξ ονόματος ε, της μεγάλης πλειοψηφίας ε, εδώ στο Κοινοβούλιο ότι σας καλωσορίζουμε θερμά εδώ, ανάμεσά μας. Και σίγουρα δείχνει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά όλοι κατά πλειοψηφία εργαζόμαστε για να βελτιώσουμε την Ευρώπη αυτή για τους πολίτες ακόμα και αν ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, διαφωνούμε για το πώς πρέπει να γίνει αυτό και θα συνεργαστούμε ακόμα πιο και θα εργαστούμε ακόμα πιο σκληρά για να εκπροσωπούμε πιο καλά την ε, ποικιλία τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ στο Κοινοβούλιο. Η Γερμανία αναλαμβάνει τα ενία της Προεδρίας σε δύσκολου καιρού και η κρίση του COVID-19 είναι μια ιστορική δοκιμασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή τη κρίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση παραλίγο να διασπαστεί σε μεμονωμένα τμήματα και η εμπιστοσύνη των πολιτών στην κοινή Ευρώπη ε, επλήχθη. Η κρίση όμως αποτελεί και μια ευκαιρία, μια ευκαιρία επιτέλους να οικοδομήσουμε αυτή την ε, Ευρώπη της αλληλεγγύης την οποία χρειαζόμαστε τόσο καταπηγόντως και αυτό επαφείται σε εσά, κυρία Καγγελάρια και στην κυβέρνησή σας. Θα πρέπει να αξιοποιήσετε την ευκαιρία αυτή για να μπορέσετε να ενώσετε εκ νέου την Ευρώπη και θα ήθελα να σας συγχαρώ για αυτό το γαλλογερμανικό ταμείο ανάκαμψης γιατί χρειάζεται τόλμη για να υπάρξει αλληλεγγύη και να μην επικρατήσουν οι εθνικοί προστατευτισμοί και αυτό είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε να το έχουμε πετύχει και πιο νωρί, αλλά τι να γίνει. Δεν είναι όμω τίποτα ακόμα σίγουρο. Χρειάζεται σκληρή δουλειά μέχρι ότου πραγματικά να δημιουργηθεί αυτό το ταμείο και χρειάζεται στενέ εταιρικέ σχέσει. Και εμεί οι πράσινοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε διατεθειμένοι να υποστηρίξουμε ένα φιλόδοξο τέτοιο σχέδιο για να υπάρχουν οι επενδύσει του μέλλοντο και να προλαμβάνει το έδαφο για μια οικολογική μεταρρύθμιση της οικονομίας. Ένα ταμείο το οποίο θα βοηθήσει τι πιο πολλέ ε, ευρωπαϊκέ χώρες χωρί να εκτοξεύσει τα χρέη κάποιων κρατών μελών για την αλλαγή του κλίματος, να μην επαναλάβουμε τα ασφάλματα του παρελθόντος, για να θέσουμε όρους ε, επιζήμιους από την Τρόικα. Αυτό θα υποστηρίξουμε εδώ στις Βρυξέλλες και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και αυτή η φρικτή κρίση του κορονοϊού καταδεικνύει ότι μπορούμε να δράσουμε από κοινού και να πετύχουμε στόχους. Αυτή την τόλμη, αυτή την αποφασιστικότητα τη χρειαζόμαστε και για την αλλαγή του κλίματος. Γιατί η αλλαγή του κλίματος δεν πρόκειται να περιμένουμε να συνέλθουμε από τα υπόλοιπα. Είμαστε η πρώτη γενιά η οποία πραγματικά νιώθει στο πετσί της ε, την αλλαγή του κλίματος. Ε, ε, είτε πρόκειται για τις θύελες, είτε πρόκειται για τις κατακλυσμούς, είτε πρόκειται για τις μεγάλες ξηρασίες. Και είμαστε και τελευταία γενιά, αν θέλετε, η οποία μπορεί κατά κάποιο τρόπο να ανακάμψει την αλλαγή του κλίματος. Έχουμε τις απαντήσεις για τις ανανεώσιμες ενέργειες, για το πράσινο μέλλον, για την βιώσιμη κυκλοφορία. Πρέπει όλα αυτά όμως να τα υλοποιήσουμε, να τα εφαρμόσουμε και η Γερμανική Προεδρία μπορεί να συμβάλλει προς την κατεύθυνση αυτή. Και βασικό είναι η κλιματική νομοθεσία και η κλιματική στόχη μέχρι το 2030. Θα πρέπει να είναι φιλόδοξη όμως, γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε να μας ακολουθήσουν και άλλες αυτή είναι η ιστορική μας ευθύνη και γι' αυτό λοιπόν ζητούμε από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση μείωση των αριθμών θερμοκίων 65% μέχρι το 2030. Και σας απευθύνω έκκληση να δείξετε τόλμη στην Ευρώπη, να δείξετε τόλμη και για την αλλαγή του κλίματος, γιατί ο κόσμος περιμένει τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποτραπεί η περαιτέρω κρίση στα πλαίσια του κορονοϊού και για το κλίμα. Χρειαζόμαστε όμω και εσά προ την κατεύθυνση αυτή, κυρία Εγκλάρια. Ευχαριστώ πολύ. Σα ευχαριστώ. Εκ μέρου τη ομάδα ΕΣΥΑΡ, ο πρόεδρος Ραφαέλ Εφίτο. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ την καγκελάριο Μέρκελ για την παρουσία της σήμερα εδώ στην Ολομέλεια όπου μας παρουσίασε τις προτεραιότητες της γερμανική προέδρια. Η Γερμανία αναλαμβάνει την Προεδρία ίσως την πιο δύσκολη στιγμή στην ιστορία της Υπήρους Υπήρου μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, βραδιπόρησε χωρίς πνεύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών και αδράνησε. Χθε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε τις προβλέψεις της ε, για την ανάπτυξη ε, μείωση κατά 8% στο, στην Ευρωζώνη, για την Ισπανία και την Αιλία μείωση ανάπτυξη κατά 8%. Πρέπει λοιπόν τώρα να δράσουμε. Ήδη μείναμε πίσω. Θα πρέπει την επόμενη εβδομάδα οπωσδήποτε να καταλήξουμε σε συμφωνία για τον προπολογισμό. Είναι απολύτω απαραίτητο. Θα πρέπει να φτάσουν τα κονδύλια το συντομότερο δυνατό στου Ευρωπαίου πολίτε, στι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει. Είναι καθήκον μα. Είναι ευθύνη μα. Και γι' αυτό δεν θέλουμε μία ε, συμφωνία προ τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Θέλουμε μία φιλόδοξη συμφωνία. Και η Γερμανία έχει τεράστια ευθύνη στη διάρκεια τη Προεδρία τη θα πρέπει να αφήσουμε κατά μέρου τους εθνικούς εγωισμούς και να επανέλθουμε στο πνεύμα αλληλεγγύης τη Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποφεύγοντας τα σφάλματα του παρελθόντος. Θα πρέπει επίσης να θέσουμε ένα τέρμα στη λιτότητα. Θέλουμε και πάλι να εμφυσίσουμε πνοή ενέργειας προς την ανάπτυξη. Θέλουμε μια θετική εμπορική πολιτική για να ανακάμψει η εσωτερική αγορά αλλά θέλουμε μια ισορροπημένη εσωτερική αγορά. Χρειαζόμαστε περισσότερη ευελιξία για τις κρατικέ ε, ενισχύσεις, κάτι όμως που δεν θα πρέπει να οξύνει περαιτέρω τις διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Επίση, είπατε ότι θα πρέπει υπεύθυνα να χρησιμοποιήσουμε του πόρου. Σωστά, αλλά να θέσουμε και κάποια όρια, όχι όμως εις βάρος εθνικής κυριαρχίας. Θέλουμε περισσότερη περιβαλλοντική αηφορία, σύμφωνα, χωρίς όμως να αμφισβητούμε την οικονομική επιβίωση των επιχειρήσεών μας. Αν δεν συμφωνήσουμε, όποια συζήτηση και αν κάνουμε για το μέλλον της Ευρώπης θα φανεί ω υποκριτική. Δεν χρειαζόμαστε κεντρικές διαταγές από τις Βρυξέλλες. Θέλουμε μια Ευρώπη που να σέβεται τα εθνικά προνόμια και τις εθνικές ευθύνες και αρμοδιότητες. Οι εθνικές κυβερνήσεις ε, που έχουν τη δημοκρατική νομιμοποίηση δεν θα πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ότι παραβιάζουν τον κράτος δικαίου επειδή δεν βρίσκονται στην ίδια γραμμή πλέψη με τις Βρυξέλλες στο ίδιο μήκος κύματος. Επίσης, χθε ε, η Ιταλό Υπουργός αναγνώρισε ότι πολλά κράτη-μέλη ε, εγκαταλείφθηκαν στη μοίρα του για την διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Οπότε δεν μιλούμε μόνο για τη μεταρρυθμίση του ασύλου. Θα πρέπει να ε, προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά μας σύνορα απέναντι στην ανεξέλεκτη μετανάστευση. Επίσης να καταπολεμήσουμε το εμπόριο ανθρώπων, τη λαθροδιακίνηση στην ε, Μεσόγειο. Και ο Ερδογάν χρησιμοποιεί εκβιασμό στο μεταναστευτικό ζήτημα. Είναι απαράδεκτο ε, η Τουρκία να διευρύνει τη σφαίρα επιρροής της στη Μεσόγειο εκμεταλλευόμενοι τη σιωπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία και με το Ηνωμένο Βασίλειο, να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία, να αναπτύξουμε το διεθνέ μα εμπόριο. Τεράστιε προκλήσει και θα τις υλοποιήσουμε σε συμφωνία με τους εταίρους μας. Θέλουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν θα φοβάται πια την Κίνα, που θα επιμείνει απέναντι σε κάποια κράτη-μέλη που κλείνουν το μάτι στο Πεκίνο και εγκαταλείπουν το Χονγκ Κόνγκ μόνο για να εξυπηρετήσουν τα οικονομικά του συμφέροντα. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε επίση τι αθέμητε πρακτικέ, να καταπολεμήσουμε τι επιθετικέ εξαγορέ. Ε, ο Ζωζέ Φρατσιγκέρ, ε, που είναι συμπατριώτης σα, ήταν πραγματικά ε, φίλο Ευρωπαίος και Ευρωπαίος πατριώτης. Όταν μιλούσαν άλλοι δεν διακόπτονται και δεν ενοχλούσατε. Είναι έλλειψη σεβασμού. Θα πρέπει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ακούγονται όλες οι φωνές. Ή η χώρα του Ζωζεφ Ράτσιγκερ που ήταν πραγματικός Ευρωπαίος πατριώτης. Ε, ε, πάπας που επανειλημμένος ε, δήλωσε ότι δεν μπορούμε να σκεφτόμαστε έναν κοινό ευρωπαϊκό οίκο όταν αρνούμαστε τις κοινέ μας αξίες και την ταυτότητά μας. Ελπίζω λοιπόν η Πρόεδρος να λάβει υπόψη και αυτό το δίδαγμα και να μην επαναλάβουμε τα σφάλματα του παρελθόντος. Σας ευχαριστώ. Εκ μέρους τώρα της ΓΚΟΕ, κύριος Χίρντερμαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Καγκελάρια. Με την Προεδρία αυτή έχετε μία δεύτερη ευκαιρία γιατί αυτή η Ευρώπη που πολλοί αναφέρουν σήμερα δεν ξέχασε ότι η απάντηση της Γερμανίας τότε στην κρίση την οικονομική ήταν η λιτότητα και τότε λοιπόν την πλήρωσαν το τιμήμα ε, ο κόσμος της ε, Νοτιάς Ευρώπης ε, με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών με χαμηλότερες συντάξεις, χαμηλότερους μισθούς. Αυτή την πολιτική λοιπόν, αυτή η πολιτική σχεδόν διάλυσε την Ευρώπη τότε και ελπίζω στην Προεδρία σας αυτή τώρα να καταφέρετε να διορθώσετε τα ασφάλματα τα αλλοντινά. Γιατί αντί για λιτότητα η πολιτική χρειάζεται μια πολιτική αλληλεγγύης σήμερα. Και κυρία Καγκελάρια, θα κριθείτε από το κατά πόσο θα μπορέσετε να ελέγξετε τις ε, κοινωνικές συνέπειες της πανδημίας, αλλά δεν μιλάμε καθόλου για αυτούς οι οποίοι τις τελευταίους μήνες κράτησαν ε, όρθια την κοινωνία, μέρα με τη μέρα, οι νοσοκόμοι, οι γιατροί, αυτοί που εργάζονταν στις, στα σούπερ μάρκετ, στα ψιλικατζίτικα, θα πρέπει να φροντίσουμε λοιπόν τους ανθρώπους αυτούς, να τους προστατεύσουμε από την φτώχεια, από τις επισφαλείς όρους εργασίας. Αυτό είναι καθήκον μας ως πολιτική και έχουν βαρεθεί πλέον οι πολίτες. Θα πρέπει πριν από το καλοκαίρι, καλοκαίρι να έχουμε μια απάντηση για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και για την ανάκαμψη. Και ακούγοντας εδώ κυρία Καγκελάρια και από τους εκπροσώπους της ε, πολιτικής σας ομάδας και από την Πρόεδρο Τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει αυτές οι, αυτά τα κονδύλια να συνδέονται με όρου επιτροφής πάντα δηλαδή και πάλι τέτοια αλληλεγγύη. Θα ήθελα να σα δώσω μία συμβουλή κυρία Μέρκελ. Ο Όλαφ Σόλτ πάντα μπλόκαρε διάφορε. Ε, ψηφιακέ ε, μεταρρυθμίσει και έκανε αναφορά στον ΩΣΑ. Η Γερμανία θα πρέπει να σταματήσει να μπλοκάρει σημαντικέ ε, αποφάσει στο Συμβούλιο πέρα από το ψηφιακό φόριο αυτή την ε, αναφορά χώρα αναχώρα. Θα πρέπει να σταματήσει λοιπόν να μπλοκάρει η γερμανική κυβέρνηση τέτοιες αποφάσεις. Αυτή η κοινωνική ανάκαμψη λοιπόν θα αποτελέσει ένα σημαντικό έργο για το μέλλον τη Ευρώπη. Χρειάζεται μια πολιτική για το κλίμα που θα ακολουθεί τη Συμφωνία του Παρισιού και αυτή η Πράσινη Συμφωνία όπως την έχετε παρουσιάσει σήμερα, όπως την παρουσιάσει η κυρία Φόντερ Λάιεν είναι απέχει πάρα πολύ από την Συμφωνία του Παρισιού. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λοιπόν και μια συμφωνία με τον Μερκοσούρ. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπως και εγώ, ότι ο ακραίος Πολσονάρου της Βραζιλίας ε, καταστρέφει τα παρθένα δάση του Αμαζονίου και θεωρώ ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε συμφωνία με ακροδεξιές και εξτρεμιστικές δυνάμεις. Αναφέραμε τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν θα έχουν καμία σημασία γιατί στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτές οι αξίες πνίγονται καθημερινά με τους ανθρώπους αυτούς που πνίγονται στη Μεσόγειο. Τους ανθρώπους αυτούς δεν τους βοηθάμε με διάφορες ε, συμφωνίες ε, νοσηρές με ληστάρχους και ακραίους πολιτικούς. Αυτή η εμπιστοσύνη λοιπόν στην ευρωπαϊκή δημοκρατία μπορεί να ενισχυθεί κυρία Μέρκελ, μπορείτε εσείς να την ενισχύσετε αν περιορίσετε την επιρροή των λόμπι στο Συμβούλιο και αν τονίζετε και το θέμα της διαφάνειας στο Συμβούλιο, το είπατε άλλωστε, η διαφάνεια είναι το leitmotiv της Προεδρίας σας. Αυτό θα είχε μεγάλη επιτυχία. Αυτό θα είχε, ήταν ένα σκόπιμο βήμα προκειμένου να ανακάμψει η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και να ενωθούν τα κράτη-μέλη με στόχο μια οικονομική, κοινωνική και οικολογική Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Από τους για εγγεγραμμένους, ο κύριος Σόνεμπορ, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλή όρεξη κυρία Μέρκελ. Ποιος θα βγάλει ε, από την κρίση ε, την Ευρώπη αν όχι η Γερμανία στην Ευρώπη υπάρχει μια νοσταλγία ε, να ε, ε, υποταγούν στη γερμανική κυριαρχία. Γιατί τους έπιασε αυτό τώρα και όχι πριν από τα 80 χρόνια. Θα είχαμε γλιτώσει από πάρα πολλά δεινά. Με τον Όρμπαν τι κάνετε, δεν πάτε και πολύ καλά και στην Ευρώπη. Θέλετε να απαγορεύσετε την κλιματική αλλαγή και θα μας καρχάζουν οι Κινέζοι. Θέλετε να ε, χαλιναγωγήσετε την μετανάστευση για να επηγαίνετε τους μετανάστες εκεί που δεν φαίνονται. Ούτε εσείς ούτε τα 750 δισεκατομμύρια σας ε, θα επιτρέψουν να ξανανεύει η ομάδα του Αμβούργου στην πρώτη εθνική. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ζήτησε το λόγο και πάλι η κυρία Μέρκελ μετά τον πρώτο γύρο τοποθετήσεων των προέδρων των πολιτικών ομάδων. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστώ όλους ε, κύριους που μου δώσατε ευχές το μαζί, το από κοινού, δεν αφορά φυσικά τα κράτη-μέλη, αλλά και τη συνεργασία μόνο και τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πολύ διαφορετικές οι απόψεις ε, ακόμα και ας προς το ζητούμενο και στο Κοινοβούλιο. Άρα τη λύση δεν θα πρέπει να τη βρούμε μόνο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, θα πρέπει όλοι να κάνουμε βήματα, ο καθένας προς την κατεύθυνση του άλλου, για να προχωρήσουμε. Αναφέρθηκα στο κράτος δικαίου ε, και στα θεμελία δικαιώματα συνειδητά και για τη Γερμανική Προεδρία στην Ευρώπη. Ε, αυτά είναι απόλυτη προτεραιότητα. Παρόλα αυτά, όμως, θα πρέπει να δημιουργήσουμε τη βάση για να μπορέσουμε να δουλεύουμε και εδώ ε, ανήκει και το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ήδη από τώρα θα ήθελα να πω ότι ε, και το συζήτησαμε και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ με το Κοινοβούλιο χρειαζόμαστε ένα πνεύμα ε, συμβιβαστικό. Το είπε και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, γιατί ακόμα οι απόψεις ε, αποκλίνουν πολύ μεταξύ των κρατών μελών. Κάτι που είναι απαράδεκτο είναι ε, κάτι απόψεις που ακούμε που είναι υπερβολικά σίγουρες για την αλήθεια ε, και ε, δεν βοηθούν τέτοιες υποτιμητικές εκφράσεις για τους υπολείπους ούτε εξυπηρετούν κανένα σκοπό. Μίλησε ο κύριος Βέμπερ για τους ιδίους πόρους. Το κατανοώ ότι αυτό είναι αμέλημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από την άλλη όμως υπάρχουν κάποιοι πόροι που τώρα ε, μπορεί να θεωρούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήδη οι πόροι είναι προγραμματισμένοι στους εθνικούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει λίγο να προσέξουμε γιατί είναι και δύσκολη η οικονομική καιρή. Ε, το ήδη οι και δεν μιλώ εδώ για τη φορολόγηση των ε, ψηφιακών εταιριών, αλλά ε, να μην δημιουργούμε τεχνητές λανθασμένες εντυπώσεις επιβολής νέων φόρων ή αύξησης της φορολογίας, γιατί αυτό θα ήταν δύσκολο. Ε, για το ψηφιακό φόρο βεβαίως είναι πάντα καλύτερο αν καταφέρουμε ένα φόρο να τον συμφωνήσουμε παγκόσμια και διεθνώς. Και το θεωρώ πολύ ε, θεμητό να περιμένουμε πρώτα τις εργασίες του ΟΟΣΑ, γιατί όλα τα υπόλοιπα ενδεχομένως να μας οδηγήσουν σε δύσκολους εμπορικούς ε, πολέμους. Το έχουμε ξαναδεί στην Ευρώπη. Αν όμως δεν διαφαίνεται διεθνής λύση, τότε θα πρέπει σοβαρά να προβληματιστούμε, να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε μία λύση για την Ευρώπη, γιατί δεν επιτρέπεται ε, ένας κλάδος ε, δημιουργίας ε, αξίας ε, στο ψηφιακό κόσμο να ξέρετε από τη φορολογία και μάλιστα διαρκώς αυξανόμενος. Έχουμε κάνει καλά βήματα και για τη διαφάνεια σε φορολογικούς παραδείσους. Δυστυχώς αυτό με το ψηφιακό φόρο δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Και ένα τελευταίο, θα πρέπει να κάνουμε σαφή διάκριση ανάμεσα στην κρίση του ευρώ ή την χρηματοπιστωτική κρίση, την παγκόσμια που ζήσαμε, και τη, τη σημερινή πανδημία. Δεν χωράει καμία αμφιβολία και είναι αδιαφυσβήτητο ότι όλοι μας, όλα τα κράτη-μέλη, ε, είμαστε σε διεθνή ανταγωνισμό και μπορούμε να ε, βιώνουμε ε, την οικονομία όπως θέλουμε αν ε, ε, δεν κάνουμε το ε, μοντέλο μας ευάλωτο, αν δεν είμαστε εκτεθειμένοι σε υπερχρέωση. Καλό ήταν αυτό που έγινε για τις μεταρρυθμίσεις και φυσικά το αντίβαρο ήταν η αλληλεγγύη. Εδώ σκέφτομαι τον ESM τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό σταθερότητα και τα άλλα μέτρα. Αλλά τώρα εδώ δεν πρόκειται για κρίση χρέους, πρόκειται για ένα ιό ε, ε, που μας βρήκε όλους με πολύ διαφορετικό τρόπο κάθε κράτος ε, και κανείς δεν φέρει ευθύνη. Και εδώ χρειάζονται τελείως διαφορετικά εργαλεία και τελείως διαφορετικές απαντήσεις. Γι' αυτό προωθώ αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Κασπάρη, παρακαλώ για ένα λεπτό. Αξιότιμη κυρία Εν ώψη των αρνητικών οικονομικών εξελίξεων στην Προεδρία, θα ήθελα να μην συνεχίσουμε όπω ε, ω τώρα. Γιατί έχουμε επιχειρήσει οι οποίε βρίσκονται στο χείλο τη καταστροφή. Έχουμε ε, εργαζόμενου ε, που είναι άνεργοι. Θα πρέπει να του δώσουμε μια προοπτική, κάποια αισιοδοξία. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τι παλιέ δομέ και να τι διατηρήσουμε μάλιστα με τεχνητού τρόπου. Θέλουμε λιγότερε δηλαδή δαπάνε. Αντί για λιγότερε δαπάνε, θέλουμε πιο πολλέ επενδύσει για το μέλλον και θα πρέπει να τα δαπανίσουμε τα χρήματα αυτά και να αποφασίσουμε τι γίνεται και με τις επιστροφές σε ό,τι αφορά δηλαδή τον προπολογισμό. Δεν μπορούμε απλά να το μειώσουμε. Πώς θα επενδύσουμε στην κοινοτομία, πώς θα διαμορφώσουμε την Ευρώπη και θα έχουμε ασφάλιστα σύνορα. Θέλω να μην μιλάμε μόνο για χρήματα, αλλά να μιλάμε και για την πολιτική ένωση, να συνεχίσουμε να την αναπτύσσουμε, να ενισχύσουμε την Ευρώπη σε θέματα όπως ε, η υγεία, ε, το κλίμα, το εξωτερικό εμπόριο. Όλα αυτά τα θέματα είναι θέματα στα οποία χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη. Και σας εύχομαι λοιπόν ε, κάθε επιτυχία στην ατζέντα της Προεδρίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριος Γκάιερ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Καγκελάρια κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Η ανάκαμψη της ε, ευρωπαϊκής ε, κοινωνίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας είναι κοινό έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή θα τα καταφέρουμε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ή θα τα καταφέρουμε καθόλου. Το είπατε αυτό κύριε Καγκελάρια και η ανάπτυξη δυναμικού ανθεκτικότητα στο εσωτερικό του ευρωπαϊκού προπολογισμού είναι ένα, μέλλον, ένα βήμα μελλοντοστραφέ, αν θέλετε. Θα πρέπει να το αναλάβει αυτό από κοινού το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και έχουμε παραδείγματα στο ευρωπαϊκό Προπολογισμό, σε ό,τι αφορά τη ε, κοινή διαμόρφωση των δαπανών, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Θέλουμε διαφάνεια, διαφάνεια και προ τον κόσμο για το πακέτο ανάκαμψη και πώ θα χρησιμοποιηθεί. Χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν κατεπηγόντω το ζητώ, κυρία Καγκελάρια, να ζητήσετε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να έχει δικαίωμα στην απόφαση και να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα στο έπακρο από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Σασμάνη για ένα λεπτό. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και θα ήθελα να καλωσορίσω την καγκελάρια κυρία Μέρκελ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου έχουμε προφανώ υψηλέ προσδοκίε από τη Γερμανική Προεδρία. Η Ευρώπη θα πρέπει να πετύχει συμφωνία για το του ζωνικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψη ε, εν το μέσο μια ε, κρίση ενό προηγουμένου. Ωστόσο, δεν χρειαζόμαστε απλά ανάκαμψη, χρειαζόμαστε μια ευφυή ανάκαμψη. Η Ευρώπη θα πρέπει να καταδείξει τη φιλοδοξία να εξέλθει πιο ισχυρή από την κρίση αυτή. Αυτή είναι η χρονική στιγμή να δοθεί ε, μια πνοή και μια ανάσα στι οικονομίε μα με βιώσιμο τρόπο. Είναι επίση η στιγμή να ενισχυθεί η δημοκρατία η Ευρώπη επιμένει να ενισχύει τους όρους για το κράτος δικαίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το σκέλος αυτό και ελπίζω να συμφωνεί μαζί μου η Καγκελάριος και θα ήθελα να ακούσω λοιπόν πώς η Γερμανική Προεδρία θα α, πετύχει την ρεσιμότητα αυτή. Και έχουμε και άλλες προκλήσεις φυσικές στον ορίζοντα Χρειαζόμαστε πρόοδο στο πακέτο μετανάστευσης, να αποφύγουμε ένα σκληρό Brexit χωρίς ε, συμφωνία και να καθοδηγήσουμε την Ευρώπη σε έναν κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Θα θέλαμε λοιπόν να σας τίνουμε χειρά βοηθεία για να σας βοηθήσουμε σε αυτές τις σοβαρές προκλήσεις. Κυρία Μέρκελ, να σας κοιτάξω στα μάτια και να σας ρωτήσω, θέλετε μαζί μας να ανανεώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό, κύριο Άνεμανς. Συνάδελφοι, σε αντίθεση με αυτά τα οποία θα περιμέναμε, η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Brexit δεν χαμήλωσε καθόλου τον τόνο τον οποίο μιλούσε και όλα αυτά βλέπουμε ότι παθάει στον γκάζι και θέλει να επιμένει σε ό,τι αφορά αυτό το ευρωπαϊκό νοητοποιητικό κράτο. Και ε, αυτά φυσικά χωρίς να λαμβάνει υπόψη την ε, ευρωπαϊκό πληθυσμό, τον κόσμο της Ευρώπης. Κυρία Μέρκελ, νομίζω στην Προεδρία αυτή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρείται ότι είναι ευτυχής ε, αυτή η χρονική στιγμή και ότι είναι, ε, θα δώσετε μια καλή καμπή στην κρίση. Αλλά να σα πω το εξή ότι είναι πάρα πολλοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επικριτικοί σε ό,τι αφορά αυτέ τι φεντεραλιστικέ τάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τώρα ανησυχούν ε, ακόμα πιο πολύ τώρα που οι Γερμανοί θα ε, βάλουν το βάρος τους υπέρ της φεντεραλιστικής αυτής διαμόρφωσης. Πρόκειται για επικριτικού πολίτε, γιατί θεωρούν αυτοί οι πολίτε ότι είναι διπλή απειλή τη Προεδρία σα. Και θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σα σε αυτό. Δεν θα πρέπει λοιπόν να καταπιέσουμε όλε αυτέ τι επιχειρήσει. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κυρία Ντελβό. Καγκελάρια, μπορεί να είμαστε πεπισμένοι φιλοευρωπαίοι, ακόμη και φεντεραλιστές ε, και να έχουμε ταυτόχρονα επίγνωση ότι αντιμετωπίζουμε πραγματικά πλανητικής διάσταση, τεράστια προβλήματα, αλλά έχουμε και ανησυχίες για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε το Brexit και δύο χώρε μέλη αξιοποιούν τι αδυναμίε της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ε, παράλυση που έχουμε καταλήξει για να υποβα... επιβάλλουν αυταρχικά καθεστώτα και να ελέγξουν, να προσπαθήσουν να ελέγξουν τη δικαιοσύνη, τα μέσα μαζική ενημέρωση, την αντιπολίτευση. Αυτό θα είναι πολύ κακό παράδειγμα γιατί δίνουμε την εντύπωση ότι Μόνο προειδοποίησει ε, είναι ε, η απάντηση σε τέτοιες παραβιάσεις. Μα υπενθυμίσατε την ιστορία και πραγματικά είναι αξιόλογη η πορεία σας ε, άμεμπτη και η επιρροή σας μεγάλη. Γι' αυτό θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είναι υποδειγματική γερμανική προεδρία, ε, θαραλέα, πιο θαραλέα από τη φιλανδική ε, για, τα θέματα του κράτους δικαίου και θα ήθελα να μην ε, βάλετε τα οικονομικά και διπλωματικά συμφέροντα πάνω από τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριος Κούσμιου, και ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καγκελάρια, κύριε Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η χώρα σας δεν είναι μόνο μεγαλύτερο συνεισφέρον στον ε, ευρωπαϊκό προϋπολογισμό πάνω από 300 ε, δις, αλλά και ο μεγαλύτερος δικαιούχος της εσωτερικής αγοράς ε, πάνω από πολλαπλάσιο από τις συνεισφορές που κάνετε. Και είναι σημαντικό λοιπόν να, να διεκδικείται αλληλεγγύη προς χώρες που πλήγησαν περισσότερο ε, από το, στα Πάνω από ένα δισεκατομμύριο δώσατε κρατικέ ενισχύσει στι επιχορηγήσει. Αν όμω η οικονομική κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση παραταθεί, η γεωργική οικονομία που στηρίζεται στι εξαγωγέ πολύ πιθανόν να πληγεί και εκείνη στο μέλλον. Γι' αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε το συντομότερο δυνατό τι δημοσιονομικέ διαπραγματεύσει και να εγκριθεί το σχέδιο ανάκαμψη ε, ήδη φέτο για να βοηθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη. Επίση, η κοινωνική γεωργική πολιτική είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, τη θέση των γεωργών που για 500 εκατομμύρια Ευρωπαίου εξασφάλισαν επιστηστική ασφάλεια. Θέλουμε να ενισχύσουμε το γεωργικό προπολογισμό την επόμενη επταετία να εξασφαλίσουμε τους αγρότες και να τους ε, αναμίξουμε και αυτούς στην υλοποίηση της Νέας Πράσινης Συμφωνίας. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό, κυρία Ρόζα Νταμάτο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Έχω μόνο ένα λεπτό για να απευθυνθώ στην Καγκελάριο, στη γυναίκα που θεωρείται το αφεντικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυρία μάλιστα Φοντερ Λάιεν, πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, διατέλεσε υπουργό της κυβέρνησής σας. Τώρα και οι δύο μπορείτε να διορθώσετε τα λάθη που έχετε διαπράξει. Ε, το COVID έκρουσε τον κόδωνα, τον κόδωνα του κινδύνου. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε το σχέδιο ανάκαμψη ε, με πολλά κονδύλια το συντομότερο δυνατό, μέσα στο χρόνο και να μην ε, υποχωρήσουμε σε σχέση με την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και το ΠΔΕΛΤΑΠΗ είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, ε, θέλουμε ιδίου πόρου. Η Ιταλία επλήγει ε, ιδιαίτερα το υγειονομικό τη σύστημα ε, από την λιτότητα. Οπότε θα πρέπει ε, να, όπως διδαχτήκαμε από τους Έλληνες, ε, δεν θα πρέπει να εκποιήσουμε ε, τον κρατικό πλούτο και να ιδιωτικοποιήσουμε τις επιχειρήσεις μας. Δεν θα πρέπει να αφήσουμε τις κινέζικες επιχειρήσεις να εξαγοράσουν τις στρατηγικές μας επιχειρήσεις και να αναλάβουν τους στρατηγικούς μας κλάδους. Επίσης δεν θα πρέπει να σιωπήσουμε και να μην αναγνωρίσουμε τις θυσίες των Ευρωπαίων πολιτών. Και επίση, η εσωτερική αγορά θα πρέπει να ευνοεί τους πάντες, θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα στους φορολογικούς παραδείσους και το συντομότερο δυνατό να κρίνουμε έναν ε, ενιαίο ευρωπαϊκό κατώτατο μισθό και επίσης ε, να καταπολεμήσουμε το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων ε, να σταματήσουμε να χρηματοδοτούμε τα ορυκτά καύσιμα και τα συμφέροντα και θέλουμε θάρρος και φιλοδοξία και για τις εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Η κυρία Γκιόρη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να ε, βοηθήσετε την ανάκαμψη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γερμανία είναι σε θέση με την Προεδρία της να ξανακάνει ε, πάλι ισχυρή την Ευρώπη. Ουγγρική Προεδρία ε, είχε θέσει ως ε, σύνθημά της ε, τα μικρά βήματα που θα οδηγήσουν σε μεγάλη πρόοδο. Τώρα ήρθε η ώρα ε, με συνεργασία να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Χρησιμοποιήστε την ισχύ σα για, να, για να συμφωνήσουμε σε έναν ισορροπημένο προπολογισμό, να ενισχύσουμε την πολιτική συνοχή που ήταν επιτυχημένη στο παρελθόν και να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα. Αντιλαμβάνεστε τι ιδιαιτερότητε των χωρών τη Ανατολική Ευρώπη και μπορείτε να βασιστείτε σε εμά, αλλά και εμεί θέλουμε να υπολογίζουμε σε εσά. Σα αφήσουμε πίσω τι διαφορέ μα, σα αφήσουμε πίσω τι ε, οι ιδεολογικές μας ε, διαφορές και τον ψυχολογικό πόλεμο που κάνουν μερικέ φορές τα κράτη-μέλη μεταξύ τους. Επίσης, για το κράτος δικαίου θα πρέπει να ξεπεράσουμε τις προκαταλήψεις. Με βάση τις συνθήκες θα πρέπει να ισχύουν οι ίσες προϋποθέσεις για όλα τα κράτη-μέλη και θέλουμε την υφαλιότητα της Γερμανίας για να συμφωνήσουμε με το Ηνωμένο Βασίλειο και να αποδεχθούμε το γεγονό ότι επέλεξε την αποχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνούμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι από του σημαντικού πολιτικού και οικονομικού μα εταίρου. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καγκελάρια, η Γερμανική Προεδρία ξεκινά σε πολύ χαλεπούς καιρούς. Η Ευρώπη έχει γονατίσει από την πανδημία COVID-19 και τις ε, κοινωνικο-οικονομικές συνέπειες που προκάλεσε. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια απάντηση και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και των προκλήσεων. Αναλαμβάνετε την ε, Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, λίγες μέρες μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που εκλήθη να δεχτεί το σχέδιο ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μπορούμε να υπαναχωρήσουμε σε σχέση με το σχέδιο αυτό. Θέλουμε όντως να οικονομήσουμε την Ευρώπη που μας περιγράψατε. Μια εύρωστη, ρωμαλαία και αλληλέγγυη Ευρώπη αν θέλουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει τα, οι προτεραιότητες του εξαμήνου να βρεθούν στο επίκεντρο της Ευρώπης αυτής. Μας περιγράψατε τις προτεραιότητες της ε, Γερμανικής Προεδρίας. Το Συμβούλιο υπάρχει, αλλά υπάρχει ταυτόχρονα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που εξελέγει άμεσα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι λοιπόν που θα υπολείπεται των προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δεν θα δίνει ε, ελπίδες στου Ευρωπαίου πολίτες. Η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το σημείο φετηρία και δεν θα πρέπει να είναι το σημείο προορισμού. Δεν θέλουμε άλλες εκπτώσεις και άλλες ε, περικοπές κονδυλίων. Κάθε μήνα που χάνουμε χάνουμε και ποσοστά στο, στην άψη του ΑΕΠ μας. Σας εύχομαι καλή τύχη και καλή επιτυχία και δεν το λέω ηρωνικά. Θέλουμε τα διορατικότητα και θάρρος και θα βρεθούμε στο πλευρό σας αν τα επιδείξετε όλα αυτά. Σας θερμό παρακαλώ να μην υπερβαίνετε το χρόνο σας. Η κυρία Μπέρ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Καγκελάρια. Όποιος ε, σήμερα δεν είναι απόλυτο θα χάσει. Η Ευρώπη χρειάζεται τόλμη, ε, ταχύτητα και ε, θέληση για μεταρρυθμίσεις. Πολλά μπορεί να πετύχουμε με τα χρήματα, αλλά όχι όλα. Ας μην θεωρήσουμε ότι με το χρήμα μπορούμε να αντισταθμίσουμε βασικές και θεμελιώδεις και διαφορετικέ ελλείμματα. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το πακέτο για τον κορονοϊού έχει πάρα πολύ όγκο και πολύ πολύ λίγο μέλλον. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την Ευρώπη προς τα μέσα με μια με ένα προπολογισμό ο οποίο θα είναι υπέρ τη καινοτομία, τη καινοτομία και τον εξυγχρονισμό με έναν μηχανισμό κράτου δικαίου για μια δημοκρατία, για μια δημοκρατική ένωση και για μια νέα πολιτική για το άσυλο και τη μετανάστευση χωρί την αρχή του Δουβλίνου αλλά με ευρωπαϊκό πόλο έλξη, για μια πιο ανθρωπιστική Ευρώπη και πιο ειλικρινή Ευρώπη και πιο ισχυρή προ τα έξω με μια Ευρωπαϊκή Ένωση με μια ισχυρή φωνή και με πιο έντονη παρουσία σε όλο τον κόσμο με τις αντίστοιχες θεσμικές ε, δυνάμεις. Ε, μια πολιτική, λοιπόν Ευρώπη δεν θα πρέπει να είναι διασπασμένη και δεν θα πρέπει να είναι και χρεωμένη. Αυτή θα πρέπει να είναι η φιλοδοξία στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Μάντισον, για ένα λεπτό. Äh, Κύριε Μέρκελ, σας άκουσα με μεγάλη προσοχή τονίσατε την ενότητα και την αλληλεγγύη. Πώς μπορούμε όλα αυτά να τα κατανοήσουμε όμως τη στιγμή που η Γερμανία σε διάφορες περιστάσεις έχει διευκρινίσει ότι η αλληλεγγύη ισχύει με πληκτικό τρόπο. Θέλετε καλές τιμές για το αέριο, θέλετε ευνοϊκές τέτοιες τιμές. Αγνοείτε Επίσης, ε, τα δικαιώματα των εταίρων σας στον τομέα της ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώς λοιπόν βγαίνετε και μιλάτε για αλληλεγγύη όταν σήμερα πολλοί Ευρωπαίοι αγρότες, δύο τρίτα υποστηρίζουν, ε, μάλλον ε, η Γερμανία είναι κατά της υποστήριξης των αγροτών γιατί πολύ απλά δεν θέλουν να χάσουν το τμήμα αυτό της ενιαίας αγοράς. Αυτή η αλληλεγγύη λοιπόν τι σημαίνει για σας. Σημαίνει ότι η Γερμανία ελέγχει τη μετανάστευση στα σύνορα και όταν ένα πρόβλημα διωγγώνεται πολύ απλά βάζετε ποσοστώσεις. Εγώ τέτοιου είδου Ευρώπη δεν τη θέλω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. μισή λεπτό ο κύριο Γκίγκολ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Καγκελάρη, θα σας προκαλέσει έκπληξη, αλλά σας συγχαίρω. Σας συγχαίρω γιατί με την ε, γαλλογερμανική πρόταση για το Ταμείο Ανάκαμψης ε, σπάσατε τρία ταμπού της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής ως τώρα. Αυτά τα τρία ταμπού λοιπόν είναι το εξή. Οι επιδοτήσεις αλληλεγγύης και επενδύσεις σε ό,τι αφορά αυτά που λέγονται για την Ένωση των Μεταφορών. Κατά δεύτερον, η κοινή χρέωση για τις μεγάλες επενδύσεις αντί για την αιώνια αυτή συζήτηση για ευρωομόλογα και τέλος την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Φόρου. Αλλά κυρία Καγκελάρια, αυτό αποτελεί μια στροφή 180 μοιρών από την πολιτική που ασκήσατε στην ευρωπαϊκή αυτή, στην κρίση του ευρώ. Το ερώτημα είναι τι θα ακολουθήσει γιατί όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να είναι πέρα από κενά λόγια και πράξεις. Ναι, χρειάζεται λοιπόν αντιμετώπιση της κρίσης. Αυτό θα είναι κάτι το προσωρινό, αλλά η αλληλεγγύη θα πρέπει να αποτελέσει μια μακροπρόθεσμη αξία στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν θέλουμε λοιπόν μόνο μια φορά να κάνουμε πολιτική αλληλεγγύη, αυτή η στροφή 180 μοιρών θα είναι μια πυρουέτα και μόνο. Και γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να αφήσουμε την Ευρώπη να διαλυθεί περαιτέρω με την ε, κρίση του COVID-19. Το θέμα είναι, θα δούμε λοιπόν τώρα, κυρία Μέρκελ, κατά πόσο είσαστε μόνο υπεύθυνοι για τη διαχείριση κρίσεων ή αν είσαστε αρχιτέκτον της Ευρώπης. Μόνο μία διαρκής, μακροπρόθεσμη τέτοια διαμόρφωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης θα κάνει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση έτοιμοι για το μέλλον. Χρειάζεται απόλυτη σαφήνεια και απόλυτη δέσμευση από πλευρά σα. Ευχαριστώ κύριος Γκόικινγκ για ένα λεπτό παρακαλώ. Ε, Ψηλέ προσδοκίες ε, έχει η Γερμανική Προεδρία στους ώμους της, δεν χωρά καμία αμφιβολία. Και ρίχνει τη σκιά και η COVID-19 και οι επιπτώσεις της. Μαζί θα πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και να την καταπολεμήσουμε. Είναι σαφές. Κοιτάξτε ε, και το θέμα ε, των ομολόγων ε, σχετικά με αυτό. Η Γερμανία σε αυτή την Προεδρία έχει κάνει σημαία της στην κοινωνική πολιτική. Εγώ είμαι πρόεδρος ε, κόμματο της οικογένειας στη Γερμανία θα πρέπει επιτέλους να ασχοληθούμε με την εγγύηση για τα παιδιά με ένα επίδομα τέκνων για να βγουν ε, πολλά παιδιά, ε, εκατομμύρια από τη φτώχεια, από την κρίση της COVID και πραγματικά η κοινωνία μας να είναι προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Γιατί μια ισχυρή Ευρώπη που χρειαζόμαστε ε, παγκόσμια βασίζεται στην ισχυρή οικογένεια. Και εκεί ποντάρω εγώ στη Γερμανική Προεδρία και ελπίζω στην υποστήριξή σας όχι ωραία λόγια και κυριακάτικα κηρύγματα. Επιτέλους να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια των οικογενειών και την παιδική φτώχεια. Ο κύριος Πούτσδεμον παρακαλώ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κυρία Καγκελάρη, τα προβλήματα της νεολαίας δεν είναι μόνο οικονομικά. Βεβαίως έχουμε κρίση και θα πρέπει σήμερα ε, να ε, ξεπεράσουμε τις ανισότητες ε, και τη φτώχεια γιατί είναι οι συγκρούσεις του μέλλοντος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προλαμβάνει τις κρίσεις. Τα προβλήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η δημοκρατία. Το να βγούμε από την οικονομική κρίση για να μπούμε σε μια κρίση δικαιωμάτων και ελευθεριών δεν θα σώσει την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε το πρόγραμμα της ανάκαμψης να συνδέεται με τη δημοκρατική εδραίωση. Θα πρέπει να ζητήσουμε και να απαιτήσουμε χώρες που αμφισβητούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως είναι η Ισπανία, να σέβονται το κράτος δικαίου. Να σταματήσει η δίωξη των ιδεών, οι αυθαίρετες φυλακίσεις πολιτικών, αντιφρονούντων, καλλιτεχνών ή δημοσιογράφων αυτό είναι ηθική υποχρέωση και νομική υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν μπορεί πλέον να αποφεύγει. Η κυρία Μονσεράτ, ευχαριστώ πρόεδρε. Στην Ισπανία, ενώ ε, ζούμε ε, τον πόνο από την απώλεια χιλιάδων ε, πολιτών και αντιμετωπίζουμε τη χειρότερη οικονομική και ε, κοινωνική κρίση μας έδειξε ο ιός ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να εξυγχρονιστεί και η Ισπανία και η Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ισχυρούς ηγέτες σήμερα στην Ευρώπη. Φόντερ Λάιεν στην Κομισιόν, ε, Μέρκελ στη Γερμανική Προεδρία είναι ελπίδα για εκατομμύρια Ευρωπαίων με ισχυρή στήριξη ε, στο Ταμείο Ανάκαμψης το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στηρίζει και χειροκροτεί την Προεδρία και τα προγράμματα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι θα προστατεύσουμε την υγεία μας, θα αναζωογονηθεί η οικονομία και ο παραγωγικός συστός, θα δημιουργηθούν δουλειές που είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική. Η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να συνοδεύεται από φιλόδοξες εθνικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε η Ευρώπη και η Ισπανία να είναι ε, πιο ανταγωνιστική, με βιομηχανία, με ψηφιακή οικονομία, χωρίς να απεμπολούμε ποτέ την ισότητα και την ελευθερία αν πετύχει η Ευρώπη θα αποτύχουν οι εθνικισμοί ε, και οι λαϊκισμοί. Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως μεγάλοι ευρωπαϊστές που είμαστε και δημοκράτες θα είμαστε στο πλευρό σας. Ο κύριος Ερτούγκ για ένα λεπτό. Παρακαλώ Ισμαήλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμη κυρία Καγκελάρια, καλώς ορίσατε στο σπίτι της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας. Χαίρομαι που σας βλέπω. Στο πρόγραμμά σας γίνεται μεγάλος λόγος για την προστασία του κλίματος και την ψηφιοποίηση. Ένα λοιπόν είναι σαφές, χωρίς τεχνολογία δεν υπάρχει πράσινη συμφωνία. Ο μετασχηματισμός ε, έχει μεγάλες ευκαιρίες και θα πρέπει να τις δούμε. Ε, ε, γαλλογερμανική πρωτοβουλία yeah, μπορεί να μας βοηθήσει να σπάσουμε παγκοσμίω τα μονοπόλια. Στόχος μας θα πρέπει να είναι παγκόσμια να είμαστε ηγέτες τεχνολογικά, ιδιαίτερα στη τεχνολογία υδρογόνου και ε, στις ε, μπαταρίες για τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Η στρατηγική του υδρογόνου παρουσιάστηκε σήμερα και σε ευχαριστώ κυρία Φόντερ Λάιεν. 10 δισεκατομμύρια ευρώ προγραμματίζονται στην επόμενη δεκαετία. Αλλά και οι μπαταρίες είναι πολύ σημαντικό και εδώ είναι ο Μάρο Σε ευχαριστώ γιατί είναι δικό σου τέκνο αυτό. Αλλά και εδώ, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία. 250 δισεκατομμύρια ευρώ ε, ε, είναι η αξία του 2025 και 5 εκατομμύρια οι νέε θέσει. 100 δι έχει ήδη ε, εξαγγείλει η βιομηχανία ότι θα επενδύσει. Κυρία Επίτροπε, ε, κυρία Πρόεδρε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρία Μέρκελ Πρέπει να σας πω ότι σα σήμερα πριν από 30 χρόνια έγινε η Γερμανία παγκόσμιο πρωταθλητή στο ποδόσφαιρο. Και ε, είναι γούρι, η κυρία Μίλλερ. Αξιότιμη κυρία Καγκελάρια, ως πολιτικό ε, πολιτικός από τα συντήματα τα γεωργικά της ε, Renew Europe, σας ζητώ να υποστηρίξετε την γεωργία. Στην κρίση COVID οι Ευρωπαίοι αγρότε παρήγαγαν, συνέχισαν να παραγάγουν ασφαλή τρόφιμα υπό δύσκολου όρου και αυτό το οφείλουμε στο ευρωπαϊκό γεωργικό μοντέλο. Οι μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, επιχειρήσει, επιχειρήσεις, οικολογικέ και συμβατικέ επιχειρήσεις εργάζονται υπό το πλαίσιο, υπό την αιγίδα τη κοινή γεωργική πολιτική. Στο μέλλον θα υπάρξει ένα μελλοντικό μοντέλο για την κοινή γεωργική πολιτική και θα αξιοποιήσει τη διαφάνεια όχι μόνο δηλαδή θα υπάρχει ανταμοιβή για την τηρήση των κανόνων. Κύριε Καγκελάρη, σας χρειαζόμαστε στο πλευρό μας να ενισχύσετε την αγορά, να αγωνιστείτε για μια ε, ισχυρή, ένα ισχυρό προπολογισμό για τα γεωργικά και αυτά χρειάζονται για τον παγκόσμιο ανταγωνισμό και για την νομική βεβαιότητα. Με μια ισχυρή γεωργία θα μπορέσουμε και στο μέλλον να τα στις μελλοντικές κρίσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σκοφόντ, Για ένα λεπτό. Σας ευχαριστούμε κυρία καγκελάριε, για την παρουσίαση των προτεραιοτήτων της Γερμανικής Προεδρίας. Οφείλω να σας εκφράσω την ανησυχία μου, τη σοβαρή μου ανησυχία με αυτά που μας αναγγείλατε. Είπατε ότι θα τα καταφέρουμε. Πάνω από ένα εκατομμύριο άνθρωποι ε, ήρθαν στην Ευρώπη από την Αφρική και τη Μέση Ανατολή. Η πολιτική, ε, μεταναστευτική πολιτική, η πολιτική για το άσυλο δεν είναι η σωστή. Έχουμε τεράστιες και ανεξέλεγκτες μεταναστευτικές ροές. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τις κοινωνίες μας, όχι να κλειστούμε στον εαυτό μας, αλλά να τις προστατεύσουμε. Επίσης δεν θα πρέπει η Ευρώπη να γίνει εστία Ισλαμισμού. Ε, και εστία Ισλαμιστών που θέλουν να υπονομεύσουν και να υποσκάψουν την ειρήνη και τη δημοκρατία μας. Μέχρι στιγμής ε, η πολιτική σας ε, δεν είχε επιτυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τις ζημίες που ήδη αναγγέλλονται από την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό το λόγο έχει ο κύριος Κνασροτέμψκι. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Καγκελάρια κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η ύφεση λόγω της πανδημίας μπορεί να οξύνει τις οικονομικές ανισορροπίες και διαφορές στην Ευρώπη. Ε, πολύ, πολύ ε, φοβόμαστε ότι οι ισχυρότερε και πιο εύφορες χώρες θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο και πιο αδύναμες θα έρθουν σε ακόμη μειονεκτικότερη θέση. Ε, επίσης, ε, δεν μπορούμε την Επρασίνη Συμφωνία να την εφαρμόσουμε σε καιρό ύφεση. Είναι προφανές ότι κάποιες α, χώρες λόγω ιστορικής γεωγραφικής κατάστασης δεν μπορούν να υλοποιήσουν χωρίς τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα τους α, περιβαλλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Ταμείο Δίκης Μετάβασης ίσως αυρύνει κάπως τις επιπτώσεις, αλλά δεν μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα. Από τη Γερμανική Προεδρία περιμένουμε ρεαλιστική εξέταση των περιβαλλοντικών πόρων και μια ρεαλιστική στρατηγική για την υλοποίηση αυτών των περιβαλλοντικών στόχων. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο για ένα λεπτό έχει ο κύριος Χαλίτσκι, αξιότιμη κυρία Καγκελάρια. Ε, στο μέλλον θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τεράστιες προκλήσεις ε, την οικονομία, το σχέδιο ανάκαμψη, τα δισεκατομμύρια που θα μα βοηθήσουν να εξέλθουμε από την κρίση. Μερικοί μιλούν για δεύτερο σχέδιο Marshall για την ευρωπαϊκή μα κοινότητα αλλά θα πρέπει να έχουμε υπόψη και τη δημοκρατία. Θέλουμε ένα σχέδιο Marshall και για την ανοικοδόμηση της δημοκρατίας και την προάσπιση των θεμελιωδών μας αξιών, που είναι η βάση της ε, κοινότητάς μας και μία από τις βασικές αξίες είναι η αλληλεγγύη, γιατί η αλληλεγγύη είναι το εχέγγυο της ασφάλειας. Ε, το γνωρίζουμε στην Πολωνία το σύνθημα της αλληλεγγύης. Χωρίς αλληλεγγύη δεν νοείται ελευθερία και αλληλεγγύη απέναντι σε όλους. Και μερικοί δεν ε, καταλαβαίνουν, δεν αντιλαμβάνονται τη διάσταση αυτή τη λέξη τη αλληλεγγύη. Από την κρίση αυτή η Ευρώπη θα πρέπει να εξέλθει ισχυρότερη και πιο αλληλέγγυη. Ο, κύριο Αντρίου για ένα λεπτό, παρακαλώ. Κυρία Καγκελάριε, η Γερμανική Προεδρία έχει τεράστιες ευθύνες να υπομειστεί. Περισσότερο από ποτέ η Ευρώπη θα πρέπει να είναι εδώ για να ε, βοηθάει τους ε, πολίτες και τα κράτη στην Ένωση και να τους είναι χρήσιμη και σήμερα και αύριο. Για το λόγο αυτό οφείλεται να επιτύχετε στην πρώτη φάση της Πράσινης Συμφωνίας με ουσιαστική ε, μεταρρύθμιση της κοινή γεωργικής πολιτικής που θα πρέπει να συνάδει με τις ε, τεράστιες αλλαγές κλιματικές, κοινωνικές, οικονομικές. Η τεράστια αλλαγή θα είναι και δημοσιονομική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται ίδιους πόρους για να χρηματοδοτήσει το σχέδιο ανάκαμψη και επιπλέον και το ε, πολιετές δημοσιονομικό της πλαίσιο. Μάλιστα, θα χρειαστεί φόρος επί των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ε, στα κέρδη των πολυεθνικών και ιδιαίτερα των ψηφιακών εταιριών και ένα συντορισμένο φόρος ε, στους πολυεκατομμυριούχους και στους δισεκατομμυριούχους στην Ευρώπη. Να πάψει αυτή η φορολογική κούρσα και ο ανταγωνισμός και για τα κλιματικά. Και τέλος θα πρέπει να συνδέεται ε, το κράτος δικαίου οικονομική ενίσχυση και να καταπολεμήσουμε την φοροαπάτη ε, και φοροδιαφυγή. Δεν έχουμε χρόνο για να αποτύχουμε. Θα πρέπει να είμαστε στο πλευρό σας για να ε, πετύχουμε σε αυτό το στίχημα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γκάρι Κάνο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Φόντερ Λάιεν και κυρία Μέρκελ που ήρθατε. Κυρία Μέρκελ, καταλαβαίνω ότι ε, θα είναι τεράστιο επίτευγμα και μεγάλη ανακούφιση η Συμφωνία για την Ανάκαμψη, το μεγάλο πακέτο. Κανείς δεν το περίμενε αυτό να το δει, αλλά λυπάμαι ένα τέτοιο επίτευγμα δεν ε, είναι αρκετό. Όπως είπατε επανειλημμένα, χρειαζόμαστε ένα σχέδιο αποπληρωμής. Έχουμε ένα σχέδιο για να αποπληρώνουμε τα χρέη μας. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να αναβάλουμε για 7 χρόνια ε, το, το, τη λύση. 505 μέλη του Κοινοβουλίου μας ε, έχουν την πρόταση για τους ιδίους πόρους που θα εξασφαλίσει το οικονομικό μέλος της Ευρώπης. Το σύστημα θα είναι πολιτικά βιώσιμο γιατί οι μεγάλοι ρηπαίνοντες και μεγάλες εταιρείες ε, θα πρέπει να βάλουν το χέρι στη τσέπη. Κάντε το αυτό στόχο της Προεδρίας σας, να έχει ένα σύστημα ιδίων πόρων η Ευρωπαϊκή Ένωση με γερά οικονομικά και ευημερούσες οικονομίες. Μην το αφήσετε αυτό για άλλα 7 χρόνια. Ευχαριστώ κυρία Μπιτσότο για ένα λεπτό. Καλώ ήρθατε, καγκελάρια Μέρκελ. Θεωρείστε ηγέτη τη Ευρώπη. χτίζεται όμως μια Ευρώπη με τα συμφέροντα της Γερμανίας. Το είδαμε αυτό την περίοδο της λιτότητας. Η Ιταλία θέλετε να μπει κάτω από τη... το πόδι των Βρυξελών. Ποιος σας δίνει όμως ε, τη δύναμη να αμφισβητείτε και να καταπατάτε την Ιταλική ανεξαρτησία. Δεν θέλουμε τέτοιες εξουσίες από τη Βρυξέλλα. Οι Ιταλοί θέλουν τα χρήματά τους πίσω, τα πραγματικά τους χρήματα τα εκατοντάδες εκατομμύρια τα οποία έχει ε, δωρήσει η Ιταλία τα τελευταία χρόνια στην Βρυξέλλες. Θέλουμε να σώσουμε τη ζωή ε, εκατομμυρίων ε, ανθρώπων και επιχειρήσεων. Θέλουν απλά δουλειά. Να σας υπενθυμίσουμε ότι η Ιταλία καθορίζεται από τους Ιταλούς πολίτες, όχι από τους Γερμανούς. Η επικυριαρχία μας, η κυριαρχία μας λοιπόν δεν είναι προς πώληση, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Η κυρία, ε, ο κ. κυρία Καγκελάρια, πολλοί θεωρούν ότι αυτό είναι το πολιτικό σας σκληροδότημα. Υπάρχει η κλιματική καμπή. Έχω την εντύπωση ότι έχετε εγκαταλείψει σε ό,τι αφορά την ε, σε ό,τι αφορά την, ε, το Ταμείο Ανάκαμψη, μιλάμε για μεγάλο ποσά. Πώ όμω θα δαπανηθούν αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια, δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική. Ο κ. Βίσκο από τι Ιταλικέ Τράπεζε είπε ότι η Ιταλία δεν χρειάζεται χρήματα, χρειάζεται μεταρρυθμίσει. Χρειάζεται λοιπόν εξοικονόμηση. Η φτώχεια στην Γερμανία και στην Ολλανδία παράλληλα αυξάνεται. Εσείς αλλάζετε την νομισματική ένωση και τη μετατρέπετε σε μια ένωση μεταφορών. Αυτό θα είναι το κληροδότημά σας, ένα βουνό χρεών. Και δυστυχώς η Γερμανία ακολουθεί τέτοιους ηθικισμούς. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα πρέπει να χάσουμε. Να, δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε την πραγματικότητα και να επιδεινώσουμε την περαιτέρω την κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ραγιζέλη για ένα λεπτό. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καγκελάρια Μέρκελ, αφήστε να σας πω ως Ευρωπαίος, ως ε, εκπρόσωπος Ευρωπαίων, ως Πορτογάλος, ως μέλος του ΕΛΚ και ως μέλος του ΠΕΣΔ. αφήστε με να σας διαβεβαιώσω ότι έχετε την υποστήριξή μας και τη δέσμευσή μας υπέρα της Ευρωπαϊκής Δέσμευσης και Προσήλωσης που μας αναφέρατε. Θέσατε δύο ξεκάθαρες ερωτήσεις που συνδέονται με την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Μιλήσαμε πολύ για κράτος δικαίου και δημοκρατία στα κράτη-μέλη, αλλά θέλουμε δημοκρατία και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Καταρχήν, για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα ευρωομόλογα που χρειαζόμαστε που ε, απ' την άλλη θα μας φέρουν και τεράστιες δαπάνες ευρωπαϊκές. Γι' αυτό θα πρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία έγκρισης αυτού του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, θα πρέπει να έχει ευρία συμμετοχή, θα πρέπει να έχει μεσοπρόθεσμο προσανατολισμό. Και επίσης ε, να είμαστε ανοιχτοί αν αποφασιστεί ε, να είμαστε ε, ανοιχτοί και για μεταρρύθμιση των συνθήκων προκειμένου να ενισχύσουμε την δημοκρατική νομοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πύρη για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κύρια Καγκελάρια Μέρκελ. Ε, στη διάρκεια πολλών κρίσεων δείξατε ότι είστε πραγματική ευρωπαϊκή ηγέτης. Και τώρα οι προσδοκίες των πολιτών είναι υψηλέ. Θα πρέπει να προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις ε, σε δυσχερείς οικονομικούς και κοινωνικούς καιρούς και συνθήκες. Πέραν της ε, οικονομικής αλληλεγγύης όμως θα πρέπει να είμαστε δίκαιοι και απέναντι στις θεμελιώδεις μας αξίες και η δική μου οικογένεια μεγάλωσε πίσω από το σίδερο παραπέτασμα και συμφωνώ με την πεποίθησή σας ε, μιας ε, ενωμένη και δημοκρατικής Ευρώπης. Ξέρουμε πώς είναι να ζει κανεί σε δικτατορικό καθεστώς. Κυρία Μέρκελ, δείξτε θάρρο στην προάσπιση του κράτου δικαίου. Υψώστε στεντόρια τη φωνή σα απέναντι στον Όρμπαν ή σε όσου υποσκάπτουν τα θεμέλια των ελεύθερων κοινωνιών μα. Και δράστε αποφασιστικά και με πυγμή την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Να δείξετε αποφασιστικότητα υπέρ τη αιρεσιμότητα με το κράτο δικαίου στον επόμενο επταετή προπολογισμό. Αν δεν σταθείτε στην προάσπιση των θεμελιωδών αξιών, θα πληρώσουμε ένα τίμημα που πραγματικά θα είναι δυσβάσταχτο για την Ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χαράντζοβα, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κύριε Καγκελάρια όποτε αντιμετωπίσαμε παγκόσμιες προκλήσεις είτε με τον Πούτιν είτε με τον Ερδογάν ήσασταν ο άνθρωπος που πήρε το προβάδισμα και με ηγετικό ρόλο ένωσε την Ευρώπη. Αυτό όμω που θα κρατήσω από την ηγετική σα θέση είναι η ικανότητά σα να βρείτε ε, ρεαλιστικέ λύσει σε πραγματικά προβλήματα και να καταφέρατε να μετατρέψετε τα έργα τα λόγια συγγνώμη σε έργα τις λέξεις σε πράξεις. Και αυτή τη δεξιότητά σας ε, και την αποτελεσματικότητά σας τη χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ στην Ευρώπη για το μακρυπρόθεσμο προϋπολογισμό μας, για την ανάκαμψη της οικονομίας μας. Μα ζητήσατε να διαδραματίσουμε μεσολαβητικό ρόλο. Θα ήθελα και εγώ να ζητήσω από εσά να παίξετε το ρόλο ενός έντιμου διαμεσολαβητή εδώ στην Ευρώπη. Σας ζητώ να εργαστείτε όχι μόνο ε, για μια γαλλογερμανική λύση, αλλά για μια λύση που θα ε, εξυπηρετεί το Βορρά και το Νότο, την Ανατολή και τη Δύση, το Βερολίνο, το Παρίσι, αλλά και την Πράγα. Και θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμβαστική λύση που θα μας ενώνει. Πιστεύω ότι αυτή την ισορροπία μπορεί να τη βρει η Γερμανία και να είναι η φωνή όχι μόνο της Γερμανίας, αλλά της ευρωπαϊκής συνένεσης. Κάτι τέτοιο χρειαζόμαστε περισσότερο από ποτέ. Η κυρία Μπάρλι για ένα λεπτό. Αξιότιμη ε, κυρία ε, Καγκελάρη, Υπουργέ, ε, σας καλωσορίζω στις Βρυξέλλες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μεγάλες οι προσδοκίες, αλλά βλέπω ότι είναι θωρακισμένη η Προεδρία. Και πραγματικά με την Γερμανική πρωτοβουλία δείξατε ότι θέλετε να δράσετε ευρωπαϊκά. Μιλήσατε για πάθος. Για μένα το μεγάλο μου πάθος είναι το κράτος δικαίου. Και Προς μεγάλη μου χαρά αναφερθήκατε ήδη από την αρχή στα θεμελιώδη δικαιώματα. Τώρα απευθύνω έκκληση τα λόγια αυτά να γίνουν και έργα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι δημοκρατία, κράτος δικαίου, εξάρτητη δικαιοσύνη, ελεύθερο τύπο σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε ένα μηχανισμό κυρώσεων αποτελεσματικό. Γι' αυτό πραγματικά θέλω να εμείνω. Ε, μην αφήσετε να σας κάψουν εκείνοι που θέλουν να αλλάξουν, ε, να παρακάψουν την πλειοψηφία των δύο τρίτων. Μην υποκύψετε, γιατί ακριβώς το θέμα δεν είναι να συμμορφωθούν οι συγκεκριμένες κυβερνήσεις, αλλά να καταλάβουν οι πολίτες ότι είμαστε με την πλευρά της δημοκρατίας. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Τσε κυρία ε, Μέρκελ, ε, στην Ουγγαρία είναι κρίσιμα τα πράγματα. Πριν από ένα μήνα ε, και κάτι, ένα μέλος της αντιπολίτευσης συνελήφθη από την αστυνομία γιατί στο Facebook είχε επικρίνει τον Όρμπαν. Επίσης, με το μεγαλύτερο ιδιαισιογραφικό site αγωνίζεται να επιβιώσει. διαφθορά οργιάζει και η κρατική ευθερεσία. Δέκα χρόνια ε, κυβερνάει ο Όρμπαν και δέκα χρόνια εσείς ολιγορείτε. Γιατί μας λέτε ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Όχι. Θα πρέπει να πηγαίνουν τα ευρωπαϊκά κονδύλια στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις ΜΚΟ, στους ανθρώπους που τα χρειάζεται. Και όχι σε μία ε, διεφθαρμένη κυβέρνηση που ε, τα υπεξαιρεί και τα καταχράται. Δεν μπορείτε αυτό να το υποστηρίξετε. Η αδράνεια είναι και αυτή η επιλογή. Είναι μια επιλογή ολέθρια στην ε, σταθερότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι ακόμα ένα καρφί στο φέρετρο της ε, Ουγγρικής Δημοκρατίας. Για ένα λεπτό, η κυρία Φρίτσον, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Καγκελάριε. Χαίρομαι για το φιλόδοξο πρόγραμμα της Γερμανικής Προεδρίας. Το σύνθημά σας είναι καλό. Πραγματικά θα πρέπει να επιδείξουμε ενότητα, αλληλεγγύη, αποφασιστικότητα. Χρειαζόμαστε φιλοδοξία, ρεαλισμό και ευθύνη ε, στο πρόγραμμα ανάκαμψης. Επίσης, θα πρέπει να προετοιμαστούμε για μια νέα οικονομία πράσινη, μεταρρυθμισμένη, όπου τα κοινωνικά δικαιώματα και η ελευθερία να είναι τα γερά θεμέλια. Ε, θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια, ε, την παιδική, ε, την ανεργία. Καταλαβαίνετε ότι τα μικρά παιδιά όταν ζουν στη φτώχεια πλήττονται περισσότερο. Οι γυναίκες επίσης θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ε, σε όλα τα όργανα διοίκησης στην Ευρώπη ε, ε, και η ανάπτυξη να είναι πιο δίκαιη και πιο ελεύθερη. Αυτό το οφείλουμε στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Ευχαριστώ για ένα λεπτό η κυρία Βάουτμανς. Αγαπητή Καγκελάρη, δεν είμαι σίγουρη αν επιτρέπετε ακόμα να το πούμε στην εποχή του Me αλλά ε, είστε πραγματικά από τους λίγους πολιτικούς που έχετε τα κότσια και καταλαβαίνετε τι εννοώ για να πάρετε αποφάσεις και να δράτε. Ε, καταφέρετε ε, να έχετε ηθικό ανάστημα κατά τη διάρκεια της κρίσης, ακόμα και αν ήταν απέναντί σας η κοινή σας γνώμη ο ίδιος σας ο υπουργό Οικονομικών. Και πραγματικά, ε, στη δική σας ηγεσία υπολογίζουμε για να ηγηθείτε στην Ευρώπη. Με τη γαλλογερμανική πρόταση και την πρόταση της Κομισιόν πραγματικά είναι το σωστό. Πιέστε να περάσει. Και τέλος θα ήθελα να σας καλέσω να πάρετε άλλη μια σημαντική απόφαση. Νέα στρατηγική με την Κίνα. θα πρέπει να μπει στην ημερήσια διάταξη η συμπεριφορά τη Κίνα και η πάταξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Χονγκ Κονγκ. Θα πρέπει να τολμήσετε να αντιμετωπίσετε την Κίνα. Καλή τύχη και μπορείτε να υπολογίζετε σε εμά, θα είμαστε στο πλευρό σα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπούλμαν. Για λεπτό έχει το λόγο. Κυρία Καγκελαρία. Η συζήτηση καταδεικνύει πόσο μεγαλε είναι οι ελπίδε οι οποίε βαρύνουν, αν θέλετε, την ε, Γερμανική Προεδρία και θεωρώ ότι είναι σωστό γιατί έχουν γίνει τα σωστά βήματα. Και οι πρώτε ενδείξει των τελευταίων εβδομάδων και μηνών ε, είναι λεπιδοφόρε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από εκείνο τα πράγματα. Οι σοσιαλδημοκράτε στη Γερμανία πάντα ζητούσαν να υπάρχει αλληλεγγύη, αλληλεγγύη και ανανέωση. Και καταφέραμε να αλλάξουμε πολλά παλιά πράγματα. Σπάσαμε ταμπού και μάλιστα αναχρονιστικές τέτοιες ε, πρακτικές. Αυτό είναι καλό, αλλά θα πρέπει να υπάρξει οικολογική και κοινωνική ανανέωση, γιατί χρειαζόμαστε μια ισχυρή Ευρώπη στον κόσμο, γιατί τα δείγματα των καιρών τα βλέπουμε στη Νέα Υόρκη. Ο, ο κόσμος ε, συγκλονίζεται από τον COVID-19. Μόνο αν ανοικοδομήσουμε λοιπόν την Ευρώπη σε αυτό το προοδευτικό πνεύμα θα καταφέρουμε να συμβάλλουμε αυτά που μας αναλογούν. Και τέλος, αυτή η συζήτηση για το κράτος δικαίου Μιλώντα με τους σκανδιναβούς φίλους μας, θα δούμε πόσο μεγάλε είναι οι αμφιβολίες για τις ε, καταχρήσεις του κυρίου Ορμπάν. Δεν θέλουν οι ολιγάρχες να επικρατήσουν. Θα πρέπει να δώσουμε λοιπόν τα χρήματα στους δημάρχους ε, στις μικρές επιχειρήσεις που ξέρουν τι θα κάνουν τα χρήματα αυτά, τα κονδύλια αυτά και θα τα χρησιμοποιήσουν στο έπακρο. Ευχαριστώ κυρία Κέλλη για ένα λεπτό. Κυρία Καγιαλάρια, στις 15 Μαΐου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με μεγάλη πλειοψηφία ενέκρινε ένα ισχυρό ψήφισμα για το σχέδιο ανάκαμψης. Στις 18 Μαΐου εγκαινιάσατε μια πρωτοβουλία μαζί με τον πρόεδρο Μακρόν που στη συνέχεια εστερνίστηκε και η πρόεδρος Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Κυρία Καγκελάρια, η ταχύτητα εφαρμογή αυτού του σχεδίου ανάκαμψη θα έχει αποφασιστική σημασία. Πώς ε, θα εξασφαλίσετε μέσα σε 10 μέρες ε, ισχυρή συμφωνία στο Συμβούλιο για να ε, ενισχύσουμε ήδη από αύριο τις επιχειρήσεις και τους πολίτες να ορθοποδήσουν μετά την κρίση. Ε, θέλουμε χρηματοδότηση με ιδίους πόρους όπως πρότεινα κάποια συνάδελφοι. Επίσης, στα θέματα της μεταναστευτικής κρίσης, είστε έτοιμοι να ταχθείτε υπέρ μιας πολιτικής συμφωνίας για το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο. Κυρία Καγκελάρη, αγαπητή Άγγελα Μέρκελ, καλή επιτυχία στην Προεδρία σας, στα γερμανικά, κυρία Κελέρ. Σα Σας ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Σεφτσοβιτς έχει τώρα το λόγο εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητή Καγκελάρια Μέρκελ, αξιότιμη Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά για την πραγματικά δυναμική και ζωηρή ευρωπαϊκή συζήτηση και ευχαριστώ την Καγκελάριο για την γνήσια ευρωπαϊκή ηγεσία που δείχνει. Και νομίζω ότι Είμαστε σε μια πρόκληση της ευρωπαϊκής ιστορίας και η αποφασιστικότητα υπέρ τη χαλογερμανικής πρόταξης δίνει ευκαιρία και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σας ε, υποβάλει μια πρωτοφανή πρόταση αναζητώντας τρόπους για να συνδυάσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το επόμενο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με το σχέδιο ανάκαμψης, στο Next Generation EU. Δεν πρόκειται να επισέλθω σε λεπτομέρειες γιατί η συζήτηση θα αποκολουθήσει, θα επικεντρωθεί στο σημείο αυτό και θα έχουμε ε, την συζήτηση παρουσία και του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του κυρίου Μισελ. Οπότε εγώ θα ακολουθήσω μια άλλη κατεύθυνση ε, για άλλα σημεία που θα χαρακτηρίσουν την Γερμανική Προεδρία. Χαίρομαι που ταχθήκατε υπέρ των ευρωπαϊκών αξιών, τονίσατε τη σημασία της αλληλεγγύης και είπατε πόσο σημαντικά είναι τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μερικές φορές ξεχνάμε στις ε, σφοδρές συζητήσεις που έχουμε και στο Συμβούλιο, ξεχνάμε ότι η συνοχή είναι η βιώσιμη επένδυση στο μέλλον και ένα επιτυχημένο σχέδιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση που την καθιστά πιο ισχυρή και πιο αθεκτική στο μέλλον. Και νομίζω ότι αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε. Και νομίζω το διαπιστώσατε και από τη συζήτηση, κυρία Μέρκελ, ότι θα πρέπει να καταπολεμήσουμε τον επικίνδυνο λαϊκισμό, την, το μίσος, τη ρητορική του μίσους και να προασπίσουμε το κράτος δικαίου θέματα προσφυλή για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ε, περάσαμε σε ένα... Είχαμε την εμπειρία ενό καθεστώτο που δώσαμε μάχη την Ευρώπη και τώρα χαιρόμαστε για την ε, επιτυχία που είχαμε και μπορούμε να ταξιδεύουμε ελεύθερα στην Ευρώπη. Για μας είναι πολύ διαφορετικό όταν μιλούμε για τη σημασία τη δημοκρατία και τι ευαισθησίε ε, απέναντι στις θεμελιώδεις ελευθερία και πόσο σημαντικό είναι να επανέλθουμε στο σύστημα Σέγγεν το σύντομότερο δυνατό γιατί είδαμε πώ είναι να μην έχουμε αυτή την ευκαιρία τη ελεύθερη διακίνηση. Όλοι ελπίζουμε και είμαστε αισιόδοξοι για την επόμενη εβδομάδα ότι θα καταλήξουμε σε μια ιστορική συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανική πάντως Προεδρία θα συμπέσει με μια ε, κρίσιμη στιγμή της ευρωπαϊκής συζήτησης και ιστορίας. Και αν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταλήξει σε συμφωνία, τότε θα ξεκινήσει το πραγματικό έργο. Και σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ξεκινήσουμε ε, ένα πολύ δυναμικό και έντονο εξάμεινο νομοθετικών πρωτοβουλειών με φρενήριες ρυθμούς για να δώσουμε πραγματικά ε, νέα παλμό στην ευρωπαϊκή οικονομία να ανακάμψει, να γίνει ανθεκτικότερη, να περάσει το ψηφιακό ε, μετασχηματισμό, να γίνει πιο περιβαλλοντική και οι σωρευτές οι μπαταρίες κύριε Ερτούγκ είναι από τις προτεραιότητές μας. Σας ευχαριστώ θερμά για την πολύ σημαντική συζήτηση που είχαμε και ευχαριστώ και την καγκελάριο Μέρκελ για το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα για το επόμενο εξάμεινο της Γερμανικής Προεδρίας που χρειάστηκε να το προσαρμόσει στις συνέπειες της κρίσης COVID. Πάντως ελπίζω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα καταλήξουμε σε σημαντικότατες, βαρισίμαντες συμφωνίες που θα ανοίξουν ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ιστορία και ένα νέο κεφάλαιο στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο ε, ο λόγος στην κυρία Μέρκελ για να απαντήσει. Παρακαλώ, κυρία Καγκελάρη. Σύντομα, για να κλείσουμε, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές και σε αυτό το δεύτερο γύρο αποκρισταλώθηκε και πάλι ε, το θέμα της δράσης για το κράτος δικαίου. Το κάνουμε ως Γερμανία και κατονομάζουμε τα ζητήματα και τα θέτουμε υπόψη των συναδέλφων. Ακόμα και είναι ο Βίκτορ Όρμπαν και διαφωνούμε για τα τεκτενόμενα στην Ουγγαρία. Και αυτό είναι πραγματικά θεμητό συμφέρον απολύτως και του Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να ε, καταλήγουν τα κονδύλια στους ε, νόμιμους δικαιούχους και πραγματικά επαγρυπνούμε και φροντίζουμε γι' αυτό. Θέλω να καθησυχάσω και εκείνου που λένε να μην κάνουμε μόνο ε, γαλλογερμανικές προτάσεις. Γνωρίζουμε ότι η Ευρώπη αποτελείται από 27 κράτη-μέλη, αλλά όταν διαφωνούν πολύ η Γαλλία με τη Γερμανία δεν προάγονται τα ευρωπαϊκά ζητήματα. Βεβαίως ε, μπορούμε να κάνουμε και το άλλο ε, αλλά φυσικά δεν εννοείται ότι η γαλλογερμανική πρόταση μόνο είναι ευρωπαϊκή. Ε, θα το κάνουμε τις επόμενες εβδομάδες. Χαίρομαι που αναφερθήκατε εδώ στο θέμα της ε, γεωργίας. Αν το κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά, ε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις. Βλέπε μόνο τον πυλώνα 1 και τον πυλώνα 2 της ε, γεωργικής πολιτικής. Αν θέλουμε όμως να είμαστε μια οικολογική ήπειρος, πρέπει να έχουμε και οικολογική παραγωγή τροφίμων και παραγωγή τροφίμων καν στην Ευρώπη ε, θα πρέπει ε, να δεχόμαστε τους αγρότες, να τους αναγνωρίζουμε στη δουλειά τους, αλλά να τους θέτουμε υπόψη ότι χρειάζεται βιώσιμη διαχείριση των εδαφών, ευημερία των ζώων και στην κτηνοτροφία. Ε, όλα αυτά όμως θα πρέπει να συνοδεύονται από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για τη σωστή λειτουργία. Χαίρομαι επίσης που μιλήσατε για την τεχνολογία και έπαιξε ρόλο αυτό το θέμα. Ε, μπορούμε προσωπικά, προσωρινά μάλλον, να δανειζόμαστε, αλλά θα πρέπει να αποπληρωθούν αυτά. Ε, ε, πότε θα γίνει αυτό στην επόμενη προγραμματική περίοδο ή ε, μήπως στην ερχόμενη ε, να αρχίσει η αποπληρωμή. Γιατί το θεωρώ σημαντικό, γιατί ε, ο δανεισμός στο δίνεκες δεν μπορεί να είναι η απάντηση της Ευρώπης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και στην κούρσα. Από τη μια θα πρέπει να ποντάρουμε στις νέες ε, τεχνολογίες και ελπίζω αυτό να φανεί και στο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί. Αν έχουμε από τη μια τα διορθωτικά ταμεία και από την άλλη τις δαπάνες για την καινοτομία, αλλά και εκεί η Γερμανία ε, θα αφιερώσει αρκετά κονδύλια, θα ζητήσει να αφιερωθούν στην τεχνολογία. Ε, και χαιρετίζω το γεγονό ότι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πήρε απόφαση για τη στρατηγική για το υδρογόνο. Έχουμε αντίστοιχη και στη Γερμανία και υπάρχουν και άλλα κράτη που το έχουν. Είναι στρατηγικό το συμφέρον μα πέρα από την παραγωγή των μπαταριών που ε, έχει ξεκινήσει καλά αυτό το θέμα και στην εκβαντική τεχνολογία θα πρέπει να αναλάβουμε δράση. Και θέλω να πω σε εκείνους ε, που ε, λένε ε, αν θα πρέπει να ανανεώνουμε την Ευρώπη φυσικά καθημερινά ο κόσμος αλλάζει και αν παραμείνουμε στάσιμοι θα μείνουμε πίσω προφανώς και η Γερμανία επικρίνεται και σωστά επικρίνεται ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στο μέλλον. Θα πρέπει όλοι να καταβάλουμε την προσπάθεια να γίνουμε καλύτεροι και να χρησιμοποιήσουμε εκεί την ανάκαμψη. Ε, σας ευχαριστώ που αντέξατε μέχρι ε, τέλους αυτή τη συζήτηση και εύχομαι καλή συνεργασία το επόμενο εξάμεινο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την πρόεδρο, την πρόεδρο Μέρκελ, την Γελάριο Μέρκελ και τώρα θα διακόψουμε για ένα λεπτό και μετά θα ξεκινήσουμε με το επόμενο θέμα στην ημερησία διάταξη. E Αγαπητοί συνάδελφοι, επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Ε, πριν συνεχίσουμε, σας ενημερώνω ότι στις 4.30 θα αρχίσει ο πρώτος γύρος των ψηφοφοριών. Ε, ε, είπαμε και στην αρχή της συνεδρίασης. Άρα αυτός ο γύρος ε, ψηφοφορίας θα ε, τελειώσει στις 6 παρατέταρτο. 16 και 30 με 17 και 45 θα διαρκέσει. για τα διάφορα θέματα που σας ανέφερα, για το ελεγκτικό συνέδριο, για την Χέλγα Μάγιο για την ε, τραπεζική αρχή. Όλα αυτά θα γίνουν με μυστική ψηφοφορία οι βουλευτές μπορούν να ψηφίσουν κανονικά, αλλά ε, ε, το ψηφοδέλτιο που θα υπογράψουν ε, θα αναφέρει μόνο ότι ψήφισαν, όχι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οι άλλες ψηφοφορίες θα είναι μυστικές, ε, ονομαστικές, συγγνώμη. Και η επεξηγήσεις ψήφου ε, κατ' εξαίρεση θα φτάνουν τις 400 λέξεις. Στις 8 θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα. Σύμφωνα με την μέρη σε διάταξη ακολουθεί κοινή συζήτηση ε, για τη συνεδριάση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19 η Ιουνίου και 17 και 18 Ιουλίου 2020. Ε, Καλωσορίσατε κύριε Μισελ a cui do subito la parola per il suo intervento introduttivo. Prego, Presidente. Κύριε Πρόεδρε, έκλεισε το μικρόφωνο του μιλητή. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καταρχάς, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που έχουμε ε, να συζητήσουμε. Η COVID-19 έδειξε ότι δεν μπορεί κανείς πάντα να ελέγχει όσα του συμβαίνουν. Αυτό που μπορούμε όμως να ελέγχουμε είναι η απόκρισή μας. Ας μην λησμονούμε ότι η πανδημία είναι ακόμα εδώ αυτή τη στιγμή που μιλούμε συνεχίζεται ε, και καταστρέφει ε, ζωές, επιχειρήσεις και ε, θέσεις εργασίας. Μία και μόνη στατιστική δείχνει πόσο δραματική είναι η εικόνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να χάσει 1,5 δισεκατομμύρια το 2020-2021 και μόνο. Είναι πραγματικά πολύ ζωφερή αυτή η προοπτική. Όπως γνωρίζετε, στις 23 Απριλίου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έρθει με ένα σχέδιο ανάκαμψης και τον Ιούνιο οι ηγέτες είχαν την πρώτη συζήτησή τους για την πρόταση ευρωπαϊκή Επιτροπής. Θα σας πω περισσότερα σε λίγο. Κάποια στοιχεία της ε, πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ακόμα απαράδεκτα ε, για κάποια κράτη-μέλη. Για το λόγο αυτό, μετά τη συνεδρίαση μας, ε, αρχίσαμε τις διμερείς επαφές ε, με ε, όλους τους ηγέτες και στις 17 και 18 Ιουλίου έχω συγκαλέσει την πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου με αυτοπρόσωπη παρουσία. Υπάρχουν κάποια ζητήματα που θέλω να τονίσω. Το πρώτο είναι η ενημέρωση που σας κάνω, η τακτική, η παραδοσιακή για το τι έγινε τον Ιούνιο και το δεύτερο είναι να σας πω τι έγινε στις διμερείς μου επαφές και να μοιραστώ μαζί σας τις προθέσεις μου για το ερχόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Και τέλος θα ήθελα να απευθύνω ισχυρή έκκληση για φιλόδοξη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και με εσά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να δράσουμε από κοινού αν θέλουμε να λειτουργήσει σωστά το σύστημα. 19 Ιουνίου η τελευταία ε, βιντεοδιάσκεψη ήταν η πρώτη φορά όπου συζήτησαν οι ηγέτες τις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ε, πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο και το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό ήταν σημαντικό βήμα για να προετοιμαστούμε για ε, τις αποφάσεις που θα πάρουμε σε, βάση με, τη, σχέση με τη σημερινή φάση διαπραγματεύσεων. Ποιοι ήταν οι τομείς όπου ε, υπάρχει η συνένεση ή διαφαίνεται. Πρώτον, συμφώνησαν τα κράτη-μέλη ότι θα πρέπει από κοινού να αντιμετωπίσουμε το θέμα του PDP και το Ταμείου Ανάκαμψης. Επίσης, στο δεύτερο, συμφώνησαν ότι ε, η κρίση αυτή άνευ προηγουμένου, ε, προηγουμένου χρειάζεται άνευ προηγουμένου απάντηση και επίσης θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε ε, τομείς και περιφέρειες που έχουν πληγεί περισσότερο. Αλλά επίσης παρατηρήσαμε και τομείς όπου οι απόψεις μας χρειάζεται ακόμα να συγκλίνουν. Για παράδειγμα, η ιδέα ε, ε, του δανεισμού για τις επιχορηγήσεις είναι πολύ δύσκολο να γίνει δεκτή από κάποιους ηγέτες και τα κριτήρια ε, που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατανομή τους. Γιατί θεωρούν ότι δεν συνδέεται η παρούσα πρόταση με την κρίση COVID-19 και τις συνέπειές της. Την περασμένη εβδομάδα ε, ολοκλήρωσα τον πρώτο γύρο διμερών επαφών που είχα. Ήταν εντατικές και καμιά φορά και δύσκολες, ίσως ε, και πολύ δύσκολες, αλλά πάντα σε επικοδομητικό πνεύμα. αυτό μου επέτρεψε να δω ποια είναι τα έξι κεφάλαια της μελλοντική συμφωνίας που νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε τη σωστή πολιτική ισορροπία. Πρώτον, το μέγεθος του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ξέρετε ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για το μέγεθος που είναι αποδεκτό και το δεύτερο που συνδέεται με το πρώτο είναι το ζήτημα ε, των διορθώσεων των επιστροφών, rebates, ε, που για κάποια κράτη-μέλη είναι πολύ σημαντικά, ενώ για κάποια άλλα πρέπει να καταργηθεί. Αυτό θα είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν ε, σε μια συνολική ενδεχόμενη συμφωνία. Επόμενο θέμα, το επίπεδο του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι πρότεινε. Όλα τα κράτη-μέλη δεν συμφωνούν με την άποψη αυτή ότι θα πρέπει να γίνει δεκτό ε, το ποσό. Επόμενο θέμα είναι η, ε, τα δάνεια και οι επιχορηγήσεις και η ίδια η ε, έννοια των επιχορηγήσεων που δεν θα αποπληρώνονται προβληματίζει κάποια κράτη-μέλη και επίσης η αναλογία των δύο μεταξύ του. Και το πέμπτο σημείο ε, θα ήθελα λίγο να σταθώ εδώ, είναι τα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων στα πλαίσια ε, ε, του Ταμείου. Πολλά κράτη-μέλη τον Ιούνιο εξέφρασαν δισταγμούς και επιφυλάξεις. Η πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε στοιχεία πριν ξεσπάσει η πανδημία. Δηλαδή ήταν το, το επίπεδο ανεργίας και το αντίστροφο ΑΕΠ και ο πληθυσμός. Δεν είναι αρκετά δυναμικά αυτά τα κριτήρια, ούτε προσφέρονται, θεωρούν κάποια κράτη, για να λάβουν υπόψη την πραγματική κατάσταση σε περίπτωση οικονομικού και κοινωνικού αντικτύπου ε, για τις χώρες που πλήττονται περισσότερο. Για το λόγο αυτό εξετάζουμε την ιδέα ε, να φέρουμε μια πιο δυναμική προσέγγιση στα κριτήρια κατανομής των κονδυλίων. Το έκτο, πολύ σημαντικό, είναι η σχέση ε, των μεταρρυθμίσεων και της διακυβέρνησης και των διαφόρων θεσμών με όλα αυτά. Ε, αυτό αφορά άμεσα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και ε, σε σύνδεση λοιπόν με το Ταμείο Ανάκαμψης υπάρχει το κράτος δικαίου που θα πρέπει να συζητηθεί και το ζήτημα της κλιματικής διάστασης. Πολύ σημαντικό επίσης. Θυμάστε ότι πριν από λίγους μήνες, πριν αρχίσει η κρίση, προτείναμε ένα σημαντικό κεφάλαιο του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου να συνδέεται με τις κλιματικές φιλοδοξίες. Και θυμάστε ότι το Δεκέμβριο ήταν πολύ μεγάλες φιλοδοξίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο να φτάσουμε στην ουδετερότητα για το κλίμα το 2050. also other. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία διακυβεύονται. Και ξέρω ότι είναι κρίσιμα για σας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καταρχάς, το θέμα των ιδιών πόρων και αντιλαμβάνουμε ότι αυτό είναι η κλειδί για τη συμφωνία σας. Ε, πολλά έχουμε ακούσει για τα πλαστικά απορρίμματα, για το ETS, το σύστημα εμπορία ρήπων και υπάρχουν διάφορες δισταγμοί. Αλλά εξετάσαμε και άλλες, ε, άλλους πόρους ε, που έχουν υποστηριχθεί ψηφιακός φόρος, φόρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών, η ευελιξία για το πολιτικό δημοσιονομικό πλαίσιο σε ό,τι αφορά και την γεωργία αποτελούν σημαντικά θέματα για κάποια Και έχουμε και άλλα δύο θέματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε συμφωνία. Καταρχά, ε, το θέμα του front-loading στο Ταμείο Ανάκαμψη ε, και το θέμα των δεσμεύσεων και των πληρωμών και τη χρονική στιγμή και το θέμα της, ε, του πότε θα ξεπληρωθούν τα χρήματα αυτά. Ξέρουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τώρα αυτό να γίνει όχι στη διάρκεια του τρέχοντος ε, πολίτε δημοσιονομικού πλαισίου, αλλά στο επόμενο, στην επόμενη περίοδο. Ίσως θα υπήρχε, θα ήταν σκόπιμο να προταθεί να ξεκινήσει πιο νωρί. Τα επόμενα βήματα, όπω θα ξέρετε, ανακοίνωσα ότι σκοπεύω να δημοσιεύσω ένα πραγματευτικό κοιτίο μέχρι το τέλο τη εβδομάδα. Με τη Γερμανική Πρόεδρε θα συζητήσουμε όλα αυτά, στην Κορεπέρ με όλους τους πρέσβες. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να προετοιμάσει τη σύνοδο του Ιουλίου. Να σας διαβεβαιώσω ότι κάνω ότι περνάει από το χέρι μου για να πετύχουμε συμφωνία. Θα πρέπει να βρούμε μια σωστή λύση. Έχω την εντύπωση μετά από το γύρο αυτών διαβολέψεων που ήταν πάρα πολύ δετικός τις τελευταίες ε, ημέρες και τελευταίες εβδομάδες ότι δεν είμαστε ακόμα στο τέλο των διαπραγματεύσεων, δεν έχουμε ολοκληρώσει τι διαπραγματεύσει. Ε, είναι τεράστιο ογκός της εργασίας που επιμένει να γίνει. Έχουμε ωστόσο προχωρήσει. Υπό τον όρο αφενός ότι τα κράτη-μέλη θα δείξουν διάθεση να συνεργαστούν ε, περαιτέρω και θεωρώ ότι αυτό θα είναι απαραίτητο για την, αποτελεσμα... για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης και υπό τον όρο ότι θα αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων για την κινητοποίηση των πόρων αυτών και θα πρέπει όλοι να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και το Κοινοβούλιο σε συνεργασία με την ε, Προεδρία προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε αποτελέσματα και είμαι Επίση, πεπισμένο ότι θα τα καταφέρουμε αν ο καθένα όλοι αποδεχτούν να προσεγγίσουν αλληλού. Αν κάθε κράτος και αν κάθε θεσμικό όργανο παραμείνει τελματωμένο και περιχαρακωμένο στις θέσεις τους δεν θα βρεθούμε λύση και δεν θα μπορέσουμε να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων γιατί πιστεύω ότι αυτή είναι η μοναδική λύση να κάνουμε ένα βήμα προς αλλήλους για να υπάρξει φιλοδοξία, αλλά και μια ρελιστική υπεποίθηση. Για να μπορέσουμε να πάρουμε από κοινού απαντήσει. Αυτή την έκκληση θέλω να απευθύνω προ όλου σα. Και όλα αυτά είναι θεμελιώδη σημασία γιατί θέλουμε έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό για τα επόμενα 7 χρόνια και ένα ταμείο ανάκαμψη. Είναι τεράστιο λοιπόν το έργο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα έχει τρει στόχου. Ότι δεν ε, μπορούμε να περιμένουμε, θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα. Καταρχά, ο στόχο να ακολουθήσουμε τη σύγκληση. Αυτό ήταν από αρχή ο στόχο μα. Να συνεχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε προ ε, την κατεύθυνση αυτή τη σύγκληση τη ευρωπαϊκή. Ε, άκοπα επίσης να εργαστούμε για την ανθεκτικότητα. Αυτό το χρειαζόμαστε σε ιστορικό επίπεδο για να μπορέσουμε να διδαχθούμε από τα παθήματα της κρίσης ε, και να μπορέσουμε να έχουμε δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε. Και τρίτος στόχος ε, τον οποίο θα επιδιώξουμε θεωρώ είναι να έχουμε υπόψη μας την μεταμόρφωση, τη μεταμόρφωση του ευρωπαϊκού οράματος σε ψηφιακό επίπεδο και να χρησιμοποιήσουμε αυτή την κρίση ως μια ευκαιρία για να δώσουμε ένα έναυσμα να αγωνιστούμε προς την κατεύθυνση αυτή και μάλιστα με αξιόπιστο και αισιόδοξο τρόπο. Είναι δύσκολη αυτή η στόχη και είναι και μεγάλο το διακύβευμα, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αλλά είμαι πολύ αποφασισμένος να προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά με τέτοια ταχύτητα που να μπορούν να ακολουθήσουν όλοι. Με διάλογο επικοδομητικό, θετικό με τα θεσμικά όργανα και προφανώ και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα. Σα ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μισελ. Τώρα το λόγο έχει ο κύριος Σεύκοβιτς, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, όπως συζητήσαμε και νωρίτερα. Μια μεγάλη κρίση βιώνει η Ευρώπη όχι μόνο η Ευρώπη βέβαια, αλλά και ολόκληρος ο κόσμος ε, πενθεί. Πραγματικά η COVID-19 έχει τεράστιο οικονομικό και ανθρώπινο κόστος, ε, αλλά ε, επιφέρει και αλλαγές και φαντάζομαι θα συμφωνήσετε μαζί μας προς το ότι δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω σε ό,τι ίσχυε προ-COVID-19. Δεν υπάρχει επιστροφή προς τα πίσω, άρα πρέπει να κοιτάξουμε το μέλλον. Και αν δρούμε αποφασιστικά μπορούμε να βρίσκουμε λύσεις. Το ίδιο πρέπει να γίνει και σε αυτή την περίπτωση. Ξέρετε, πολλέ φορέ λέω ότι εδώ χτυπάει η καρδιά τη Ευρωπαϊκή Δημοκρατία, το Ευρωκοινοβούλιο. Εδώ συζητούνται οι πολιτικέ, εδώ χαράσσονται οι πολιτικέ. Όμω ε, δεν αρκεί να συζητούμε για τι πολιτικέ προτεραιότητε. Πρέπει να έχουμε και τα απαραίτητα κονδύλια να τι εφαρμόσουμε στην πράξη. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εν ώψη αυτή τη συνόδου θα ήθελα να σα αναφέρω δύο πολύ σημαντικά για μα ζητήματα και για το μέλλον μα. Πρώτα απ' όλα το καθεστώ σε σχέση με το σχέδιο ανάκαμψη ε, Next Generation EU και το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Έχουν κατατεθεί προτάσει. Θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την πολύ επικοδομητική, ε, προνοητική θα έλεγα, προσέγγιση που ακολούθησε και τι έντονε διμερεί επαφέ που είχε με του αρχικού κρατών και κυβερνήσεων. Και επίση για τη στενή συνεργασία του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλα αυτά είναι απαραίτητα και αναγκαία, διότι πρόκειται για ένα πολύ φιλόδοξο πακέτο, το οποίο ανταποκρίνεται με άμεσο και αποφασιστικό τρόπο στι ανάγκε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το προσεχέ π ενισχύεται ε, με αυτό το εργαλείο για την αντόση της κρίσης, το Next Generation EU. Σχεδόν 2-3 εκατομμύρια ευρώ είναι η δύναμη πυρός ε, από οικονομικής πλευράς. Η ε, εντυπωσιακά βέβαια τα ποσά. Άρα αναγκαία και σίγουρα πρέπει να ανταποκριθούμε στην κρίση. Πρόκειται για κάτι άνευ προηγουμένου στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό το σχέδιο στόχο έχει όχι μόνο να ε, περάσουμε τα πρώτα χρόνια προ την ανάκαμψη, αλλά γιατί θέλουμε να έχουμε και ε, ενίσχυση των προτεραιοτήτων ε, μέχρι το 2027 και επέκεινα και να μπορέσουμε να τις υλοποιήσουμε. Και θέλω να ε, παναλάβω. πόσο ζωτικό είναι ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτή τη διαδικασία. Αργότερα σήμερα η πρόεδρο Φοντερ Λάιν μαζί με τον πρόεδρο Μισελ, την καγκελάριο Μέρκελ και τον πρόεδρο Σασόλη θα συναντηθούν δυνάμει του άρθρου 324 οπότε και θα ξεκινήσει χάρη στους ηγέτες η πρώτη απόπερα σύγκλησης απόψεων ώστε να έχουμε πρόσφορο έδαφος για την επίτευξη συμβιβασμού της 17ης και 18ης ε, Ιουλίου στη Σύνοδο Κορυφής. Ήταν ενθαρρυντικές οι συνομιλίες των γητών σε μια πρόσφατη βιντεοδιάσκεψή τους και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρούμε ότι υπάρχει ε, θετική δυναμική για την υποστήριξη των προτάσεων που μόλις ε, περιγράψαμε. Και Ειδικότερα υπάρχει μια συμφωνία ως προς ε, ε, την έκτακτη αντιμετώπιση για αυτή την έκτακτη κρίση και η χρηματοδότηση θα γίνει με δανεισμό από πλευράς ε, κομισιών. Υπάρχει επίσης συμφωνία σε ό,τι αφορά την αύξηση του ανώτατου ορίου, της οροφής των ιδιών πόρων. Θεωρούμε επίσης ότι υπάρχει συμφωνία προς το ότι οι προσπάθειές μας θα πρέπει να είναι στοχευμένες προς τις πλέον πληγήσεις περιοχές Ένωσης για ενίσχυση της συνοχής και της σύγκλησης η κρίση αυτή και η αντίδραση στην κρίση θα δημιουργήσουν μοναδικές ε, ευκαιρίες για να κάνουμε πιο πράσινες, πιο ψηφιακές και ανθεκτικές τις οικονομίες μας. Η προτινόμενη δέσμη μέτρων αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό τι ε, προσδοκίε του Κοινοβουλίου από το ψήφισμα τη 15η Μαου και ειδικότερα θέλω να σα ευχαριστήσω για τη συνεχή υποστήριξή σα ε, προ ε, του νέου ιδίου πόρου. Όπω και εσεί, έτσι και εμεί είμαστε πεπισμένοι πω αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. Με του νέου ίδιου πόρου μπορούμε να προωθήσουμε του κοινού μα στόχου, να αναπληρώσουμε ότι θα δανειστούμε μέσω του Next Generation EU, αλλά χωρί να δημιουργήσουμε κίνδυνο για το μέλλον των προγραμμάτων και θα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες ελπίζοντας ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία και θα έχουμε κάποιες προτάσεις επιτάπτως για να κάνουμε αυτό το ποιοτικό άλμα, το γιγαντιαίο άλμα ε, για το μέλλον και ιδίως ε, ξεκινώντας από τον χρόνο θα θέλουμε να έχουμε έναν οδικό χάρτη για να πετύχουμε ε, τη μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδίων πόρων. Και βασίζομαι σε εσά να περάσετε το μήνυμα και στις πατρίδες σας, στις κυβερνήσεις των χωρών σας, ε, στις περιφέρειές σας, στα εθνικά κοινοβούλια, να τους εξηγήσετε πόσο πολύ χρειαζόμαστε την υποστήριξή τους, διότι ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία και χρειάζεται ηγετική στάση από εμάς πάνω απ' όλα. Λίγες εβδομάδες μόλις μας απομένουν, διότι όλοι γνωρίζουμε πως είναι απολύτως αναγκαίο να αντιδράσουμε στην κρίση και άρα να πετύχουμε συμφωνία πριν τις θερινές διακοπές. Αυτό βέβαια εφόσον θέλουμε πριν τα τέλη του έτους να έχουμε ολοκληρώσει και τη διαδικασία εθνικής ε, κύρωσης ε, των αποφάσεων για τους ιδίους πόρους διότι αλλιώ δεν μπορούμε ε, χωρί αυτή την απόφαση να ξεκινήσουμε ούτε το δανεισμό, αλλά εάν μάλιστα τα εθνικά κοινοβούλια δεν εγκρίνουν ε, τη συζήτηση, τα αποτελέσματα και τα νέα αυτά μέσα και εργαλεία, δεν θα υπάρχει και δημοκρατική νομοποίηση των ε, προτάσεων αυτών. Παναλαμβάνω, είναι άνευ προηγουμένου ε, και τεράστια κλίμακα ε, και χρειάζεται αυτή η δημοκρατική νομοποίηση. Πρέπει επίση να υπογραμμίσω το γεγονό ότι με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέα εργαλεία όχι μόνο για τη βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη, αλλά και για να δείξουμε ξεκάθαρα ότι οι δημοκρατικοί κανόνες είναι αυτοί που πάντα θα υπερέχουν, ακόμη και εν καιρό κρίσης. Άκρος επικοδομητική προσέγγιση λοιπόν είναι κάτι που απαιτείται από όλα τα θεσμικά όργανα και νομίζω ότι πρέπει να ακούσουμε ένα τον άλλο και να προσπαθήσουμε κάπως να συμφιλιώσουμε τις διαφορετικές μας απόψεις στην όλη αυτή διαδικασία. Δεύτερον, η συμμετοχή του Κοινοβουλίου σε όλες αυτές τις πτυχές είναι θεμελιώδης σημασία. Ο το κάθε ευρώ που θα δαπανηθεί θα πρέπει να φέρει τη σφραγή του Κοινοβουλίου. Συναποφασίζεται, ελέγχεται μέσω της διαδικασίας απαλλαγής, ε, ασκείτε τον κοινοβουλευτικό σας έλεγχο Έχουμε αυτό το έκτακτο σύστημα που απαιτείται για την έκτακτη αυτή κρίση. Όμως το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρέπει επίσης να διαδραματίσουν σε πλήρη βαθμό το ρόλο που τους αναλογεί. Εμείς είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί σας και με το Συμβούλιο σε ό,τι αφορά μια θεσμική διακήρυξη. Για να ξεκινήσουμε λοιπόν να δώσουμε το επίσημο αναρτήριο λάκτισμα και να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη δυνατή συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Αξιότιμοι βουλευτέ, κυρίε και κύριοι, όπω σα είπα, ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο, όμω αν έχουμε το σωστό μείγμα ρεαλισμού, ηγεσία, φιλοδοξία, νομίζω ότι μπορούμε να τα αποκριθούμε στι προσδοκίε των Ευρωπαίων πολιτών. Θα χρειαστεί τη βοήθειά σα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να είμαστε ταχεί σε όλε τι φάσει τη διαδικασία, σε ό,τι αφορά παραδείγματο τη συμφωνία για να ξεκινήσει το σχέδιο ανάκαμψη ε, στο, και στο πλαίσιο του ΠΔΕΛΤΑΠ. Όσο το όσο το συντομότερο ε, ξεκινήσουμε και με το ReactEU και με το SURE, τόσο το καλύτερο. Το δεύτερο που έχω να πω σήμερα ε, είναι σε σχέση με το Brexit. Όπως γνωρίζετε, ο συνάδελφος Μισελ Μπαρνί είναι στο Λονδίνο σήμερα. Εκεί λαμβάνει χώρα ένας ακόμη γύρος διαπραγματεύσεων και νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό. Έξι μήνε μόλι μα χωρίζουν από το τέλο τη μεταβατική περίοδου. Αποκινούμε το Ενωμένο Βασίλειο προσφάτω. Κάναμε τον απολογισμό των ε, διαπραγματεύσεων που είναι σε εξέλιξη και τονίσαμε ότι εμεί είμαστε πρόθυμοι να καταβάλουμε κάθε πιθανή και δυνατή προσπάθεια που θα οδηγήσει σε ένα συμβιβασμό ε, και στην υπογραφή μια μοναδική εταιρική ε, σχέση, μοναδική στο είδο τη. από τότε όμω μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει πρόοδο και η απλή αλήθεια είναι ότι ε, Ούτω ή άλλω, με τον έτομο τρόπο, σε λίγου μήνε αυτέ οι διαπραγματεύσει θα ολοκληρωθούν. Αν θέλουμε να ολοκληρωθούμε μια συμφωνία, θα πρέπει να γεφυρώσουμε τι αποκλήσει που μα χωρίζουν σε μια σειρά από ζητήματα, όπω για παράδειγμα ε, τι εγγυήσει, ε, τι ασφάλειε, ε, η μια ισορροπημένη συμφωνία για την αλληλεία, ένα πλαίσιο διακυβέρνηση ε, κτλ. Τα ξέρετε πολύ καλά, ε, είμαι βέβαιο, αυτά τα ζητήματα. Ξέρετε πόσο σημαντικά είναι και για εμά, γιατί έχουμε και τι αρχέ του δικαίου ανταγωνισμού, την ανάγκη προστασία των πολιτών πολιτών. Αρχές ε, που είναι στο κέντρο, στην καρδιά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ε, και πιστεύω ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί συμφωνία. Θα κάνουμε πάντο δυνατό. Ο χρόνος και εδώ είναι λίγος. Δεν ξέρουμε πού θα έχουμε φτάσει μέχρι τα τέλη του χρόνου. Και αν βέβαια καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία, εξακολουθεί να είναι πολλά αυτά που θα αλλάξουν στις μελλοντικέ μας σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, για του πολίτε, για τις επιχειρήσεις, για τι εθνικέ διοικήσει. Και πρέπει να προγραμματίσουμε για αυτέ τι αλλαγέ, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τι εθνικέ αρχέ και άλλου ε, εμπλεκομένου φορεί ε, στην προετοιμασία του. Και με τι διαπραγματεύσει αυτή και τόνισε προ του ηγέτε η κυρία Φοντελάιν, μαζί με τι διαπραγματεύσει πρέπει να συνεχίσουμε το έργο μα ε, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρη εφαρμογή τη συμφωνία αποχώρηση, που είναι και προϋπόθεση για την διατήρηση τη εμπιστοσύνη Έχουμε την ε, μεικτή αυτή επιτροπή, είμαι μέλος της και παραμένουμε πάρα πολύ προσεκτικοί και παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις όλες τις πτυχές των συζητήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διδραματίσει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και σε αυτήν ε, την διαπραγμάτευση και σας είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων ε, για την υποστήριξή σας ε, όπως και αυτή φαίνεται στη, στο ψήφισμα στις 18 Ιουνίου. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι, κύριε Μισελ, σας ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στη διάθεσή σας για να σας υποστηρίξουμε στις προσπάθειές σας τον επόμενο εβδομάδα και μηνών ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεύκοβιτς, Πρόεδρε Σεύκοβιτς και τώρα θα ακούσουμε τις πολιτικές ομάδες. Ο Πρόεδρος Μισελ ζήτησε να πάρει πάρει και πάλι το λόγο στο τέλος αυτού του πρώτου γύρου ώστε να ακούσουμε τους εκπροσώπους των ομάδων. Ο κύριος Μούρης, αναξενόματος του Λαϊκού ε, Κόμματος. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε Μισελ, καλώς ορίσατε στο Ευρωκοινοβούλιο. Σα ακούμε, σα ε, ανησυχούμε, ε, ανησυχούμε μάλλον και δεν συμφωνούμε μαζί σα γιατί ακριβώ δεν εμπλέκεται το Κοινοβούλιο στι συνομιλίε περί προπολογισμού όπως τα οφείλατε διότι πρόκειται για το δεύτερο σκέλος ε, αρμόδιο για τον προπολογισμό και θέλουμε έναν προπολογισμό που να μπορούμε να κάνουμε περισσότερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα με, με μικρότερο προπολογισμό. Δεν είναι μαγικό φασό που μεγαλώνει μόνο όταν το κοιτάμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να δώσει τη συγκατάθεσή του στο ΔΕΛΤΑΠ όταν αυτό συμφωνεί και χρηματοδοτεί τα όσα έχουμε μαζί συμφωνήσει. Έχουμε συμφωνήσει την γεωργία και τη συνοχή καταρχάς ως προτεραιότητες και αυτές πρέπει να χρηματοδοτηθούν καταρχάς. Έπειτα νέες προτεραιότητες, ψηφιοποίηση, πρασίνισμα, προστασία περιβάλλοντος, έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, εξωτερικά σύνορα, μετανάστευση, δεν μπορούμε να λύσουμε τη λύση του κορονοϊού δημιουργώντας προβλήματα σε άλλους τομείς μέσω της υποχρηματοδότησης. Τα, εμείς πρέπει να σας δώσουμε το μήνυμα αυτό. Δεν μπορούμε να κρύψουμε ένα μικρότερο ε, πι δέλτα πι πίσω από το πακέτο ανάκαμψης. Για το πακέτο ανάκαμψης τα χρήματα θα πρέπει να δαπανηθούν για τον εξυγχρονισμό της Ευρώπης και για τα σύνορα με προστιθέμενη αξία. Έπειτα, όσο περισσότερα χρήματα δαπανηθούν, τόσο καλύτερο έλεγχος πρέπει να γίνεται. Και έπειτα, Κάθε πολίτης, κάθε εταιρεία όταν παίρνει μια πίστοση πρέπει να, δώσει, να την αποπληρώσει, πρέπει να δει πώς και πότε θα μπορέσει να αποπληρώσει και το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε και εμείς ως Ένωση. Ήδη οι πόροι, και ε, θα πρέπει πριν το 2027 να το έχουμε αποφασίσει αυτό και να δώσουμε δεσμευτικό ε, χρονοδιάγραμμα για τους υπόλοιπους ίδιους πόρους. Μόνο έτσι θα μπορέσει το Ευρωκοινοβούλιο να δώσει κατάθεση στο τέλος. Και οποιαδήποτε συμβιβαστική μπορεί να βρείτε στο Συμβούλιο, είμαστε έτοιμοι να σας μιλήσουμε, να διαπραγματευτούμε μαζί σας γιατί η συμφωνία αυτή δεν θα είναι η τελική. Οι απόψεις του Κοινοβουλίου πρέπει να ληφθούν υπόψη και να συμπεριληφθούν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Μουρεσάν, η πρόεδρος των Σοσιαλιστών, η κυρία Γκαρσία Πέρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πανδημία ε, πήρε τη ζωή πάνω από 100.000 ε, ε, Ευρωπαίων συμπολιτών μας. Χωρίς θυσίες όμως δεν μπορεί να οικοδομηθεί αυτό το Ευρωπαϊκό ευρωπαϊκό όραμα. Πολλές γυναίκες από τις ε, υγειονομικές ε, υπηρεσίες θυσιάστηκαν για να μπορέσουν να μας προστατεύσουν. Έχουμε τεράστιες συνέπειες από, ε, από τα περιοριστικά μέτρα και έχουμε και μια κοινωνική τραγωδία γιατί ο ιός έχει, έχει χαντακώσει τις, προθε... τις ελπίδες εκατομμυρίων νέων Ευρωπαίων. Πολλές γενιές έχουν σχηματίσει, έχουν σφυριλατήσει τις... Ε, το χαρακτήρα τους από δραματικές, ε, δραματικά γεγονότα, ε, για... από γεγονότα που αλλάζουν τη ζωή και ο κόσμος πρέπει να αναλάβει κινδύνους. Όμως ο χρόνος καθορίζει τη ζωή. Εδώ και μήνες η πανδημία σοβεί και ο Ιούλιος θα πρέπει να είναι ο μήνα του, του πακέτου ανάκαμψη και του προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι επόμενε γενιέ πρέπει να αισθανθούν πω η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα χώρο οικονομική ασφάλεια για τη ζωή του. Και χάρη στην ισχύ αυτού του Κοινοβουλίου και αυτέ τι διαπραγματεύσει, είμαι πεπισμένη ότι αυτό θα το καταφέρουμε. Οι σοσιαλδημοκράτε δεν θα δεχθούμε λιγότερο από 500 εκατομμύρια ευρώ σε ε, επιδοτήσει από πλευρά Κομισιόν. Δεν θα δεχτούμε καμιά ε, επίση ρεσιμότητα μακροοικονομική, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά καλά τι θα πει λιτότητα. Ε, ε, ε, χειρότερες συνθήκες για τους εργαζόμενους και περικοπές στις κοινωνικές δαπάνες. Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στις πολιτικές λιτότητας και όσον αφορά τη βοήθεια η στήριξη θα εξαρτηθεί από την αυστηρή τήρηση του κράτους δικαίου και τη χρήση που θα ε, γίνει αυτών των κονδυλίων. Οι νέοι είναι αυτοί που επηρεάζονται περισσότερο από τον ιό και από τις ε, οικονομικές ε, συνθήκες. Η πανδημία δεν μπορεί να αποτελέσει δικαιολογία για να αντιμετωπιστεί η ανισότητα μέσω του κοινωνικού πυλώνα με εγγύησεις για τα ε, παιδιά και την ασφάλεια. Κανένα στην κοινωνία μας δεν μπορεί να αισθανθεί σίγουρος χωρίς να έχει δουλειά πρέπει να φροντίσουμε τη, μετα... τη μεταμόρφωση της οικονομίας μας για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις ε, κλιματικές προκλήσεις και την ψηφιακή πρόκληση και για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ε, μεταρρυθμίσεις χωρίς να στραγγαλίσουμε τους προπολογισμού των κρατών μελών θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε τους ίδιους πόρους. Είναι θεμελιώδης αυτή η συζήτηση για μας. Εάν οι λιγότερο ευνοημένες τάξεις ε, υπέφεραν από την προηγούμενη κρίση, τώρα πρέπει οι αγορές και οι πολυεθνικές να συμβάλλουν σε μια δίκαιη ανάκαμψη οι περικοπές των κοινωνικών παροχών οδηγούν στην απομόνωση, ε, στην, ριζοσπαστικοποίηση. Οι δικές μας πολιτικές πρέπει να συμβάλλουν στην επιτυχία αυτού του πλάνου. Κύριε Μισελ, θέλω να σας ζητήσω στις διαπραγματεύσει ε, τις επόμενες μέρες με τους πρωθυπουργούς να τους κοιτάξετε στα μάτια και να τους ρωτήσετε το εξή. Αν δεν μπορούμε να εγγυηθούμε στους πολίτες μας ότι η ζωή τους θα είναι καλύτερη, τότε τι κάνουμε εδώ πέρα. Πραγματικά αυτό το Ευρωκοινοβούλιο το γνωρίζει πάρα πολύ καλά και εργάζεται γι' αυτό και είμαι πεπισμένη ότι όλοι μαζί θα μπορέσουμε να υπερασπιστούμε ένα ισχυρό δίκαιο και αλληλέγγυο πρόγραμμα. Σας ευχαριστούμε Πρόεδρε Γκαρσία Πέρες και τώρα η κυρία Αγέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ε, Σασόλη. Κύριε Πρόεδρε Μισελ, το πρόγραμμα αυτό ανάκαμψη είναι πρωτοφανέ και θα πρέπει γι' αυτό να δώσει και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Θα πρέπει από το κύκλιο μα να αλλάξουμε την καθημερινότητα των Ευρωπαίων. Γι' αυτό 500 δι επιδοτήσεων είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την κοινωνική και οικονομική κατάρρευση. Και η πολιτική μα οικογένεια, Πρόεδρε, θα παρακολουθεί δύο κυρίω σημεία στενά. Πρώτα απ' όλα, αυτά που θα καθορίσουν το αν θα υποστηρίξουμε ή όχι τη συμφωνία. Δηλαδή, τους νέους ίδιους πόρους. Απαραίτητη για να αποπληρωθεί οποιοδήποτε χρέος. Δεν αρκεί η κλασική συνεισφορά. Το να υιοθετήσουμε μια κοινή προσέγγιση σε αυτό το θέμα δεν είναι κάτι απλό και δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει μόνο εδώ ε, στο δικό μας το σώμα. Αν και ξεπεράσαμε τους διχασμούς μας και το καταφέραμε. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε σε ανάκαμψη. Πρέπει αυτή τη στιγμή να γίνουν ε, κάποιο είδου δάνεια, αλλά χωρί να βαρύνουν τι μελλοντικέ γενιέ, προκειμένου να στηριχθούν τα κράτη. Και χωρί ε, να αφήσουμε ε, στο περιθώριο τι μεγάλε εταιρείε, που είναι και μεγάλοι ρηπαίνοντε, τι μεγάλε εταιρείε του ίντερνετ και να δούμε τι θα κάνουμε με την ε, πράξη, το πώς αυτά μπορούν να ε, γίνουν με έμπνευση τις συνθήκες μας για την οικονομική και κοινωνική σύγκληση. Δεν θέλουμε πλέον οι πλουτοκράτες, Κατσίνσκι, ε, Όρμπαν και άλλοι φίλοι τους να χρησιμοποιούν τους φόρους των Ευρωπαίων πολιτών για να ενισχύουν τις νεποτιστικές εταιρείε των χωρών τους και σε άλλες χώρες. Εδώ, Πρόεδρε, θα σας ευχηθώ κάθε τύχη στην θητεία σας, αλλά η πολιτική μας οικογένεια, ενωμένη εδώ το Κοινοβούλιο περιμένει να φτάσουμε στη συνοδό σα σε μια συμφωνία και να διαπραγματευτούμε προ όφελο των μελλοντικών γενεών τη Ευρώπη ένα μέλλον πράσινο και ευημερία. Ένα μέλλον δημοκρατικό. Ένα μέλλον ε, το οποίο θα βασίζεται στην αμοιβαία αναγνώριση. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Λεμπρετό για την ID. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Συμβούλιο συζήτησε στις 19 Ιουνίου το πρόγραμμα ανάκαμψης ε, της Ευρώπης και θα το ξανασυζητήσει 17 και 18 Ιουλίου με 550 δις ευρώ, ε, εκ των οποίων ε, τα 250 θα είναι δάνεια. Είμαι κατά του προγράμματος αυτού για δύο λόγους. Πρώτα απ' όλα γιατί θα υπάρχει η αμοιβαία χρέωση 500 εκατομμυρίων για όλη την Ευρώπη, κάτι που θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό ομοσπονδιακό κράτος που δεν θέλει η δική μου η ομάδα. Και θα πρέπει να είναι κανεί αφελή για να πιστεύει ότι θα δοθούν χωρί ανταλλάγματα αυτοί οι πόροι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει ε, δρακόντιου ε, όρου για να τα δεχτεί κυρίω για τι επενδύσει στην υγεία. Μόνο η Γαλλία και η Γερμανία φαίνεται να πρόκειται να πληρώσουν. Όμω η Γερμανία, εάν μπορεί να ε, επιτρέψει τον εαυτό τη μετά τη γενναιοδορία δεν μπορεί να το κάνει αυτό η Γαλλία που είναι δεχρεωμένη κατά το 120% του ΕΠ Ο πρόεδρο Μακρόν, που είναι από του εμπνευστέ του προγράμματο αυτού ανάκαμψη, άποψη, φαίνεται να έχει ξεχάσει ότι το πρώτο καθήκον ενό αρχηγού κράτου είναι να ασχοληθεί πρώτα με το δικό του το λαό. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Λάμπερτ για τους πράσινους. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Μισελ, πραγματικά έχω κάθε συμπάθεια για τη δική σας την κατάσταση εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε πετύχει πλειοψηφία. Θα πρέπει εσείς να πετύχετε ομοφωνία, κάτι κάπως διαφορετικό. Διότι αυτό που θα σας διχάσει ε, ίσως να είναι αυτό που θα καθορίσει για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Πραγματικά λοιπόν αισθάνομαι αλληλεγγύη και συμπάθεια για τη θέση σας. Από την άλλη, πραγματικά αναρωτιέμαι τι μπορείτε να τους πείτε. Διότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι πραγματικοί αντιρρησίες. Ε, και τι θα μπορείτε να ε, παρουσιάσετε. Ότι το ποσό φαίνεται τεράστιο. Εντάξει, αλλά τι λέμε, 1,5 του ΑΕΠ για τρία χρόνια. Ε, απέναντι σε μια ύφεση που θα σημαίνει το 9 ή 10% του ΑΕΠ εάν πραγματοποιηθεί. Ας δούμε τις επιπτώσεις της ΕΠΑ. Ε, μιλάμε για ποσά που ακούγονται μεν τεράστια, αλλά δεν είναι τόσο τεράστια. Θα δούμε λοιπόν τα πράγματα με κάποια απόσταση και σχετικά και πιστεύω ότι αυτό το πετύχετε. Το δεύτερο που θα μπορούσε να σα ε, προβάλλει κανεί ω διαφωνία είναι ότι το win-win δεν θα ισχύει. Ε, Μήπω τελικά χρεωθούμε ε, και τα δάνεια αυτά ε, δοθούν χωρίς ποτέ να αποπληρωθούν. Δηλαδή, μήπως θα είναι απλώς ε, δημοσιονομικά δώρα. Εδώ τίθεται το θέμα της αιρεσιμότητας. Ξέρω ότι είναι ένα θέμα που ακούγεται ως παγίδα, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Πιστεύω ότι η αιρεσιμότητα που θα πρέπει να επιβάλλουμε εδώ, οι αιρεσιμότητε στον κόσμο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, είναι η αιρεσιμότητα ως προς τη δημοκρατία και το κάτω δικαίου. Είναι η αιρεσιμότητα ως προς τις χρήσιμε, τι επωφελείς επενδύσεις. Και τι είναι πιο επωφελές σήμερα από τον επενδύσει κανεί βεβαίω σε χώρε που αντιμετωπίζουν δυσχέρειε, αλλά και σε εργαλεία τα οποία θα μπορέσουν πραγματικά να βελτιώσουν την οικονομία ολόκληρη τη Υπήρου. Πραγματικά οι επενδύσει στι οικολογικέ και αλληλέγγυε επενδύσει, οι ψηφιακέ τεχνολογικέ λύσει, ευθύ μεταφορέ. Αυτά είναι που πρέπει να κάνουμε. Διότι αν η λιτότητα πριν από μια δεκαετία ήταν η λύση για το κοινό μα προμένο, όχι, δεν θέλουμε το ίδιο. Οπότε θα πρέπει να μην βρεθούμε σε μια ε, εσφαλμένη λύση. Και το δεύτερο σημείο θα πρέπει κανεί να υπογραμμίσει και να το προβάλλει στου αντιρρησίε. Ε, τι θα κερδίσουν. Εάν το αποτέλεσμα ε, του να μην ληφθεί απόφαση υπέρ ενό ευρωπαϊκού προγράμματο ανάκαμψη θα είναι η κατάρρευση τη Ευρωζώνη, πού είναι το όφελο, ε, πού θα είναι η ευημερία για του Σκανδιναβού, πού θα είναι η ευημερία για του Αυστριακού ή του Ολλανδού, ε, όταν η νομισματική ένωση θα είναι μόνο ένα άθροισμα απολειών και κερδών. Ε, εδώ λοιπόν θα πρέπει την ευμάρειά μας, ε, την ατομική, εθνική δηλαδή, και εδώ διαφωνώ κάθετα με τον κύριο Λεμπρετό, να τη δούμε ως ευμάρεια του συνόλου. Δεν είναι το θέμα εάν θα δοθούν δάνεια χωρίς όρους, αλλά να κοιτάξουμε το ιστορικό αυτό σφάλμα, να διακινδυνεύσουμε το τέλος της νομισματικής ένωσης και της Ευρωπαϊκής κατ' επέκταση ένωσης για λόγους που θα έχουν μόνο εκλογικέ σκοπιμότητες από πίσω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε Φαν Όβερτφελ για το ECR. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε, Πρόεδρε, Επίτροπε, συνάδελφοι. Η οικονομική κρίση δεν έχει μόνο κάπως ταράξει τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των χωρών μας αυτό είναι πολύ ήπιο. Έχει πραγματικά ε, ταρακουνήσει, ε, είναι τσουνάμι ε, όσον αφορά την αβεβαιότητα Πρέπει όλα να τα βάλουμε όμως σε μια δυναμική προοπτική. Δεν γνωρίζουμε τι θα συμβεί. μπορεί να υπάρξουν νέα, νέα περιοριστικά μέτρα, να τόπους, θα υπάρξουν συνέπειες οι οποίες ακόμα είναι άγνωστες και είναι πολύ δύσκολο να εκτιμηθούν. Η δυναμική λοιπόν αυτής της κρίσης είναι πολύ σημαντική. Πρέπει να δούμε μακροπρόθεσμα τα πράγματα και αυτό ισχύει και για τις συνέπειες του Brexit. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να αυξηθεί η ε, αντίσταση, η ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας και των οικονομιών μας. Όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις για το πι είναι σαφές ότι το Κοινοβούλιο ήδη εδώ και καιρό ε, έχει λάβει θέση και έχει ανακοινώσει τους στόχους και τις επιθυμίες του. Υπάρχει μεγάλος βαθμός ομοφωνίας στην ε, ε, στο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και χρειάζεται όλοι οι φορεί Κομισιόν, Συμβούλιο και Κοινοβούλιο να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξει θεσμικό μπλοκάρισμα. Υπάρχει δυνατότητα, υπάρχει πιθανότητα, με συγχωρείτε, αλλά θα πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία. Εγώ μίλησα για τη σημασία της καταπολέμησης των αβεβαιοτήτων, αλλά αν υπάρξει τέτοιο μπλοκάρισμα διαθεσμικό, τότε η αβεβαιότητα ε, και η δυναμία θα, ανάκαμψης ε, θα είναι ακόμα πιο χαρακτηριστική. Ευχαριστώ πολύ. Ο Μπρι, εξ ονόματος της ε, Γκουε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τη στιγμή που συζητάμε σήμερα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο διαπραγματεύεται ε, κρυφά αυτό που παρα πλανητικά αποκαλείται Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης. Με, όμως ε, πίσω από αυτό το βαρύκδουπο όνομα πώς μπορούμε να μιλάμε για σχέδιο ανάκαμψης ενώ σε το μεγαλύτερο τμήμα αυτών των χρημάτων θα πρέπει να, να, να επιστραφεί. Η συζήτηση για την κατανομή ανάμεσα στα δάνεια και τις επιδοτήσεις δεν έχει τελειώσει και αυτό είναι θεωρητικό γιατί τελικά τα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να επιστρέψουν τα χρήματα και άρα η ευρωπαϊκή λαοί θα πληρώσουν την ύφη. Πώς τολμάτε να μιλάτε για σχέδια ανάκαμψη, ενώ πρόκειται για ένα ισχνό ε, σπρόξιμο 0,25%. Ε, ε, πώς τολμάτε να μιλάτε για σχέδια ανάκαψης όταν μόνο το 1 τέταρτο των κονδυλίων θα δοθεί μέχρι το 2023 και ε, τώρα χρειάζονται τα χρήματα τα ευρωπαϊκά κράτη η ευρωπαϊκή βοήθεια θα φτάσει κατόπιν εορτής παράλληλα ο ευρωπαϊκός προπολογισμός μάλλον θα μειωθεί και αυτό είναι ο κίνδυνος που περιμένουμε. Δηλαδή τι σημαίνει άντε μια από τα ίδια. Ε, πώς τολμάτε να μιλάτε για σχέδιο ανάκαψης χωρίς να έχει γίνει, να έχει οργανωθεί καμία δημοκρατική συζήτηση. Κα, ποιος μπορεί εδώ να εγγυηθεί ότι το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει, να πει, θα έχει λόγο ώστε να εξασφαλίσει πως αυτά τα χρήματα δεν θα δοθούν χωρίς οικολογικό και, οικονομικό και κοινωνικό αντιστάθμισμα. Ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό θα αποφύγει τη, ε, ε, τις κοινωνικές, ε, τα κοινωνικά κλεισίματα με σαν, όπως η Σανόφια, Ερμπάς και τα λοιπά ε, κλείνουν και κανείς δεν βοηθά τους εργαζόμενους. Η μόνη βεβαιότητα που έχουμε είναι ότι η Κομισιόν θα βγει από όλα αυτά ενισχυμένη και θα ενισχύσει και τη λιτότητα στα κράτη-μέλη. Διαπιστώνω επίσης ότι η κυρία Βαντελάιον όλο ένα και πιο ξεκάθαρη είναι ως πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για, για την επιστραφή από την πίσω πόρτα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και άρα του δημοσιονομικού ελέγχου και της λιτότητας. Το σχέδιο ανάκαμψης λοιπόν καμία σχέση δεν έχει με το όνομά του. Εάν υπάρξει ανάκαμψη είναι ανάκαμψη της φιλελεύθερης ε, ιδεολογίας σας. Πρόκειται για ένα τεράστιο σχέδιο επικοινωνιακό για να καταπιεί ο κόσμος το χάπι του φιλελευθερισμού. Και όμως μπορούσαμε να ακολουθήσουμε άλλο δρόμο, να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να απαντήσουν αμέσω στην κρίση, μέσω δανείων αμέσων ε, της ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα ε, και τη ακύρωσης του χρέους και έπειτα φτιάχνοντας ένα μεγάλο σχέδιο οικολογική ανασύστασης. Αυτό χρειαζόμαστε. Ένα σχέδιο ανοικοδόμησης ε, και στην πράξη εφαρμογής του, όχι σλόγγαν ε, και λόγια και ε, παραπλανητικά και σκηνοθεσίες από πλευράς του περίφημου γάλλο-γερμανικού ζευγαριού. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκιόν και από του εγγεγραμμένου. Ε, ευχαριστώ πολύ. Όλοι νιώθουμε ότι υπάρχει μια επίκουσα ανάγκη να εγκριθούν ε, στο επόμενο συμβούλιο τη επόμενη εβδομάδα ε, το Ταμείο Ανάκαμψη, το οποίο δεν τα πει για λόγου αλληλεγγύη. Όλοι μίλησαν για την αλληλεγγύη. Τον Απρίλιο όμω την ιδέα των ευρωμολόγων τη σκότωσαν στο Eurogroup και η μόνη πρόταση ήταν αυτή που θα μπορούσε να είχε μεταφέρει το χρέο από το επίπεδο των κρατών μελών στο ευρωπαϊκό επίπεδο αυτομάτω και έτσι να μεταφέρει το χρέο και και μαζί με αυτό να απορροφηθεί και το κόστος της ύφεση από τα κράτη-μέλη να πάει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ε, χρέος. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή αυτό το σχέδιο ανάκαψης δεν βλέπω πώς θα πάνε αυτά τα κονδύλια στους πλέον ευάλωτους απελπισμένους πολίτες, επιχειρήσεις, ε, μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις. Ούτε βλέπω τις εγγύησεις ότι αυτά τα κονδύλια ουσιαστικά δεν θα οδηγήσουν σε αύξηση του χρέους των κρατών μελών. Κάτι που τελικά θα οδηγήσει στη λιτότητα εκ νέου και στη την αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Πραγματικά με αποτροπιάζει αυτή η ιδέα της ε, διανομής των κονδυλίων από τις κυβερνήσεις ε, που ουσιαστικά ε, τα έχουν πλακάκια με τις πολυεθνικές, τους μεγάλους ομίλους ή με την εγχώρια ολιγαρχία. Πώς μπορούμε να περιμένουμε ποτέ τέτοιες συνθήκες να ε, πάνε στους πλέον ενδεείς αυτά τα κονδύλια. Γι' αυτό λοιπόν ε, σε αυτή τη συμφωνία θα πρέπει να περιληφθούν και αυτές οι εγγύησεις προτού εγκριθεί το Ταμείο Ανάκαψης και το ΠΔΕΛΤΑΠΗ. Ευχαριστώ. Πρώτα θα δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον κύριο Μισελ, για να δευτερολογήσει. Παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σα ευχαριστώ πολύ για τι παρεμβάσει και για τα μηνύματα. Ε, δεν κατάλαβα ακριβώς ε, τι είπε ο κύριος Μούρεσαν, ε, γιατί εγώ νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Κομισιών και Κοινοβουλίου είναι κάτι ανευπροηγουμένου και θα συνεχίσουμε να κινητοποιούμε ώστε όχι μόνο στο τυπικό επίσημο στην Ολομέλεια σήμερα για παράδειγμα, αλλά και στο πιο ανεπίσημο επίπεδο να έχουμε στενό μόνιμο διάλογο και εμείς από πλευράς μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και είπαμε ότι υπάρχει αυτή η διάθεση, υπάρχει ευρηματικότητα, υπάρχει. Υπάρχουν φάνταστες προτάσεις. Δεν θέλω να επαναλάβω κάθε ώρα και κάθε μέρα και με ε, απειλητικό τρόπο ότι πρέπει να είμαστε στο ραντεβού ε, εκεί και ότι πρέπει να σηκώσουμε τα μάτια και να στρωθούμε στη δουλειά. Ε, πώς να τα πω πιο ξεκάθαρα. Θέλουμε μια στεναρή, σταθερή Ευρώπη και το έχουν δείξει τα πράγματα ε, και θα πρέπει να μην αυταπατώμεθα πλέον. Δεν θα βοηθήσει η εθνική επαναχώρηση, η ομφαλοσκόπηση. Ε, κάνουν λάθος όσοι πιστεύουν ότι κάτι τέτοιο μπορεί να πετύχει. Χρειαζόμαστε στεναρή Ευρώπη, στέρη Ευρώπη απέναντι στις προκλήσεις. Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που μπορεί να φέρει το λάβαρο τη δάδα αυτή τη φιλοδοξία. Με τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας και είναι και σαφή τα, τα όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Ξέρουμε ότι έχουμε το ψηφιακό θεματολόγιο και ε, την ψηφιακή, την ψηφιακή της αντιπράσινη συμφωνία κτλ. Ε, θέλουμε να αντιλήσουμε τα διδάγματα, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη όμως και το τι ε, επέφερε η πανδημία της COVID-19 και Έχουμε αυτά τα κονδύλια, τα έκτακτα. Ε, όλα αυτά ε, θα πρέπει να σημάνουν ε, ένα μετασχηματισμό, μια μεταμόρφωση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και ίσω στο σχέδιο του Ευρωπαϊκού Οικονομικού να είμαστε σε ένα μετέχνιο. Γι' αυτό είναι τόσο πολύ δύσκολη από πολιτική πλευρά αυτή η συζήτηση, γιατί υπήρχαν, τα είπε κυρία υπήρχαν διαφορετικέ απόψει σε ό,τι αφορά του ίδιου πόρου, για παράδειγμα. Και βλέπω και εντό των διαφορετικών ε, πολιτικών οικογενειών που εκπροσωπούνται και στο Συμβούλιο, αλλά και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, υπάρχουν αποκλίνουσε διαφορετικέ μεταξύ του απόψει. Θέλω να ευχαριστήσω ε, και τον κύριο Λάμπερτ, πολύ λογικά λέει ότι δεν είναι ομοφωνία η πλειοψηφία και ε, με την πλειοψηφία μπορούμε κάποιες φορές να πετύχουμε, να κάνουμε το βήμα προς τα εμπρός. Ε, δεν άκουσα ακριβώς τα ίδια μηνύματα ε, από όλου. Και σίγουρα φαίνεται να υπάρχει κοινή θέση από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου και αυτό είναι θετικό, ενθαρρυντικό και το λαμβάνω υπόψη. Στο Συμβούλιο πρέπει να εργαστούμε για να προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε ομοφωνία. Δεν είναι απλό αυτό. Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι. Αυτό είναι σημαντικό και γι' αυτό είμαστε κινητοποιημένοι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τι αξίε και το κράτο δικαίου, όπω και πολλοί από εσά είπατε, η διακυβέρνηση, το κράτος δικαίου, οι θεμελιώδει αξίες πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι σπονδυλική στήλη αυτού του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Θα πρέπει να το λέμε υπόψη και αυτή είναι η πολιτική στιγμή, η χρονική στιγμή για να βαθίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, με αυτή τη φιλοδοξία. ολοκληρώνοντα θέλω να σα πω ότι από τη δική μου την πλευρά ε, και αυτό το έδειξε η κρίση, η ευημερία δεν τη κανεί με ένα δίκτυ την ανάπτυξη, την ποσοτική ανάπτυξη. Εδώ και δεκαετίες θεωρούμε ότι η πρόοδο μπορεί να μετρηθεί με μία παράμετρο μόνο, με ένα κριτήριο που είναι το, το ποσοστό του ΑΕΠΑ. Δεν αρκεί δεν αντικατοπτρίζει αυτή τη στιγμή ε, τη συγκεκριμένη εντύπωση που έχουν οι πολίτες ε, των δεδομένων χωρών της Ένωσης. Ε, πώς νιώθουν ότι ζουν, ζουν καλύτερα από πέρυσι ή από κάποιες χρονιές. Αυτό είναι ο δείκτη. και γι' αυτό σε αυτή τη φάση μετασχηματισμού που βρισκόμαστε θα πρέπει ίσω να διορθωθούμε και πώς θα προωθήσουμε αυτές τις οικονομικές και κοινωνικές μεταρρυθμίσεις, αλλά να κάνουμε μια δημοκρατική συζήτηση ε, για να θέσουμε στόχους, ε, τους επιθυμητούς ε, στόχους, ευκταίους στόχους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε το θέμα του περιβάλλοντος, της εκπαίδευσης, της, του περιορισμού των ανισοτήτων, πρόσβαση σε ποιοτικέ υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις. Αυτές είναι οι παράμετροι που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για να μετρήσουμε την πρόοδο που είναι εφικτή χάρη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα, χάρη στο ευρωπαϊκό εγχείρημα που πρέπει να συσπηρώνει και όχι να διαιρεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Πρόεδρε Μισελ. Συνεχίζουμε τη συζήτηση. Ο κύριος Νόβακοφ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, θα μιλήσω την ε, μετρική μου γλώσσα, βουλγαρικά. 60 δευτερόλεπτα δεν αρκούν για μια πραγματική ομιλία. Εμεί όμω οι Βούλγαροι θεωρούμε ότι αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε είναι πράξεις και όχι λόγια. Καλή τύχη στη Γερμανική Προεδρία. Ξεκινά πραγματικά ε, στο μέσο μια ε, κρίση, τη κρίση του COVID-19. Και επίση πρέπει να αναλάβουν και ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα που μπορεί να προκαλέσει καινούργια κρίση. Οι προτεραιότητε τη Προεδρία έχουν στόχο διτό τη ζωή και την υγεία των ανθρώπων και το να σώσουμε την οικονομία και τι θέσει εργασία. Δεν ξέρω τι θα γίνει με την υγεία τη Ένωση τη ίδια, αλλά ο COVID-19 φαίνεται να έχει πλήξει την κοινή τη λογική. Το πακέτο αυτό είναι μόνο μια αρχή και πραγματικά για όλους τους συναδέλφους θα ψηφίσουν υπέρ. Ε, ξέρετε ε, τι ψηφίζετε πραγματικά, το διαβάσατε, ε, έχετε την αίσθηση ότι προστατεύετε τα δικαιώματα των εργαζομένων. Και εγώ αυτό επιθυμώ. Αλλά αυτή τη στιγμή μιλάμε το να εργάζονται ευθύ εξ αρχή και να έχουν έστω ένα μισθό, κάποια αμοιβή. Πρέπει λοιπόν να ψηφίσουμε κάτι που να έχει κάποιο νόημα. Δεν θα έχουμε καμία επιτυχία κλιματικέ αλλαγέ και την καταπολέμησή του, αν κυκλοφορούν άδεια φορτηγά και τα σε όλη την Ευρώπη. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει και με τους οδηγούς φορτηγών και ταλικών. Πρέπει να ε, διαλέξουμε μεταξύ του σωστού ε, και του εσφαλμένου. Ε, ο κύριος Μπενιθέη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της επόμενης εβδομάδας θα έχει μια ζωτική αρμοδιότητα να πετύχει συμφωνία για τον προπολογισμό και τα δημοσιονομικά και αμέσως με το πρόγραμμα ανάπτυξης το ε, Κοινοβούλιο έχει χρησιμοποιήσει ω σημείο εφετηρία την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όμω, αν κάποιο στο Συμβούλιο θεωρεί ότι θα πρέπει να πιέσει το Κοινοβούλιο να δεχτεί κάτι, σφάλει. Το Κοινοβούλιο είναι έτοιμο να απορρίψει οποιαδήποτε συμφωνία που θα είναι χειρότερη από την αρχική πρόταση που έχουμε μπροστά μα, επιτάπητο. Ω Ευρωβουλευτέ, γνωρίζουμε ότι σήμερα πρέπει να δείξουμε τόλμη. Το περιμένουν εκατομμύρια πολίτε που αυτού του μήνε έχουν υποφέρει από την πανδημία. Απλώ μια νέα φάση τη ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης ε, δεν μπορεί απλώς να μας βγάλει από την κρίση πιο ισχυρούς και πιο ε, ε, ενωμένους. Χρειάζονται και ήδη πόροι. Χρειάζονται φόροι για τους γίγαντες του ίντερνετ, για την καταπολέμηση της φορολογικής κερδοσκοπίας, σε όσους έχουν συμβάλει ελάχιστα για την ευημερία των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μας. Το, το Συμβουλίο πρέπει να λάβει μια ιστορική ευθύνη άνευ προηγουμένου και πρέπει να βρεθεί στο των περιστάσεων και εμεί πρέπει να υποστηρίξουμε ε, από την πλευρά μας τους πολίτες. Το Συμβούλιο θα πρέπει να δείξει ότι είναι διατεθειμένο να κάνει το ίδιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βιλίμσκι για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, ε, εδώ και λίγες μέρες είχαμε μια, εδώ και, λίγο, και λίγες είχαμε μια σοβαρή διακοπή για να βρεθούμε αδύναμοι και να καταλάβουμε πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να ξεπεράσουμε κάθε πρόβλημα. Εδώ στο, μέσος, στο μέσο μιας κρίσης πρέπει να παραδεχτούμε ότι εκεί που πολλές φορές ε, μπορούν να λυθούν πολλά πράγματα σε εθνικό επίπεδο από ό,τι πετυχαίνουμε να κάνουμε εδώ. Και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πολλές φορές δεν είναι εκείνη που επιλύει τα προβλήματα, αλλά ακριβώς ε, υποδαβλίζει τις πρικαγιές. Θα πρέπει λοιπόν πολλά προβλήματα να τα δούμε ε, από άλλη οπτική γωνία. Και εδώ για το Συμβούλιο αυτό και τα δημοσιονομικά θέματα, το να ε, εκμεταλλευόμαστε την κρίση του κορονοϊού για να πάρουμε στα χέρια μας και περισσότερες αρμοδιότητες, περισσότερε εξουσίε και να πιέσουμε περισσότερε προποθέσει στα κράτη-μέλη είναι κάτι που θα δημιουργήσει προβλήματα. Όχι και άλλε αρμοδιότητε τη Βεξέλη, το ανάποδο, πίσω στα εθνικά κράτη. Αυτό θέλουμε να ευχηθούμε. Ευχαριστώ πολύ. Για ένα λεπτό ο κύριο Άντρεσεν. χρόνο χρόνο χρειάζεται ώστε οι αρχικοί κρατών και κυβερνήσεων να αφήσουν του εθνικού του εγωισμούς και τα όρια που επιβάλλουν. Πρέπει να δουν ότι το μέλλον μα πρέπει να είναι κοινό. Τα εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν πρέπει να είναι συμβατά με την κλιματική συμφωνία που θα βρεθεί και να υπάρχουν περισσότερε προσπάθειε από όλου. Ε, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων πρέπει να ε, λάβουν μεν την υποστήριξη, αλλά αυτά θα τα μπορούν να τα διαχειριστούν μόνο οι, αρχι... οι άρχοντε τη τοπική αυτοδιοίκηση επιτόπου και οι εθνικοί κυβερνήτε. Θα πρέπει λοιπόν να δείξουμε εμπιστοσύνη στην δημοκρατία μα και ε, θα πρέπει για τον κοινό μα προπολογισμό να βρούμε μια συμβαστική λύση. Οι κλιματικέ αλλαγέ, η προστασία τη φύση, ε, το πρόγραμμα Εράσμου, οι αρχέ τη δημοκρατία είναι κρίσιμε αξίε και αρχέ οι οποίε δεν μπορούν να υποβιβαστούν. Εκεί θα πρέπει να επιμείνουμε στην επίτευξη μια συμφωνίας. Ευχαριστούμε. Για ένα λεπτό, ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, θα έλεγα ότι η στιγμή αυτή, το επόμενο Συμβούλιο, είναι κρίσιμη στιγμή για την Ευρώπη. Η οικονομική κρίση και οι κοινωνικέ και εργασιακέ ανισότητε, καθώ και οι φορολογικέ ή δημοσιονομικέ ανισότητε των εκδοτών, πλήττουν την ε, εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτέων. Θα πρέπει ε, να δούμε ένα φιλόδοξο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο με την πρόταση που θα διαμορφώσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ζητώντα τι κατάλληλε προσπάθειε από την οικονομία με επενδύσει σε βιώσιμου και αντιμετωπίζοντα και τη φορολογικό ανταγωνισμό μεταξύ των κρατών μελών. Δεν πρέπει να ασφάλουμε ζητώντα συμφωνίε με χαμηλότερα ποσά για χώρε που έχουν ε, μόνο ωφέλη αντλήσει από την κοινή αγορά. Δεν θα πρέπει να επιβάλλουμε προγράμματα λιτότητα, όπω με το μηχανισμό σταθερότητα ε, και το πρόγραμμα που είχε επιβληθεί επί Επιτροπή Juncker. Θα πρέπει να τα δουν αλλιώ ε, η, ε, η καγκελάριος Μέρκελ και η Γερμανική Προεδρία όχι να ε, ξαναπεράσουμε σε λατασμένες συμφωνίες. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό κυρία Νίμπλερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αγαπητοί συνάδελφοι. Το πρώτο σε ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή ε, στα κράτη-μέλη που γίνεται η συζήτηση δεν βλέπουμε καμία πρόοδο. Το είπε και ο κύριος Μούρεσαν και πραγματικά αυτό αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικαίωμα συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε αυτέ τι αποφάσει. Δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Σε ό,τι αφορά το σχέδιο ανάκαμψη, χρειάζεται ένα φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψη. Πρώτον, γιατί έχουμε εκατομμύρια ανέργων ε, ή ε, σε προσωρινή ε, ανεργία και επίση υπάρχουν πάρα πολλέ επιχειρήσει που απειλούνται με πτώχευση, με χρεοκοπία, αφήνοντα δηλαδή στο δρόμο και πολλού άλλου εργαζομένου. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχθούμε. Άρα απαιτείται γρήγορη απόφαση. Και ο δεύτερο λόγο είναι ότι αν τώρα κάνουμε οικονομίε και είμαστε φιδωλοί, θα μα κοστίσουν τα διπλά, μην πω και τα τριπλά στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει τώρα να δούμε σωστά πώς θα ε, διαμορφώσουμε το μέλλον, να επενδύσουμε στους πολίτες μας ε, στην ε, δημιουργία νέων υποδομών, ανάπτυξη υποδομών και να μην αφήσουμε στα παιδιά μας μόνο χρέη, την αποπληρωμή δηλαδή. Θα πρέπει τώρα να κανονίσουμε όλες αυτές τις εκκρεμότητες πριν αρχίσει η επόμενη και περίοδος. Ευχαριστώ πολύ. ευχαριστώ πολύ. Μορένο Σάντσεθ, ευχαριστώ πολύ. Δεν ακούγεται ο μιλητή. Τώρα, sí. Τώρα, ωραία. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το σχέδιο ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης διέρχεται μια αποφασιστική ε, στιγμή και χρειάζονται, δραστικέ χρειάζονται δραστικές αποφάσεις θα πρέπει λοιπόν ε, στην επόμενη σύνοδο κορυφής ε, να επιδειχθεί θάρρος από την Προεδρία και από τη σοσιαλιστική οικογένεια για να προχωρήσουν προς τα εμπρός ε, με ένα φιλόδοξο πρόγραμμα το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το δυνατό. Έφτασε επίση η στιγμή για να εισαχθούν νέοι διπόροι στην Ένωση, για να δώσουμε νέα ε, πνοή στις επιχειρήσεις και στους πολίτες και αισιοδοξία. Και επίσης θα πρέπει ένα ε, στεναρό γενναίο σχέδιο μετανάστευσης ε, να εγκριθεί για τις νόμιμες οδούς μετανάστευσης που είναι καλύτερη οδός καταπολέμησης της παράτυπης μετανάστευσης. Το 2015 πολλές χιλιάδες πρόσφυγες βρήκαν την καταφυγή εκεί. Θα πρέπει δύο τώρα γυναίκε από τη Γερμανία να δείξουν το, το, ίδιο στέλνο και να έχουμε αυτό το σχέδιο μεταναστευτικό. Ευχαριστώ πολύ. Last month, the commission... Πρόεδρε, την περασμένη εβδομάδα στο site της Κομισιόν έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να χρηματοδοτήσει τον προπολογισμό της μέσω του δανεισμού. Τώρα αυτό έχει διαγραφεί ο το κράτος δικαίου είναι αστείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν το ακολουθεί. Και η εσωτερική υπόθεση του από ποιο, ποιος παίρνει τα χρήματα και ποιος τα δίνει ε, είναι αναπάντητη. Η Βαντρελάιεν τονίζει ότι τα κράτη-μέλη δεν θα πρέπει να σκεφτούν μόνο το δικό τους καλό, αλλά το κοινό καλό. Μα τι ακριβώς εννοεί. Το 2011 οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες ήταν. Τώρα πρέπει να στηρίξουμε τις γαλλικές και τις ε, ε, ιταλικές τράπεζες. Πόσες ακόμα χώρες θα πρέπει να χρεωθούν ακόμη περισσότερο πριν να σταματήσει όλη αυτή η τρέλα. Ένα λεπτό ο κύριος Κορμό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Πώς να μην καταλάβουμε τις ιστορικές στιγμές που διανύουμε. Πώς να μην δούμε ότι απέναντι στις κρίσεις, τις οικολογικές, τις κοινωνικές, τις οικονομικές θα πρέπει εμείς να προστατέψουμε τους Ευρωπαίους και τις Ευρωπαίες, τις θέσεις επασχόλησής τους, τις οικονομίες μας, χωρίς να υποβαρύνουμε άλλο το κλίμα. Η Ευρώπη είναι στριμωγμένη στους διαδρόμους του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στα παζαρέματα ανάμεσα στα κρατημέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να αντιδράσει γιατί η λήψη ιδίων πόρων παραμένει φυλακισμένη ανάμεσα στους εθνικούς εχοισμούς. Ήδη οι πόροι θα σήμαινε ότι θα είχαμε τη δυνατότητα όχι μόνο την οικονομική αλλά και την πολιτική να δράσουμε. Δηλαδή να διατηρήσουμε το νόημα της ύπαρξής μας ως πολιτική οντότητα και ως σημαντικός φορέας. Ε, αν δεν επιμείνουμε γι' αυτό θα οδηγηθούμε στην εξαφάνισή μας προς μεγάλη χαρά των λαϊκιστών της Ευρώπης αλλά και προς μεγάλη χαρά των οικονομικών συμφερόντων που κερδοσκοπούν πάνω στις δικές μας αδυναμίες και προς ε, ε, μεγάλη δυστυχία των λαών. Ευχαριστώ κύριο Σταγιάννη. Για ένα λεπτό. Ο κοροναϊός έχει θέσει υπό συζήτηση την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλή η δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και η γραμμή ε, πίστοσης για προστασία της υγείας μας. Είμαι επιπισμένος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα 36-37 δις ε, για να βελτιώσει τις υγειονομικές της ε, δομές ενώπιον και μιας ίσως δεύτερης, ενός δεύτερου σχήματος της πανδημίας. Αλλά τώρα έχουμε το Συμβούλιο το Ευρωπαϊκό και 18 Ιουλίου. Πρέπει οπωσδήποτε να υπερασπιστούμε την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι βόρειες χώρες που θεωρούν ότι μπορούν να περικόψουν τις δράσεις που στηρίζουν την ανάπτυξη κάνουν λάθος. Πρέπει να συνεχίσουμε να έχουμε επενδύσει και δάνεια ώστε να μπορέσει η βιομηχανία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η γεωργία να ξανασηκωθούν, να σταθούν στα πόδια τους μετά από αυτή την κρίση. Θα ήταν λάθος να μην το κάνουμε και θα ήταν επικίνδυνο για την ίδια την επιβίωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Τώρα η κυρία Μαργαρίδα Μάρκες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, το έχω πει και το επαναλαμβάνω ότι αυτή η συνολική πρόταση της Κομισιόν για το ΠΔΠ και για το σχέδιο ανάκαμψης είναι μια πρόταση δημιουργική καινοτόμα και πρέπει να χαιρετήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μπόρεσε να βρει τις απαραίτητες απαντήσεις στο πλαίσιο της ε, ε, των αρμοδιοτήτων της. Είναι η βάση για την ευρωπαϊκή απάντηση στην κρίση. Είναι μια απάντηση που πρέπει να δοθεί αλλά και μια ανάκαμψη για τις οικονομίες μας. Ε, και ε, η Κομισιόν έχει ε, ενεργοποιήσει το άρθρο 324, το ενώ το Συμβούλιο πάει πολύ αργά σε αυτή τη διαδικασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει βρει πλειοψηφίε. Ο κίνδυνος αυτό εδώ το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι ότι η επίγουσα κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη ρεαλισμού. Όμως δεν μπορούν όλα αυτά να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον. Το σχέδιο είναι κλειδί για να μπορέσει η, κρίση να, Ευρώπη να βγει από την κρίση και το ΠΔΠ είναι το κλειδί για τις επόμενες γενναίες. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πίπερ. Κυρία Πρόεδρε, κύριε Σεύκοβιτς, 500 δις ευρώ ε, πέραν του ευρωπαϊκού προπολογισμού τεράστια ε, πρόκληση για την Ευρώπη, κυρίως για να ε, χρησιμοποιηθούν εποφελώς αυτά τα κονδύλια, για να υπάρξει πραγματικά ανάκαμψη μετά την κρίση του κορονοϊού, για να φροντίσουμε το μέλλον των νέων μας και για να επενδύσουμε και σε ένα οικολογικά λογικό μέλλον. Όμως έχω πολύ λίγη εμπιστοσύνη στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και σε κύριε δυστυχώς και αυτό φαίνεται και από τη στάση του κυρίου Μισελ εδώ τώρα. Ελπίζω στις οικονομικές και δημοσιονομικές ε, διαπραγματεύσεις τα πράγματα να πάνε αλλιώ. Θα πρέπει φορολογούμενοι ε, να δουν επιτέλους όλα αυτά που έχουν προσφέρει τα τελευταία χρόνια να αξιοποιούνται. Για θέματα όπως η ενέργεια, το εράσμος, η ψηφιοποίηση, ε, ο έλεγχος, το δικαίωμα βέτο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκή Προσταθέμενη Αξία, το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Θα πρέπει όλα αυτά να μην είναι αντίφαση. Ε, θα πρέπει απλώς να υπάρχει περισσότερη και δυνατότερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό περιμένουν από εμά οι πολίτες. Ευχαριστούμε κύριο Στάνι, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σε καιρούς ε, κορονοϊού και οικονομικής ύφεσης οι άνθρωποι θέλουν νίκες ε, και χειροπιαστέ λύσεις, όχι ε, συγκρούσεις βορρανότου. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει άμεση οικονομική υποστήριξη, επενδύσεις στην εσωτερική αγορά, όχι ε, όμως να παραβλέπουμε ε, ποιοι δεν έχουν συμβάλει ως τώρα στην ε, ευρωστία της ε, ευρωπαϊκής οικονομίας να πληρώσουν για όσα έχουν ωφεληθεί ως τώρα να μην ε, αναλάβουν στους ώμους τους ε, οι φορολογούμενοι την ανάκαμψη, να πληρώσουν ε, οι επιχειρήσεις που έχουν κερδίσει τα περισσότερα στην Ευρώπη, που είναι οι πλέον κερδοφόρες και πλούσιες. Όχι να πλήξουμε τους μικρούς φορολογουμένους και θα πρέπει να πάψουμε πλέον τους τσακωμούς και τις διαφωνίες μεταξύ μας. Οι πολυεθνικές να ε, καλύψουν ε, τις ανάγκες που έχουμε. Να έχουμε μια Ευρώπη που να είναι για όλους ε, χρήσιμη και επωφελής. Ευχαριστούμε κυρία Χόλμαγερ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, ε, κύριε Πρόεδρε της, ε, Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κυρίες και κύριοι, είναι τεράστιο το δημοσιονομικό πακέτο που έχουμε μπροστά μας και θα ήθελα εδώ να πω ξεκάθαρα ότι το ευρωπαϊκό ε, Εξάμεινο δεν είναι ο κατάλληλη διαδικασία για να ελοποιηθούν όλα αυτά. Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αυτά που δίνει το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Εδώ χρειαζόμαστε χειροπιαστές λύσεις και χρειάζονται ε, οικονομικές ροές που να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα project και προγράμματα για αυτούς που πραγματικά είναι δικαιούχοι και χρειάζονται τα χρήματα. Και εμείς να μπορούμε να ελέγξουμε εάν οι ειδικέ επιτροπές ε, έχουν... Ε, να μπορούν οι οικονομικές επιτροπές να ελέγξουν κατά πόσο τα κονδύλια έχουν δαπανηθεί σωστά. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει η σωστή συγκέντρωση δεδομένων ακριβώς για όλα αυτά τα θέματα ε, με ένα ψηφιακό σύστημα που να μπορεί να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και να μπορούν όλα αυτά να δικαιολογηθούν και οικονομικώς στο κοινό, να είναι διαφανή, να μην ε, γίνεται ως τώρα επί να πλημμένει κανείς τις πληροφορίες, να πρέπει να κάνει έρευνες ε, και αναζητήσεις μέχρι να βρει τα απαραίτητα στοιχεία και για τα προγράμματα και για το θεματοβουτισίκους. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Κάρας για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Η διάσκεψη των αρχηγών κρατών κυβερνήσεων είναι λιδία διαλύθος ε, ε, για να δούμε κατά πόσο θα αναγνωριστούν αυτά τα οποία είπε η σήμερα η κυρία Μέρκελ, ποιε είναι οι ανάγκε ε, και ποιοι είναι οι στόχοι. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει τα βασικά σλόγγαν τη Γερμανική Προεδρία. δεν μπορώ να το πω αυτό για όλους ε, τους επικεφαλείς των κρατών Θέλουμε λοιπόν μια πιο ε, ισχυρή Ευρώπη και δεν θα πρέπει ε, να έχουμε τις οικονομίες, ε, την εξοικονόμηση πόρων ως μόνο γνώμονα. Θα πρέπει σίγουρα την καινοτομία, την ψηφιοποίηση να προωθήσουμε στην Ευρώπη. Και σίγουρα πιέζει ο χρόνος, ποιος δεν το αναγνωρίζει. Και αν δεν το αναγνωρίζει κλείνει το μά, τα μάτια μπροστά ε, στις ε, δημοκρατικές, κοινωνικές, πολιτικές, οικονομικές συνέπειες της κρίσης. Ε, όποιος επίσης δεν αναγνωρίζει ότι χρειάζεται σθένος, κουράγιο, επίδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης, ε, ε, γιατί περί αυτού πρόκειται, αυτό είναι το μέλλον της Ευρώπης, εκεί βασίζεται, δεν μπορεί να το, ε, μην να το αναγνωρίζει κάποιος αυτό. Υπάρχουν επίσης κάποιοι που μπλοκάρουν, αυτοί που μπλοκάρουν ευθύνονται για το μέλλον της ε, Ευρώπη, αν δεν ε, έχουμε αίσιο πέρα σε όλες αυτές τις παραπαγματεύσεις και ε, δεν θα πρέπει να την πληρώσουν. Ευχαριστώ πολύ κύριο Χριστοφόρου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κρίνω ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προβαίνει σε μια ιστορική συνάντηση και σε ένα ιστορικό συμβούλιο. Δεν κρίνεται η έγκριση η απόρριψη του οικονομικού πακέτου για να στηριχθούν οι χώρε, οι οικονομίε του αλλά και οι πολίτε κρίνεται η ίδια η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει και μπορεί να πάει μπροστά και να διασφαλίσει το μέλλον της Ευρώπης αλλά και των επόμενων γενιών. Άρα για μένα είναι αδιανόητο και θα συμφωνήσω πλήρως και με τις προηγούμενες τοποθετήσεις των συναδέλφων να υπάρξει οποιοδήποτε διαχωρισμός βορρά και νότου. Εάν ο νότος πτωχεύσει θα πτωχεύσει αυτόματα και ο βορράς και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση οποιοδήποτε διαχωρισμό είναι ενάντια τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που κάνει είναι βάζει νερό στο μήλον των λαϊκιστών και των εθνικιστών. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σέβεται το κράτο δικαίου, τι αρχέ και τι αξίε οι οποίε είναι θεμελιώδει και δεν πρέπει να δίνεται ούτε έναν ευρώ σε χώρε οι οποίε τι παραβιάζουν. Πρώτη και καλύτερη παραβιάζει αυτέ τι αρχέ και τι αξίε η Τουρκία, η οποία επιτίθεται σε χώρε μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά προσβάλλει και ακόμα και τα θρησκευτικά μα αισθήματα θέλοντας να μετατρέψει έναν οικουμενικό σύμβολο χριστιανισμού και πολιτισμού την Αγία Σοφία σε τζαμί. Αυτές οι χώρες δεν έχουν θέση στα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ προτείνω να αποκλειστεί η Τουρκία από το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Πρόεδρε. Ανάκαμψη εμπιστοσύνη δεν νοείται. Ε, εμπιστοσύνη των πολιτών. Πρέπει να την ανακτήσουμε. Βλέπουμε ότι για να γίνει αυτό χρειάζεται και κυριαρχία σε στρατηγικούς τομείς όπως είναι ψηφιακός τομέας, τα τρόφιμα, η άμυνα, η ασφάλεια φυσικά, είδαμε και η υγεία είναι σε από αυτούς τους τομείς. Και φαντάζομαι ότι εκεί πρέπει να προσανατολιστούμε για να δώσουμε μεγαλύτερη ισχύ στην Ευρώπη. Και το σχέδιο ανάκαψης θα πρέπει να έχει και ενισχυμένους ίδιους πόρους εν μέρη από το φόρο ε, του άνθρακα στα σύνορα ή των μεγάλων ομίλων, ε, ψηφιακό φόρο. Θέλουμε επίσης περισσότερη αυτονομία και ε, κυριαρχία και να αποφύγουν τον εκβιασμό κάποιων κρατών μελών που παίζουν με το μέλλον όλων των Ευρωπαίων. Θα πρέπει να ξαναβρούμε λοιπόν την αυτονομία και την κυριαρχία της Ευρώπης ε, γιατί ε, θα κάνει τους Ευρωπαίους να εμπιστευτούν την Ευρώπη και νομίζω ότι έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε μια νέα πνοή σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Κυρία Βίρκουνεν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, για το μέλλον της Ευρώπης αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι κοινέ λύσεις και απαντήσει σε τρία ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα, Ευρώπη και οικονομική κρίση. Τι απάντηση θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα. Χρειάζεται κοινή απάντηση, αυτό είναι σαφές. Οι επενδύσεις θα πρέπει να ε, βοηθήσουν στην ε, αηφόρο ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Το δεύτερο ερώτημα, πώς θα αποπληρωθούν τα δάνεια και τα κράτη-μέλη θα πρέπει επίσης ε, να να είναι κράτη δικαίου και να τηρούν στην πράξη αυτές τις ε, υποχρεώσεις τους. Θα πρέπει λοιπόν να συνδέεται η εκταμείωση των κονδυλίων με το κράτο δικαίου. Και το τρίτο είναι η μετανάστευση. Και ελπίζω και επί την γερμανική ηγεσία να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινή γραμμή και σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρο. Να δώσω στον κύριο Σεύκοβιτ, τον αντιπρόεδρο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για μια ακόμη φορά το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ μου δίνετε το λόγο. Μίλησα πολύ στις εισαγωγικέ μου παρατηρήσεις και γι' αυτό θα είμαι τώρα πιο σύντομος. Θα απαντήσω στα τέσσερα πιο συχνά ε, θέματα τα οποία αναφέρθηκαν. Καταρχάς, ε, η αίσθηση του επίγοντος που αναφέρθηκε από τον κύριο Μουρεσάν, τον κύριο Νάντερς και άλλους, αλλά και στον κύριο Ταγιάννη, ο οποίος τόνισε πόσο σημαντικό είναι να σταλεί ένα πολύ ισχυρό μήνυμα τώρα και νομίζω πως αυτή θα πρέπει να είναι η απόλυτη προτεραιότητα για τους ηγέτες μας, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο, ότι πρέπει να ληφθεί απόφαση στο επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί αυτό θα ήταν το καλύτερο μήνυμα, η καλύτερη απάντηση που θα μπορούσαμε να δώσουμε στους πολίτες μας. Ε, η καλύτερη απάντηση στην κρίση θα μας βοηθούσε να εξασφαλίσουμε θέσεις απασχόλησης, να τις ε, προστατέψουμε και θα ήταν και ένα μήνυμα προς τους παγκόσμιους εταίρους μας, τις οικονομικές, τις ε, χρηματαγορές, ότι η Ευρώπη επανήλθε, ότι ξεπερνά τα προβλήματα και ότι βγαίνει από την κρίση ισχυρότερη. Δεύτερο πάρα πολύ σημαντική ομάδα παρατηρήσεων αναφερόταν στις κοινωνικές επιτυχίες και στο κατά πόσο οι πολιτικές που προτείνουμε θα μπορέσουν να διεισδύσουν ώστε να τονίσουμε την ψηφιακή μας μεταρρύθμιση μαζί με και να αυξήσουμε την αθεκτικότητα. Ε, θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι το σχέδιο ανάκαμψης συντάσσεται από τα ίδια τα κρατημέλη. Φυσικά θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως τα ζητήματα, τα συγκεντρωμένα προβλήματα τα οποία ε, δημιουργούνται χρόνο με το χρόνο στα κράτη-μέλη θα αντιμετωπιστούν ότι σταδιακά θα μπορέσουμε να τα αντιμετωπίσουμε και να επιτύχουμε την ανθεκτικότητα στα κράτη-μέλη μας ε, που θα είναι ισχυρότερη και για ολόκληρη την Ένωση. Φυσικά ε, θέλουμε να υπάρξει η συνεργασία με τα κράτη-μέλη και είμαστε έτοιμοι να ε, ενημερώσουμε το Ευρωκοινοβούλιο, πράγμα που κάνουμε πάντοτε στις διαβουλεύσεις και υπό το διαρθωμένο διάλογο και στις ακροάσεις που ερχόμαστε μέσα στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα επιβλέπει το σύνολο των δαπανών όπως το κάνει και τώρα όταν εξετάζει τις ε, δαπάνες επί βάσης το, αυτό ήταν και το νόημα των παρατηρήσεων της κυρίας Σομπρί, του κύριου Πίρσεν συγγνώμη, και της κυρίας Χολμάγερ, ότι δηλαδή θα πρέπει να είναι διαδικασία διαφανής και ότι ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ενημερώνεται και ο ρόλος του θα ε, διατηρηθεί. Θα έρθουμε σύμφωνα με το άρθρο 324 σε, έχουμε συνάντηση με τους ηγέτες μας και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε πρόταση για θεσμική δήλωση που θα τοποθετήσει σε πολύ σαφές πλαίσιο πώς βλέπουμε δηλαδή την συνεργασία ανάμεσα στους θεσμούς για τα σημαντικά τμήματα της εφαρμογής του Next Generation EU και ε, της εφαρμογής του και εκτέλεσης αυτού του project στο μέλλον. Τέλος, Λάρσεν Μπενιφέη και άλλοι μιλήσατε για τους ίδιους πόρους και φυσικά και πρόκειται για πολύ σημαντικά ζητήματα γιατί πρέπει να προτείνουμε νέους τρόπους για το πώς θα πληρώσουμε με τα χρήματα τα οποία θα ε, βρούμε στις ε, χρηματοπιστωτικές αγορές και μέσα από το ε, μέσο ανάκαμψης. Εμείς όπως είπαμε, έχουμε το σύστημα εμπορίας εκπομπών, αλλά και το σύστημα για τον άνθρακα, αλλά και μέσω της συνεργασίας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ενιαία και το ψηφιακό ε, φόρο. Και προσπαθ... συνεχίζουμε να εργαζόμαστε επί διαφόρων ιδεών ε, για τους ίδιους πόρους και θα τα συζητήσουμε μέσα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε έτοιμοι να δουλέψουμε για να ε, δούμε, να δούμε πώς θα αξιολογήσουμε και πώς θα συζητήσουμε αυτές τις, ε, τους πιθανούς ε, ίδιους πόρους που είναι πολύ σημαντικοί όπως ξέρουμε για αυτό το κοινοβούλιο αλλά και για τα εθνικά κοινοβούλια γιατί εάν θέλουμε να αυξήσουμε τα κατόφλια και των πόρων και της χρηματοδότησης θα πρέπει να έχουμε τη στήριξη όλων των Εθνικών Κοινοβουλίων της Ένωσης. Σας ευχαριστώ λοιπόν κατακλείδη για τη στήριξή σας, για την αίσθηση του επίγοντος, για τη βούλησή σας να συνεργαστείτε με αυτό το τόσο δυναμικό τρόπο, γιατί θα χρειαστεί για το επόμενο εξάμεινο και προσβλέπω στη συζήτησή μας και πάλι να είστε βέβαιοι πως ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα διατηρηθεί όπως δει. Σας ευχαριστώ πολύ Αντιπρόεδρε Σεύκοβιτς. Τώρα η κοινή συζήτηση ολοκληρώθηκε και ε, μέχρι τις 7 ε, σταματάει η συνεδρίαση.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

το ποτό 1, 2, 3. Ξεκινάει η συνεδρίαση, ε, ξεκινάει η καταγραφή των πρακτικών. Οι αρμόδιες Γαλλικέ αρχές έστειλαν μια αίτηση στον πρόεδρο για την άρση της βουλευτικής ασυλίας ε, του κ. Γιάλκα στο πλαίσιο ε, μιας αίτησης έρευνας σε ένα γαλλικό δικαστήριο του Παρισιού ε, έχει σταλεί το αίτημα στην ε, αρμόδια επιτροπή του Κοινοβουλίου. Περνάμε στις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, για την συνολική πολιτική της Ένωσης για την πρόληψη της νομιμοποίησης των παρανομής δραστηριότητας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Το σχέδιο δράσης της Επιτροπής και άλλες πρόσφατες εξελίξεις. να πω στους συναδέλφους ότι δεν θα υπάρξουν ούτε μπλε κάρτες ούτε αυθόρμητες αγορεύσεις οπότε δίνουμε στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής το λόγο στον κύριο Ντομπρόφσκης. Καλώς ορίσατε και Καλωσορίζουμε και τον κύριο Μιχάλη Γότα από το Συμβούλιο, στον οποίο δίνω το λόγο. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμες κύριε και κύριοι βουλευτές. Είναι πρώτη φορά για μένα πριν από... Είμαι εδώ και 22 χρόνια βουλευτής ε, στο Κοινοβουλίο της χώρας μου και εδώ και 7 χρόνια ε, αναπληρωτής υπουργό ε, για τα ευρωπαϊκά θέματα. Ποτέ δεν έχω όμως μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οπότε σήμερα μιλώ εκ μέρους του Συμβουλίου και είμαι ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία και χαίρομαι για τους ε, μήνε που θα ακολουθήσουν και θα είμαι πάντα στη διάθεσή σας και χαίρομαι για την επικοδομητική και επικριτική συνεργασία που θα έχουμε σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Η καταπολέμηση του ξεπλήματο βρώμικου χρήματο και της ε, χρηματοδότησης της τρομοκρατίας είναι ένα από τα κεντρικά θέματα της ε, Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου. Όπως γνωρίζετε είναι ένα θέμα το οποίο ε, βρίσκει το Συμβούλιο να αφιερώνεται σε αυτό με μεγάλη προσοχή και το, ε, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή έχουν συνεργαστεί τα τελευταία χρόνια για να βρουν ένα κοινό σύστημα για την καταπολέμηση της ε, νομοποίησης εσόδων παράνομης δραστηριότητας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. μπορούμε να πούμε ότι έχουν γίνει σημαντικές πρόοδροι και ε, με τη σχετική νομοθεσία χάρη στη δική σας δέσμευση ε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ε, να υπενθυμίσω την αλλαγή της οδηγίας για την καταπολέμηση του ξεπλήματος, την κανονισμό για την Ευρωπαϊκή Αρχή Επιτήρησης των Τραπεζών και διάφορα άλλα νομοθετικά μέσα τη χρήση οικονομικών δεδομένων για την δίωξη άλλων εγκλημάτων. Αλλά κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να επαναπαυόμαστε στις δάφνες μας. Συχνά θυμόμαστε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές υποθέσεις ε, ε, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών τραπεζών. Κάτι απαράδεκτο. Στο ενδιάμεξο εσείς και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχετε αναπτύξει έναν ολοκληρωμένο διάλογο και συζήτηση για το ποιο θα είναι το πλαίσιο για την καταπολέμηση τη νομιμοποίηση εσόδων παράνομη δραστηριότητα και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία με πιο αποτελεσματικό τρόπο στο μέλλον. Τι πρέπει να κάνουμε, τι μπορούμε απλά να βελτιώσουμε. Τα δικά σας ψηφίσματα, ε, τα δικά μας συμπεράσματα και η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, είναι υποδειγματικά για όλο αυτό τον προβληματισμό, αλλά δεν πρέπει να παραμείνουμε σε προβληματισμούς και συζητήσεις. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα που καθιστούν σαφές ε, το πώς εμείς έχουμε δεσμευτεί το Δεκέμβριο του 2018 το Συμβούλιο ε, ψήφισε ένα συγκεκριμένο σχέδιο ε, δράσης για την καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος. Το Δεκέμβριο του 2019 ξεκίνησε με την υιοθέτηση στρατηγικών συμπερασμάτων το Συμβούλιο όπου οι Κομισιόν και οι υπόλοιποι ε, ε, αναζήτησαν μέσα ώστε στον τομέα του ξεπλήματος μαύρου χρήματος να υπάρξει μεγαλύτερη εναρμόνιση. Και πρέπει να δούμε το ερώτημα ότι ποια πλεονεκτήματα και ποια μειονεκτήματα υπάρχουν ε, εάν υπάρξει μία αρχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τελευταίο παράδειγμα της δικής μας δέσμευσης είναι τα συμπεράσματα του Συμβουλίου για τη βελτίωση των ε, οικονομικών ερευνών της 17 η Ιουνίου, πριν από μερικές εβδομάδε δηλαδή εγκρίθηκε. Αξιότιμες κυρίε και κύριοι, αγαπητοί βουλευτές, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να προχωρήσουμε περισσότερο και ουσιαστικά. Στις 7 Μαΐου η Κομισιόν ε, ψήφισε το σημερινό ε, πακέτο, μάλλον το, το παρουσίασε. Αφενός περιλαμβάνει το σχέδιο δράσης της Κομισιόν και αφετέρου πιο συγκεκριμένα συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις που θα πρέπει να ε, παρουσιαστούν για το πρώτο τρίμηνο του 2021. Εμείς χαιρετίζουμε αυτό το δέσμη μέτρων και προτείνουμε να ξαναβάλουμε στην ατζέντα του Συμβουλίου αυτό το σημαντικό θέμα. Να δούμε τα ε, θεμέλια της πρότασης της Κομισιόν, να, να τα συζητήσουμε, να τα σκεφτούμε και να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια ε, στην Κομισιόν ε, για να βρει περαιτέρω κατευθύνσει βάσει των προτάσεων του Συμβουλίου. Εμείς ελπίζουμε ότι αυτά τα συμπεράσματα της Κομισιόν για την επεξεργασία των προτάσεων που θέλει να παρουσιάσει του χρόνου θα μας βοηθήσουν ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα για την καταπολέμηση τη νομοποίηση των από δραστηριότητε και τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικό. Υπάρχει δηλαδή περιθώριο βολτίωση. Αξιότιμε κυρίε και κύριοι, και για την προετοιμασία αυτού του σημείου τη ημερησία διάταξη ε, απέκτησα διαβάζοντα την εντύπωση ότι εσεί, ο Ευρωβουλευτέ, ολόκληρο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξίσου έχουν συνείδηση του πόσο πιεστικό είναι το ζήτημα. Οπότε εύχομαι όλοι να δείξουμε πολιτική φιλοδοξία, ούτω ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα του ξεπλήματο μαύρου χρήματο όλο και πιο αποτελεσματικά. Περισσότερο αποτελεσματικά από ό,τι μέχρι στιγμή. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα το λόγο έχει ο Αντιπρόεδρος κ. Ντομπρόφσκης. Ε, ε, Πρόεδρε, Αξιότιμη Προεδρία, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ. Πρώτα απ' όλα, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε να σα παρουσιάσω την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμηση νομοποίηση εισόδων από παράνομε δραστηριότητε και την χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Θέλουμε μια συνολική αντιμετώπιση του θέματο αυτού για να προστατεύσουμε καλύτερα την οικονομία μα και τα οικονομικά συστήματα στο μέλλον. Αποτελεί μία από τι κύριε προτεραιότητέ μα και ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ στη δικιά σα στήριξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται απόλυτα ε, την άποψη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι δηλαδή πρέπει να δημιουργηθεί μια αποτελεσματική πολιτική για τον ε, τομέα αυτό, να βάλουμε όλα τα κομμάτια του παζλ μαζί και να φροντίσουμε ε, να έχουμε και τη συμμετοχή όλων των αρχών σε ευρωπαϊκό αλλά και εθνικό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης τον Μάιο προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο αυτό. Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο και πολύπλευρο με συγκεκριμένους κανόνες για τους επόμενους μήνες προκειμένου να ενισχυθεί η εποπτεία και η εφαρμογή των κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την καταπολέμηση του φαινομένου. Στόχος μας είναι να καλύψουμε ό,τι και να παραμένουν και να αρθούν κάθε αδύναμη κρίκη της αλυσίδας αυτής στους, στην εφαρμογή των κανόνων. Οποιαδήποτε επιχείρηση λοιπόν, οποιοδήποτε όργανο, οποιαδήποτε υποψία υπάρχει, ε, θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Γιατί όλες αυτές ε, οι δυνατότητες ε, που υπάρχουν σε διάφορα επίπεδα θέτουν σε κίνδυνο τα οικονομικά μας συστήματα. Κύριος στόχος μας λοιπόν είναι να διασφαλίσουμε ότι όλοι στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα τηρούν απόλυτα τους κανόνες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν κάνει ό,τι της αναλογεί και έχουμε ξεκινήσει πολλές διαδικασίες επί παραβάση έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι ενσωματώνεται η νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο και εφαρμόζονται και οι οδηγίες, οι 4 και οι 5 όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση της νομοποίησης χρήματος από παράνομες δραστηριότητες. Έχουμε λοιπόν τις οδηγίες αυτές Έχουμε ήδη προχωρήσει σε τρεις αιτιολογημένες γνώμες όσον αφορά το θέμα αυτό. Τέσσερις ε, επίσημες ε, κοινοποίησει για μη εφαρμογή των κανόνων και 17 άλλες ε, περιπτώσεις έχουμε, όπου επίσης έχουμε δραστηριοποιηθεί για την αντιμετώπιση του θέματος. Υπάρχει λοιπόν η οδηγία η οποία αναγνωρίζει και τις προσπάθειες που γίνονται από πολλές χώρες μέλη. Οι κανόνες πρέπει να είναι αποτελεσματικοί. Γι' αυτό και τον Μάιο αποφασίσαμε να στείλουμε συστάσεις προς 11 χώρες μέλη για το θέμα αυτό. Και η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει τώρα επιπλέον εξουσίες και αρμοδιότητες και ελπίζουμε να τις χρησιμοποιήσει πλήρως. Όσον αφορά τα επόμενα βήματα, Θέλω ένα εποπτικό σώμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα προβαίνει συστηματικά σε ελέγχους στις ίδιες τις χώρες μέλη, επιτόπου. Με ενισχυμένη, με ενισχυμένη επάδρωση. Πρέπει να καλύψουμε τις αδυναμίες που έχουμε. Και εδώ θα θίξω κάποια ε, συγκεκριμένα ζητήματα κλειδί. Για παράδειγμα, η περίπτωση online δραστηριοτήτων που οδηγούν στην νομοποίηση παράνομου χρήματος. Οι αρχές θα πρέπει να τα αντιμετωπίζουν αυτά. Γνωρίζουμε όμως συγχρόνως ότι οι κανόνες οι οποίοι εφαρμόζονται δεν βοηθούν πάντα τις επιχειρήσεις που δρούν νόμιμα, γιατί υπάρχουν συνέπειες στις επιχειρήσεις αυτές όταν τηρούν τους κανόνες αυτούς αυτές οι επιχειρήσεις ενώ οι ανταγωνιστές τους δεν το κάνουν. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξέρετε ότι συμφωνεί μαζί σας ότι οι εθνικοί επόπτες δεν μπορούν από μόνοι τους να ελέγχουν τα πράγματα. Αυτό έχει καταφανεί από τα πρόσφατα σκάνδαλα που είχαμε, όπου το βρώμικο χρήμα μετακινείται από τη μία χώρα μπορεί να φτάσει σε μια άλλη χώρα όπου υπάρχει πιο αδύναμη εποπτεία και ούτω καθεξής. Το βρώμικο χρήμα δεν θα πρέπει να μπορεί να κρύβεται πουθενά και γι' αυτό ακριβώς πρέπει να υπάρξει εποπτεία σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τέτοιο ευρωπαϊκό εποπτικό σώμα θα πρέπει να έχει εποπτικές δραστηριότητες σε περίπτωση που υπάρχουν ε, ε, οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή μη χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τα οποία μπορεί να κρίνονται ύποπτα για τέτοιες παράνομες δραστηριότητε. Θα πρέπει να υπάρχει και διαβούλευση και εμείς θα προτείνουμε μια νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία η οποία θα μπορεί να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Εξαρτάται βέβαια από το τι θα ακούσουμε και από τις δικές μας τι αξιολογήσεις. Θα δούμε πώς θα προσδιοριστεί αυτό. Πάντως η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα είναι ο ε, επόπτης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορεί να βοηθήσει τις αρχές και τις κυβερνήσεις. Θέλω όμως εδώ να είμαι ξεκάθαρο. Ένας ε, Ευρωπαίος επόπτης δεν μπορεί να εφαρμόσει τους κανόνες για την καταπολέμηση του φαινομένου αν σε εθνικό επίπεδο δεν υπάρχουν ε, οι αντίστοιχοι κανόνε προ τη σωστή κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα πρώτα απ' όλα να φροντίσουμε για την πρόληψη του φαινομένου και αυτό θα το στηρίξει και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και η Europol και η Eurojust. Επίσης ε, θα υπάρχει και καλύτερη προστασία για τους μάρτυρες δημοσίου συμφέροντος, τους καταγγέλλοντες με το κατάλληλο νομικό πλαίσιο. Δεύτερον, θα φροντίσουμε για ένα μηχανισμό που να ασχοληθεί και με την ροή, την κυκλοφορία και τη διαδρομή του βρώμικου χρήματος. Και να δούμε πού λαμβάνει η χώρα το φαινόμενο αυτό διασυνοριακά. Έπειτα, ε, το φαινόμενο δεν σταματάει στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε χρειάζονται αυστηροί κανόνες και σε τρίτες χώρες. Και δεν είναι όλες οι χώρες, οι τρίτες χώρες που έχουν αυστηρά καθεστώτα όσον αφορά αυτό το φαινόμενο. Έτσι λοιπόν μαζί με το σχέδιο δράσης που προσφέρει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τη δυνατότητα να αναλάβει δράση, υπάρχουν και οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με καταξιοδότηση πράξη με κατάλογο, ο οποίος πρόσφατα άρχισε να ισχύει, με τρίτες χώρες ασφαλείς ή μη ασφαλείς. Με δύο λόγια, πρέπει να πάμε προς δύο κατευθύνσεις. Η μη ασφαλης με Επιτροπή να ξέρετε ότι είναι έτοιμη να αναλάβει το ρόλο της, να προστατεύσει την εσωτερική αγορά και τα οικονομικά συστήματα από εγκληματίες. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πει ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε η συζήτηση αυτή να καταλήξει θετικά. Ξεκινάμε τη συζήτηση τώρα και πρώτος είναι ο κύριος Νταβιτ Κάσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ξέπλυμα χρήματος είναι κάτι που το χρειάζονται οι εγκληματίε. Έτσι δημιουργούν τα παράνομα κέρδη Οπότε εμεί θα πρέπει να είμαστε πιο στεγανοί και να του καταπολεμήσουμε, διότι δεν αρκεί να έχουμε ε, τη σχετική νομοθεσία. Θα πρέπει ε, ο νόμος να εφαρμόζεται. Και πολλές φορές έχουμε συμμορίες, μαθίες που έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τα δραστηριότητά του παρά το ότι υπάρχουν ξεκάθαρε αδράτε αποδείξει για το ξέβλημα. Υπάρχουν ε, λογιστέ, σύμβουλοι. Όλοι αυτοί επομένω τελικά ζουν σε ένα παράλληλο κόσμο και δεν γίνεται τίποτα από την νομοθεσία. Γιατί ε, οι θεσμοί δεν μπορούν να κάνουν την επαρκή έρευνα. Οπότε έχουμε ε, διαφθορά, έχουμε το ξέπλυμα και πάρα πολλοί ερευνητικοί ερευνητές δημοσιογράφοι όπως η Γαλίτσια έχουν ε, ψάξει το θέμα και μάλιστα η Γαλίτσια πληρώσει με τη ζωή της δεν είναι δυνατόν να τους αγνοήσουμε θα πρέπει αυτή οι κλιματίες να πληρώσουν Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Χέινε Λεώμα Έρο Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ομάδα των Σοσιαλδημοκρατών είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη που η Γερμανική Προεδρία αφοσιώνεται στα μέτρα για την καταπολύμψη του ξέπλυματος μαύρου χρήματος και χαιρόμαστε που ε, ε, δημιουργεί και τα κίνητρα η Κομισιόν. Σε αυτή την περίπτωση μιλάμε για τεράστια χρηματικά ποσά, σχεδόν 1% του ΑΕΠ ε, σε αυτό το παράνομο εμπόριο και τις παράνομες δράσεις θα πρέπει να γίνει κάτι λοιπόν γι' αυτό εμείς είμαστε ε, υπέρ δεσμευτικής νομοθεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φτάνει πια με τις οδηγίες. Έτσι λοιπόν υποστηρίζουμε να υπάρχει μια ε, ευρωπαϊκή αρχή. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή αρχή που να μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και να το καταπολεμήσει. Πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Θα πρέπει να δούμε κυρώσεις. Αυτό θα θέλαμε εμείς, πραγματικές κυρώσεις και να αναλάβει το, ο οικονομικός κόσμος και τις ευθύνες του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ ο κύριος Καρικάνο Λούις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Αντιπρόεδρε που σας ευχαριστούμε ε, για όσα μας εξηγήσατε οι εγκληματίες. Ε, ε, είναι 1% του ΑΕΠ, δηλαδή κερδίζουν 160 δις και, και 800 60 δις είναι η φοροδιαφυγή, αλλά και η απάντη για τον ΦΠΑ. Πρόκειται για ένα ξέπλυμα και μένει ατιμόρυτο. Πρόκειται για το 99% των όσων από εκεί κερδένουν έτσι αυτοί οι εγκληματίες που δεν δημεύονται, δεν κατάσχονται οπότε είναι ένα πρόβλημα αν θέλουμε να έχουμε μια πιο δίκαιη κοινωνία. Και πρόσφατα είχαμε κάποια γεγονότα για ποιες έρευνες, το Leaks, όπως είχαμε και την δολοφονία της Κορώνα Γαλήσια, ε, βλέπουμε ότι δεν γίνονται αρκετά ε, και επομένως ε, η Ευρώπη έχει μείνει πίσω σε αυτό το μέτωπο να είμαστε πιο φιλόδοξοι και θα πρέπει επομένως το ψήφισμα με, να εγκριθεί με ευρία πλειοψηφία και θα ήθελα πάντως να τονίσω τα εξής πέντε. Πρώτα πρώτα να υπάρχει μια εποπτεία που να είναι πρικοδοτημένη Επίσης να υπάρχει αυτή η υπηρεσία της οικονομικής αστυνομίας για φοροδιαφυγή, για αποφυγή και επίσης θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ε, αναβαθμιστεί σε αυτό το μέτωπο και επίσης να υπάρχει διευκόλυνση ε, έρευνα των τραπεζικών λογαριασμών και επίσης θα πρέπει να δούμε τι γίνεται όσον αφορά τις ιδιοκτησίες ότι είναι στην κυριότητα ε, κάποιων επιλήψιμων ατόμων οπότε θα πρέπει αυτό να το κάνουμε για να μην συνεχιστεί αυτή η ατιμωρησία των εγκληματικών κέντρων των Είχε Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνάδελφε, το λόγο έχει ο κύριος Μπέκ. Εκτός μικροφώνου ο κύριος ομιλητής, δυστυχώς δεν ακούμε. Το ξέπλυμα χρήματος είναι διεθνικό και έτσι πρέπει να είναι και τα μέτρα και οι κυρώσεις. Δεν πρέπει να ε, παραβλέπουμε και ένα άλλο είδος εξεπλήματος της ε, ΜΚΟ σε συνεργασία με εθνικές αρχές ε, που θεωρούν ότι η ΜΚΟ είναι ένας θαυμάσιος χώρος για εξεπλήμα χρήματος. Παρά αυτά είναι υπεράνω του νόμου με τους εμπειρογνώμονες που έχουν η Open Society Foundation με πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ επηρεάζουν μάλιστα και την κοινή γνώμη η Ουγγαρία προσπάθησε να καταγγείλει και να καταδικάσει τέτοιες ε, περιπτώσεις. Ε, αγαπητοί συναδελφοί, όταν θέλετε να μιλάτε για φοροδιαφυγή και για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, μην ξεχνάτε τις παλιές και καλές ε, δράσεις του φίλου σας Σόρος. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπρίκμον Σασκιά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το φιλόδοξο σχέδιο δράση για την καταπολέμηση τη νομοποίηση εσόδων από παράνομε δραστηριότητε και της χρηματοδότηση τη τρομοκρατία. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο ότι δεν υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνε, αλλά ότι δεν εφαρμόζονται αποτελεσματικά από τι χώρε μέλη. Γι' αυτό θα έπρεπε ήδη οι οδηγίε να προχωρήσουν και να γίνουν κανονισμοί και να υπάρξει ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας στην εθνική νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωράει σε διαδικασίες επί σε βάρος των χωρών μελών που δεν συμμορφώνονται. Είναι προτεραιότητα. Η κρίση, από ό,τι φαίνεται, προσέφερε νέες ευκαιρίες στους εγκληματίες. Και έτσι οι πολίτες, οι πιο ευάλωτοι είναι αυτοί που κινδυνεύουν. Εξάλλου, από ό,τι φαίνεται, το 98, του παράνομο αυτού χρήματος ε, δεν ανακτάται. Θα έπρεπε λοιπόν να φροντίσουμε να υπάρχει τέτοια ανάκτηση και να πηγαίνει στα πραγματικά θύματα του φαινομένου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το ξύπνο του βρώμικου χρήματο και η χρηματοδότηση τη ε, τρομοκρατία είναι οι δύο όψει ενό ε, πάρα πολύ ισχυρού επικίνδυνου αντιπάλου. Οπότε και γι' αυτό δεν θα πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε τέτοιε γκρίζε ζώνε και έχουμε δύο σημεία που θέλω να σα ε, αναδείξω. με ανησυχεί το ότι κάποιε πολιτικές πτέρυγες ε, θεωρούν ότι θα μπορούν να, ε, να ασπηλώσουν τις ε, τις ΜΚΟ μόνο και μόνο επειδή υποτίθεται ότι έχουν αυτή την πονημία χωρίς σκοπό το κέρδος. Οπότε θα πρέπει να υπάρχει έρευνα του πώς χρηματοδοτούνται και υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη στα οποία παράνομα υπάρχουν κάποιες ε, επιθετικές φορολογικές ε, πολιτικές και υπάρχουν πάρα πολλοί ε, χαλαρές νομοθεσίες. Οπότε έτσι υπάρχει μια προστασία στα τραπεζικά δεδομένα στην πράξη οι διεθνείς διοικητικές αρχές δεν μπορούν να ψάξουν αυτούς τους λογαριασμούς. Νομίζω ότι αυτό είναι απαράδεκτο και πρέπει συντόμως να διορθωθεί. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γκουσμάου Ζωζέ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμεί ζητήσαμε αυτή τη συζήτηση όχι μόνο εν συνεχεία τον Μονταλίξ και τη σπουδαιότητα αυτού του θέματο, αλλά και γιατί στη χώρα μου αυτός που κατήγγειλε ε, τον ε, κρατήθηκε για πάνω από ένα χρόνο χωρίς να υπάρχει πραγματικό κατακαρτήριο. Πολύ απλά διότι το κατήγγειλε και τώρα βρίσκεται υποκράτηση, η κράτηση και δεν έχει ακόμα δικαστεί. Ε, η χώρα μου έχει και αυτή ένα φορολογικό παράδεισο, τη Μαδέρα, που είναι μέρος όπου ξαπλάνεται χρήμα. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να καταλάβουμε, μας είναι τόσο δύσκολο σε αυτό το κοινοβούλιο, πολλές φορές λόγω πολιτικών φιλιών ή εθνικών φιλιών, διστάζουμε να θεσπίσουμε ή να καταγγείλουμε τις δικαιοδοσίε που διευκολύνουν την νομιμοποίηση εσόδων από δραστηριότητες δραστηριότητε Ζητάω λοιπόν από την Κομισιόν να δείξει κάποιο θάρρο ε, για το ξέπλυμα μαύρου χρήματο. Του το ζητάμε αυτό, αλλά αυτό πρέπει να ξεκινάει και από εμά του ίδιου, το Κοινοβούλιο. Φυσικά πρέπει να καταλάβουμε ότι ναι, πράγματι υπάρχουν ε, ε, τρίτε χώρε υψηλού κινδύνου, αλλά όλε οι χώρε υψηλού κινδύνου δεν είναι τρίτε χώρε, πολλέ είναι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χρειάζεται συνεργασία και να αλλάξουμε επίση και τι εθνικέ νομοθεσίε. Υπάρχουν πολλέ πτυχέ αυτή τη νομοθεσία πολύ σημαντικέ το τέλος των χρυσών θεωρήσεων, η προστασία των ε, καταγγελτών, ε, το One είναι πολύ μεγάλο παράδειγμα, η κατονομασία των εγκληματιών και η κατάσχεση, η δίμευση των προϊόντων του εγκλήματος. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Κολάκουσης Μισλάβ. Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς διαπιστώνουμε ότι αποτελούμε μία κατηγορία που είναι χειρότερη γιατί υποφελούμε από την πανδημία. Και μερικές φορές διαπιστώνουμε ότι μέσα σε μία μέρα κάποιοι πλουτίζουν κατά πολλά δισεκατομμύρια και 26 στον κόσμο αυτό έχουν την ίδια περιουσία όσο έχουν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο. Αυτοί λοιπόν που υποφελούνται βασίζονται σε διάφορες εκστρατείας εκφοβισμού, διάδοσης του φόβου και τελικά εποφελούνται αυτοί που έτσι αλλιώς έχουν μεγάλη περιουσία και μπορούν να αγοράσουν ολόκληρες επιχειρήσεις στη μισή τιμή από την αξία τους. Πρέπει λοιπόν να υποληθεύσουμε σήμερα ποιος τελικά χρηματοδοτεί τι στα μέσα ενημέρωσης. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Μόνικα Χόλμα έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε ε, Επίτροπε, αγαπητή Προεδρία της Γερμανίας. Βλέπω με, δυστυχία, λύπη ότι εδώ και χρόνια από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, υπάρχει έτσι μια φιλική στάση προς τα κράτη-μέλη που έχουν συνηθίσει να μην εφαρμόζουν ε, τις κατευθυντήρες γράμμες ε, και τις οδηγίες για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος η 3 ε, φαίνεται να μην εφαρμόστηκε ε, παρκώς την 4 την εφάρμοσαν κάποια μόνο κράτη-μέλη έχουν μείνει πίσω και στα πρότυπα σε σχέση με το τι προβλέπεται στις οδηγίες και στην οδηγία 5 πολλοί δεν έχουν ε, κάνει καμία μεταφορά και μεγάλο μέρος των υπολείπων δεν δηλώνει να έχει ε, ε, μεταφέρει την οδηγία ή να την έχει εφαρμόσει ούτε τα μισά κράτη-μέλη πρέπει να ακολουθήσουμε πιο αυστηρή στάση χρειάζεται ε, διαφάνεια καθαρά λόγια και στις έρευνες των αρχών σε οικονομικά τέτοια θέματα να μπορούμε να βρούμε δηλαδή δίκτυα τα οποία μπορούμε να βρούμε μόνο αν υπάρχει σωστή εφαρμογή των μέτρων σας παρακαλώ από βάθος καρδίας ε, αγαπητή Επιτροπή ε, κάντε τα πράγματα λίγο και με μεγαλύτερη αυστηρότητα μην αφήνετε τα κράτη-μέλη έτσι Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τάγκα um, Πρόεδρε ευχαριστώ πολύ Το ξέπλυμα χρήματος είναι τεράστιο, είναι κατ' εκατομμύρια, είναι χρήματα τα οποία κλέβονται, είναι παράνομα και πλήττονται πάρα πολλοί κόσμος και κυβερνήσεις και είναι χρήμα το οποίο στη συνέχεια ξοδεύεται χάρη στο απόρριτο που έχουμε και είναι άγνωστοι αυτοί που κατέχουν αυτό το παράνομο χρήμα και όμως πρέπει να μπορούν να διώκονται να φτάνουν στη δικαιοσύνη και να τιμωρούνται και είναι τροπή που δεν έχουν εφαρμόσει όλες οι χώρες μέλη την τελευταία οδηγία και δεν υπάρχει μητρό και το αποτέλεσμα είναι ότι 96 δισεκατομμύρια ρωσικού χρήματος που έχει επενδυθεί στην Ολλανδία ε, είναι με άγνωστο επενδυτή. Ναι, θέλουμε εναρμόνιση και θέλω να ενθαρρύνω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις χώρες μέλη να συνεχίσουν να αγωνίζονται υπέρ της δικαιοσύνης. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ρωμανά Στρουγκαρίου. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, παγκοσμίω, σε ένα χρόνο, έχουμε 2-5% του παγκοσμίου που είναι το ξέπλυμα. 800 δις, ένα Αμερικανικών δολαρίων. Η καταπολέμηση αυτών και των φορολογικών παραδείσων προστατεύει τις οικονομίες, σώζει ζωές, έχει επιπτώσεις στις κοινωνίες που θίγονται από το οργανωμένο έγκλημα. Να έχουμε αυτή την εποπτική αρχή και την οικονομική ευρωπαϊκή αστυνομία. Να έχουμε επίσης κάποια μητρώα των αληθών δικαιούχων. Μπράβο στην Κομισιόν για το πρόγραμμα δράσης. Όμως ξέρουμε ότι τα κράτη-μέλη δεν τα καταφέρνουν να μεταφέρουν στη νομοθεσία να τα έχουν καταφέρει να, την, να το κάνουν για αυτές τις ε, οδηγίες. Άρα χρειάζεται συντονισμός και θα πρέπει οι προτεραιότητες να γίνουν νομοθεσία και να γίνεται ουσιαστική εποπτεία της ε, εφαρμογής και των αποτελεσμάτων και κάτι τελευταίο. Για να το σκεφτούμε καλύτερα και να τα πούμε καλύτερα στα κείμενα μας. Ας δούμε και στο δικό μας περιβόλι τι γίνεται γιατί και εμείς έχουμε θέματα απορρίτου, φοροδιαφυγές και τα σχετικά. Είναι 27 δις τα φορολογικά έσοδα που ε, με κάποια φοροτεχνικά κόλπα δεν τα εισπράττει το κράτος. Άρα εδώ και τώρα κάνουμε κάτι σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Έρβεζουβάν. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, φυσικά όλοι είμαστε κατά της νομοποίησης εσόδων απαράνομης δραστηριότητε και της χρηματοδότησης της τριμοκρατίας. Τι κάνουμε όμως με συστήματα τα οποία επιτρέπουν τέτοιες δραστηριότητες χωρίς να γνωρίζουμε τελικά ποιος είναι ο τελικός δικαιούχος. Χρειάζεται γρήγορα ε, μια ρύθμιση για το ηλεκτρονικό χρήμα που μπορεί να κυκλοφορεί χωρίς να ξέρουμε ποιος είναι ο δικαιούχος. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση τη τρομοκρατία, θυμάμαι τι είπε ο Νιγεριανός Υπουργός Άμυνας στη διάσκεψη του Ντακάρ, ο οποίο είπε ότι δεν πρέπει να έχουμε ψευδεστήσει. Ξέρουμε ποιε χώρε χρηματοδοτούν την τρομοκρατία. Κάποιε από αυτέ είναι καλοί πελάτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιε από αυτέ τι χώρε είναι σύμμαχοι ή και εταίροι ακόμα στο ΝΑΤΟ και έφτασε και σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγώ φαντάζομαι εδώ πέρα ε, Βαλκάνια ή Συρία, που χρηματοδοτείται εκεί η τρομοκρατία. Η διαφορά θα γίνει αν ενισχυθούν οι αστυνομικές και υποπτικές αρχές. Ευχαριστούμε συνάδελφος κ. Βεν Κίγκολτ. Κύριε Υφυπουργέ Ρότ, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή έχει σοβαρές ε, προτάσεις ε, για το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για την καταπολέμηση της καταπολέμησης ε, του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και απαιτείται και η υποστήριξη του Κοινοβουλίου κοινή οπτική κοινή ισχυρότεροι κανόνες αλλά και πιο αποτελεσματική οικονομική αστυνομία που να λειτουργεί διασυνοριακά δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στην παραβίαση όμως ε, κάποιων νόμων. Μην έχουμε την ε, αυταπάτη ότι το παλιό δίκαιο που είναι 13 ετών από την ε, οδηγία 3 παραβιάζεται σε πολλές χώρες και στη Γερμανία και εκεί δεν υπάρχει καμία διαδικασία επί παραβάση. Οπότε απευθύνω έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Αυτό το δίκαιο που υπάρχει ήδη, ήδη ε, θα πρέπει εκεί να ακολουθείτε κάποια ε, διαδικασία επί παραβάση όταν πραγματικά γίνεται ξέπλεμα μαύρου χρήματο, όχι μόνο όταν υπάρχει μια απλή παραβίαση. Αυτό δεν έχει κάνει ακόμα η Κομισιόν. Θέλουμε περισσότερη πίεση, περισσότερη ταχύτητα, κύριε Επιτρόπε. Ευχαριστούμε. Η κυρία Λαούρα Φεράρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτό το ξέπλυμα και χρηματοδότηση τη τρομοκρατίας θα πρέπει να γίνει στρατηγική πρόκληση για την ε, Ένωση. Δεν είναι δυνατόν ε, να μην λαμβάνει υπόψη τι γίνεται με τη διαφθορά, το λαθρεμπόριο όπλων, δηλαδή το δουλεμπόριο, την φοροδιαφυγή. Οπότε ε, θα πρέπει να δούμε ότι χρειάζεται περισσότερη εποπτεία γιατί βλέπουμε πως οι εγκληματίες ε, μολύνουν τις οικονομίες μας και ε, αυτό για ακόμα χειρότερα τώρα με την πανδημία. Θα, δεν θα πρέπει να έχουμε απόκληση νομοθεσιών και παρερμηνίες ή διαφορετικές ερμηνείες του κοινοτικού δικαίου να μην ωφελούνται αυτοί ε, τους φορολογικούς παραδείσους γιατί έτσι ε, στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό, υπονομεύουν την ενιαία αγορά, θα πρέπει να στραφούμε πλήρως σε αυτό το μέτωπο, εναρμόνιση, να δούμε πού υπάρχουν οι μεγαλύτεροι κίνδυση, να υπάρχει επίσης ε, ε, γνωστοποίηση των πληροφόρων που υπαρχουν οι μεγαλύτερη κινδυση να υπαρχει επισης γνωστοποιηση των πληροφορων που εχουμε και να υπάρχει ανείγνευση των ε, ροών του χρήματος για να εντοπίσουμε τις μαφίες. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρκους Φέρμπερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επιτρόπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το ξέπλυμα μαύρου χρήματος τα τελευταία χρόνια δείχνει ότι είναι πολύ απλό. Τελικά υπάρχουν δύο σημαντικά προβλήματα. Πρώτον, η εφαρμογή και η μεταφορά του δικαίου όπως υπόθηκε ήδη. Κύριε Επιτρόπε, την περασμένη εβδομάδα για τρία κράτη-μέλη ξεκίνησε μια διαδικασία παραβάση για παράβαση τη τέταρτη οδηγία. Για την πέμπτη δεν θα μιλήσω καν. Πώ είναι η κατάσταση τη εφαρμογή. Και παρόλα αυτά, και δεύτερον, υπάρχει μια οδηγία που σημαίνει ότι ουσιαστικά έχουμε κάτι τελείω ρευστό. Ε, η εφαρμογή γίνεται τελείω διαφορετικά από το κάθε κράτος. Και το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο θα ήθελα να πω καθαρά εδώ, είναι ότι φυσικά ότι η επικοινωνία μεταξύ αρχών δεν λειτουργεί καθόλου. Το ζούμε στη Γερμανία επίσης ότι η αρχή επιτήρηση, οι αρχέ ερευνών έχουν δυσκολίε για να το πω ε, με ε, ήπια λόγια να συνεργαστούν. Πρέπει να εντοπίσουμε αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε και τις προτάσεις της Κομισιόν να υπάρχει μια κεντρική αρχή με ε, ε δικαιώματα έρευνας. Αλλιώς κάθε χρονιά θα κάνουμε τις ίδιες συζητήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μετά από τον συντονιστή του Έλκέ έρχεται ο συντονιστή των Σοσιαλιστών, ο κ. Φερνάνδε Γιώνα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Στη συζήτηση αυτή για την αντιμετώπιση της παράνομης κυκλοφορίας κεφαλαίου συζητάμε για την καταπολέμηση των ε, οικονομικών παραδείσεων αλλά είναι πράγματα ε, για τα οποία υπάρχει συνένεση. Συμβούλιο, Επιτροπή, Κοινοβούλιο και μας στηρίζει φυσικά και Ευρωπαίος πολίτης γιατί Όλοι εμεί θεωρούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιε αδυναμίε, τέτοια κενά στα νομικά μα συστήματα. Αλλά από τη μια υπάρχει αυτή η συνένεση, από την άλλη μεριά όμω δεν είμαστε σε θέση να υιοθετήσουμε νέε πρωτοβουλίε, να ε, εφαρμόζουμε τα όσα έχουμε αποφασίσει, να ελέγχουμε την κατάσταση στι χώρε μέλη και έτσι να συνεισφέρουμε και να βοηθήσουμε τον Ευρωπαίο πολίτη. Νομίζω ότι ήρθε η στιγμή όχι να αναλύουμε πώ ε, ενσωματώνονται οι οδηγίε, αλλά να υπάρχουν κανονισμοί σε αυτό το τομέα. Ένας κανονισμός πρέπει να ελέγχεται από έναν επόπτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μην υπάρχουν περιθώρια παρανομιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Ερμαν Χάιντερ. Η καταπολέμηση του ξεπλήματο μαύρου χρήματο και τη χρηματοδότηση τρομοκρατίας τρομοκρατία είναι μια απέτηση ανεξαρτήτω πολιτικών ιδεολογιών οι πολιτικών ομάδων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι πρέπει να την υποστηρίξουν με την ίδια δέσμευση. Τουλάχιστον έτσι θα έλεγε κανεί θεωρητικά. Όταν βλέπω όμω το σχέδιο δράση τη Κομισιόν για την καταπολέμηση του ξεπλήματο μαύρου χρήματο και τη χρηματοδότηση τρομοκρατία και γνωρίζοντα ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απαιτεί διαφάνεια από τα κράτη-μέλη για διάφορες κρατικές οργανώσεις, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Η κατάσταση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις κάνει μεγάλη εντύπωση. Δίνεται εντύπωση ότι αυτές οι δραστηριότητες ε, των οργανώσεων αυτών είναι νόμιμες και όποιος έχει ασχοληθεί με το θέμα έχει ανακαλύψει ότι είναι επικίνδυνες αυτές οι οργανώσεις όσον αφορά το ξέπλυμα μαύρου χρώματος παρότι ε, το Ισλαμικό κράτος και άλλοι τέτοιοι ε, οργανισμοί και άλλες τέτοιες οργανώσεις χρησιμοποιούν το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οπότε η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, ρηψοκινδυνεύουν έτσι την ασφάλεια των πολιτών. Ευχαριστούμε. Η κυρία Περέρα, παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για μας το να τους καταπολεμήσουμε αυτού από την Έχουμε 160 ε, δις που χάνονται. Υπάρχει ε, η έκθεση Γεροπόλου που λέει ότι τα πράγματα ε, επίγουν. Αυτό το ξέπλυμα χρήματο είναι ένα έγκλημα περίπλοκο. Είναι στο επίγεντρο πολλές άλλες εγκληματικές μορφές. Ε, χρηματοδότηση του, του, της τρομοκρατίας, φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή. Επομένως, το θέμα δεν είναι μόνο αυτά τα οικονομικά εγκλήματα. Είναι και θέμα ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων και κράτους δικαίου. Χρειάζεται συνεργασία, εναρμόνιση των δικαίων και χρειάζονται κάποιες δομές αποτελεσματικές. Υπάρχει κατάτμιση της νομοθεσίας, ε, οπότε θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι ευκαιρία για τους εγκληματίες. Χρειάζεται μια πραγματικά ευρωπαϊκή στρατηγική. Μόνο με περισσότερη Ευρώπη θα πετύχουμε λιγότερη εγκληματικότητα. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Αγγιλάρ. 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ πηγαίνει σε ύποπτες οικονομικές δραστηριότητες, στην διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα. Οπότε φυσικά και στηρίζω απόλυτα το σχέδιο δράση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με πρώτο στόχο την εφαρμογή τη πέμπτη οδηγία, η οποία πρέπει να ισχύει, όχι μόνο να ενσωματώνεται στην εθνική νομοθεσία, αλλά να εφαρμόζεται κιόλα. Και έπειτα υπάρχει το θέμα τη εποπτείας, ενιαία εποπτείας, ώστε όλε οι μονάδε χρηματοοικονομικών πληροφοριών να συνδέονται μεταξύ του και να αλληλοενημαρώνονται και να περάσουμε από την οδηγία στον κανονισμό Έπειτα, διεθνή συνεργασία. Όντως πρέπει να ενισχυθεί σε ένα τέτοιο προβληματικό ζήτημα. Επίσης, κατάρτιση και εγγύηση ότι θα μπορούν να εντοπίζονται οι τελικοί δικαιούχοι του χρήματος αυτού που ξεπλένεται. Μόνο τότε θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο Πράγματι, η Επιτροπή ζητάει να εφαρμοστεί η πέμπτη οδηγία από τις χώρες μέλη. Ελπίζω να το κάνουν. Ευχαριστούμε η κυρία Γκιωρή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι χρειάζεται να καταπολεμήσουμε το ξέβλημα χρήματο αλλά και τη χρηματοδότηση τη τριμοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν να επιτρέψουμε στι εγκληματικέ οργανώσει να συνεχίσουν αυτή του την διασυνορική δραστηριότητα, αλλά το ερώτημα είναι πώ θα γίνει αυτό καλύτερα. Στο παρελθόν έχουμε περάσει ένα σωρό νομοθετήματα και πολλέ φορέ ε, είδαμε ότι αυτά δεν εφαρμόστηκαν όσο επιτοπλίστων, αλλά δεν ξέραμε επίση τι να κάνουμε στην πράξη με αυτά τα νομοθετήματα. Είχαμε και ένα σωρό σκάνδαλα και επομένως γι' αυτό σας λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ούτως ώστε να υπάρξει πραγματικά η Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή. Ε, όμως να προσέξουμε διότι έτσι παραβιάζουμε την αρχή της επικουρικότητας, έτσι συρρυκνώνουμε τις εθνικές αρμοδιότητες. Θέλει το Κοινοβούλιο να κάνει βήματα προς τα εμπρός, αλλά ε, θα πρέπει να τα σκεφτούμε καλύτερα, καλύτερα για να πετύχουμε περισσότερα σε αυτό το μέτωπο και παρά τις ε, επιφυλάξεις μου εγώ θα ψηφίσω υπέρ αυτού του κειμένου. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ολοκληρωθήκε η συζήτηση, οπότε θα ακολουθήσει το Συμβούλιο και η Κομισιόν δίνουμε το λόγο στον Αντιπρόεδρο uh, τον Πρόσκης. Τον Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριοι βουλευτές από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστούμε το Κοινοβούλιο διότι μας δώσε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και εμείς έτσι να εμπλουτίσουμε το πλωστάσιό μας κατά ε, της ε, χρηματοδότησης τρομοκρατίας, ξεπλήματος ε, παρανομού χρήματος και άρα θα πρέπει να βαθύνουμε τις προσπαθειές μας και να είναι πιο αποτελεσματική η Ευρωπαϊκή Ένωση και να σταματήσει έτσι αυτή η υπονόμευση του χρηματοοικονομικού συστήματο, Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, αναφέρατε πολλά κατά αυτή την ε, συζήτηση και είπατε για το πώς θα εφαρμοστούν οι ισχύουσες διατάξεις θα πρέπει να είμαστε υποτελεσματικοί όντως γιατί έτσι θα πρέπει να δούμε πώς θα γίνουν εθνικό δίκαιο οι κοινοτικές ε, οδηγίες. Αυτό θέλει και η Κομισιόν. Θέλουμε κατηγορηματικά Θέλουμε να είμαστε αυστηροί με τα κρατημέλη για να κάνουν τα κρατημέλη αυτήν την μεταφορά στο εστρικό δίκαιο και αυτό θα πρέπει να κάνουμε ε, στο μέλλον. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε κανονισμούς, όχι οδηγίες. Ε, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έτσι η νομοθεσία θα είναι πιο αποτελεσματική σε ευρωπαϊκό επίπεδο γιατί χρειάζεται και εποπτεία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μπράβο που συμφωνήσατε πολλοί από εσά, συνάδελφοι. Και υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο το είπαν μια σειρά συναδέλφων όσον αφορά την ε, φορολογία. Όντω η καταπολέμηση φοροδιαφυγή, φοροαποφυγή, αυτό είναι κάτι που χέρι-χέρι πρέπει να αντιμετωπιστεί το οποίο που είναι παράλληλη δραστηριότητα δηλαδή με το ξύλινο χρήματο. Δηλαδή, εμεί γι' αυτό παρουσιάσαμε κάποια μέτρα, ούτω ώστε να έχουμε πιο στεγανό νομοθετικό πλαίσιο για αυτά τα φαινόμενα. Έχουμε μια ολόκληρη δέσμη μέτρων. Θα σας τα παρουσιάσουμε τα όσα προτείνουμε την επόμενη εβδομάδα. Και έχουμε στο οπλοστάσιό μας το πώς θα ελεγχθούν οι πάροχοι υπηρεσιών. Πάντως, εμείς θα μείνουμε σταθεροί στη δέσμευσή μας για αυτή μας την προσπάθεια και σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας και ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μιχάλ έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρο, αξιότιμες κυρίες και κύριοι, κύριοι βουλευτές. Πρώτα απ' όλα χαίρομαι που κάναμε αυτή τη συζήτηση ε, καταπολέμηση του ξεπλήματος μαύρου χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας πρέπει να γίνει πιο διεξοδικά. Συμφωνούμε όλοι με αυτό. Χρειαζόμαστε περισσότερη διαφάνεια, περισσότερους κανονισμούς ε, και περισσότερους ελέγχους. Πιστεύω αξίζει το κόπο να ελέγξουμε κάθε πρόταση που έχουμε επιτάπητος ε, και να βελτιώσουμε την εφαρμογή. Χαίρομαι που ανέφεραν ε, οι ευρωβουλευτές την οικονομική διάσταση της ε, νομιμοποίησης εσόδων από παρανομιες δραστηριότητες. Ε, το 1% του ΑΕΠ μιλάμε για 8% φορολογικές απώλειες. Θέλω να πω μια ιδέα εδώ, δεν ξέρω αν συνηθίζεται. αλλά θα ήθελα να πω ότι χρειαζόμαστε μια κοινωνία των πολιτών ε, η οποία να μας βοηθήσει σε αυτή τη δημοκρατική ε, δράση. Ε, αυτό αναφέρεται και στις ζωντανές μας δημοκρατίες από τις ενώσεις των νέων και από την κοινωνία των πολιτών. Ε, Κριτικέ λοιπόν μη κυβερνητικές οργανώσεις που δεν αρέσουν σε ορισμένου ευρωβουλευτέ πρέπει να κάνουν κάτι. Ε, γιατί τι κατηγορούν για ε, χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή για νομοποίηση εσόδων ή παράνομες δραστηριότητες και δεν έχουν να κάνουν με όλα αυτά που τις κατηγορούν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία για τις τροπολογίες θα λάβει χώρα αύριο και η τελική ψηφοφορία την Παρασκευή. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ε, οι δηλώσει του Συμβουλίου και της Επιτροπής ε, για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας για την εποχή μετά από την πανδημία COVID-19. Θα ήθελα για άλλη μια φορά να ενημερώσω τα μέλη ότι σε αυτή τη συζήτηση δεν θα δεχθούμε μπλε κάρτες ούτε ε, αυθόρμητες ε, αιτήσει για χρονογόρευση. οπότε ας ξαναδώσουμε το λόγο στον κύριο Μίχαλ Ρότ εκ μέρους της ε, του Συμβουλίου. Αξιότιμες κυρίες και κύριοι βουλευτές, αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, Έχουμε να κάνουμε με μια κατάσταση ιδιαίτερη όσον αφορά την υγεία που επηρεάζει σημαντικά τις κοινωνίες μας, τους λαούς μας. Τέτοιες στιγμές ε, σκεφτόμαστε τους πάνω από 100.000 Ευρωπαίους και Ευρωπαίες που μέχρι στιγμής έχασαν τη ζωή τους λόγω του ιού COVID-19. τέτοιες εβδομάδες ε, συζητάμε πολύ εντατικά για το τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και να μάθουμε από αυτή τη δύσκολη κρίση για τις ε, υγειονομικέ μας υπηρεσίες, για το συντονισμό εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο μιας πιο αποτελεσματικής και πιο προληπτικής αν αντιμετώπισης ε, των πανδημιών και συζητάμε επίσης και για τα μαζικές κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες το είπε καθαρά και η καγκελάριο σήμερα το πρωί ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα σημεία τη Γερμανικής Προεδρίας. Και είμαι βέβαιος ότι όλοι και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συμμεριζόμαστε αυτή την δέσμευση να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το συντομότερο δυνατόν, όσο το δυνατόν πιο αλληλέγγυα και όσο το δυνατόν πιο ε, ομόφωνα να βγούμε από αυτή την κρίση. Ε, εγώ υποστηρίζω ε, αυτή τη θέση και θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδία τους ε, ανθρώπους που εργάζονται στο τομέα της νοσηλείας που σε τόσο δύσκολες εποχές έκαναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να προστατεύσουν ανθρώπους, για να υπηρετήσουν και να τους ασθενείς με τον καλύτερο δυνατό βαθμό και η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας χρειάζεται ε, συγκεκριμένη οργάνωση και πρέπει να το πούμε ειλικρινά κυρίες ε, και κύριοι. Πρέπει να πούμε καθαρά τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί. Και ειδικότερα όσον αφορά την αρχή της καταπολέμησης της πανδημίας, ποια, ποιες ήταν οι αδυναμίες που αναδείχθηκαν. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε στο μέλλον να αντιμετωπίζουμε πιο καλά, πιο γρήγορα και πιο ολοκληρωμένα άλλες κρίσεις. Και όλοι ξέρουμε ότι αυτή η κρίση δεν έχει περάσει ακόμα. Εξακολουθούμε να βρισκόμαστε σε μια πολύ αβέβαιη κατάσταση σε ορισμένες χώρες. Χάρη στην αφοσιωμένη προσέγγιση φαίνεται να έχει περιοριστεί πολύ η κρίση της πανδημίας αλλά και στην Ευρώπη και στην άμεση γειτονία μας ε, βλέπουμε ότι δεν είναι τίποτα ακόμα βέβαιο. Οπότε πρέπει να είμαστε σε επιφυλακή και σε ελεύθερες δημοκρατίες όπως οι δικές μας πρέπει ε, να δείξουμε αφοσίωση και στους λαούς ε, και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα κρατημέλη πρέπει να συζητήσουμε εντατικά για το πώς μπορούμε να προστατεύσουμε καλύτερα την υγεία των πολιτών μας χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας με δυσανάλογο τρόπο. Για αυτούς τους λόγους στόχος της Προεδρίας μας είναι να καταλήξουμε σε συμπεράσματα που αφορούν τα διδάγματα που αποκομίσαμε από την κρίση του COVID-19 και να καταλήξουμε σε ε, εύχριστα ε, συμπεράσματα για μελλοντικά μέτρα. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το τεράστιο ενδιαφέρον και την αφοσίωση που δείξατε όλοι για αυτό το θέμα. Σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο στην Ευρώπη, η πανδημία συνεχίζει να επιταχύνει την ε, διαδοσή της καθημερινά. Έχουμε σχεδόν 200.000 νέα κρούσματα και γνωρίζουμε όλοι ότι προφανώς πρόκειται για μια παγκόσμια κρίση ε, τέτοια έκταση η οποία απαιτεί, όπως είναι φυσικό, παγκόσμιες απαντήσεις. Καμία χώρα, όσο καλό σύστημα υγείας και αν έχει, δεν είναι σε θέση μόνη της να καταπολεμήσει αυτή την πανδημία. Οπότε καθιστάται σαφές ότι η πολιτική του εθνικού αποκλεισμού, ε, του επιμέρους κράτους, ε, ε, μια πολιτική που αποδυναμώνει την Ευρωπαϊκή Ένωση, συνεπάγεται απαράδεκτες κινδύνους για τους πολίτες μας. Έχουμε θλιβερές περιπτώσεις κυρίες και κύριοι οι οποίες όμως μας δίνουν μεγαλύτερη αισιοδοξία για την αλληλεγγύη, για την κοινή απάντηση που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από όπως έχουμε κάνει και στο παρελθόν για να ξεπεράσουμε αυτή την πανδημία. Αυτό σημαίνει πολλή δουλειά μπροστά μας. Η οικονομική κρίση ε, θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο αν ε, μακροπρόθεσμα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τον ιό. Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί βουλευτές, μια ε, ολοκληρωμένη στρατηγική για την καταπολέμηση της πανδημίας για την Ευρώπη και για ολόκληρο τον κόσμο φυσικά απαιτεί την ανάπτυξη ε, ασφαλών ε, εμβολίων και θεραπείων και ίση πρόσβαση σε όλα αυτά όλων. Η πανδημία θα αντιμετωπιστεί μόνο αν εξαλειφθεί παντού. Μία μακροχρόνια λύση ε, μπορεί να βρεθεί μόνο στο πλαίσιο της επιστήμης και της αλληλεγγύης. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να ερευνήσει και να χρησιμοποιήσει από κοινού ε, τα πιθανά εμβόλια που θα εμφανιστούν για το COVID-19 να, το να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν όλοι αυτό το εμβόλιο. Χρειαζόμαστε ένα εμβόλιο για την Ευρώπη αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο εδώ δεν μπορούμε να στρεφόμαστε ο ένας κατά του άλλου. Πρέπει όλοι να σταθούμε ένα στο πλευρό του άλλου. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να προστατεύσουμε την υγεία των ανθρώπων ανεξαρτήτως του που ζουν στην Ευρώπη ή οπουδήποτε στον κόσμο. Χαίρομαι ιδιαίτερα που η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους διεθνείς της εταίρους έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας ένα τεράστιο ποσό των 16 δισεκατομμυρίων ευρώ έτσι ήταν η κατάσταση της 30 Ιουνίου. Ε, συγκεντρώθηκαν αυτά για την ανάπτυξη, για την παραγωγή και τη διάθεση ε, εμβολίων ε, του COVID-19 για να επιταχυνθεί αυτή η παραγωγή. Έχουμε και άλλες δράσεις μπροστά μας. Χρειαζόμαστε λοιπόν ασφαλή αποτελεσματικά εμβόλια, χρειαζόμαστε μαζική παραγωγή ούτω ώστε όλοι οι άνθρωποι να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αυτά. Επ' θα ήθελα να συγχαρώ για την πρόσφατη νομοθεσία της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία επιταχύνει την διεξαγωγή κλινικών μελετών για εμβόλια για τον COVID-19 και ε, σχετικές θεραπείες και θέλω να ευχαριστήσω και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την απόφαση που έλαβε ακριβώς σήμερα ε, να λάβει θέση για αυτό το θέμα και χαίρομαι και συμμερίζομαι ε, και συμφωνώ ναι. που θα ψηφιστεί ε, για το, το φάκελο ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί βουλευτές, η μελλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στον τομέα της δημόσιας υγείας θα εντάσσεται στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο τη Κομισιόν και υπάρχει ένα φιλόδοξο πακέτο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το EU for Health, το οποίο προτάθηκε, όπου καθίσταται σαφέ ότι η υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ύψιστη προτεραιότητα και ότι θα πρέπει να είμαστε πιο καλά έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε μελλοντικέ ε, κρίσει υγείας. Αξιότιμοι βουλευτές, χρειαζόμαστε μια ποιοτική, υψηλής αξίας και αποτελεσματική δημόσια υγεία για να προστατεύουμε τους ε, λαούς μας από τέτοιες πανδημίες. Και γι' αυτό στο Συμβούλιο δίνουμε ύψιστη προτεραιότητα σε αυτό το θέμα και ελπίζουμε με τη δική σας υποστήριξη να το έχουμε αποφασίσει και να το έχουμε συμφωνήσει μέχρι τα τέλη του έτους. Ελπίζουμε να έχουμε μια στενή, γεμάτη εμπιστοσύνη συνεργασία για αυτή την πολύ σημαντική πρόταση. Επίσης, ε, καθοριστικό θα είναι να έχουμε τη διάθεση φαρμάκων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και άλλων αγαθών ε, που χρειάζονται στην Ευρώπη και πρέπει να βελτιωθεί η διάθεση όλων αυτών. Ξέρετε ότι στην αρχή της κρίσης, όταν ξεκίνησε η κατάσταση δεν ήταν ιδανική, αλλά πιστεύω ότι ως Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τα κράτη-μέλη ε, έχουμε καταλάβει ακριβώς τι έγινε και έχουμε εξάγει τα σχετικά συμπεράσματα. Η πανδημία του COVID-19 επέτεινε το πρόβλημα που έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων, φαρμάκων και ε, πρώτων υλών εξαρτάται από τρίτες χώρες. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε μόνο την παγκοσμιοποίηση. Αυτό που πρέπει να γίνει ότι για τόσο σημαντικά αγαθά που σχετίζονται με την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμείς θα πρέπει να μπορούμε να τα βρίσκουμε με τις δικές μας δυνάμεις να παράγονται εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ευρωπαϊκή αυτοδυναμία και αυτοκυριαρχία. Επίσης πρέπει να είμαστε σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίζουμε τέτοιες κρίσεις, να συγκεντρώνουμε πληροφορίες, να μπορούμε να ε, προβαίνουμε σε αξιολογήσεις και να δράμε ε, γρήγορα. Η στενή συνεργασία είναι λοιπόν αναγκαία ε, και μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των οργανισμών και των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Έργου Πρόληψης και Ελέγχου των Ασθενειών και της Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων όπως και με τους διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκοσμίος Οργανισμός Υγείας. Ένας από τους στόχους μας είναι ο τρόπος εργασίας αυτών των ευρωπαϊκών οργανισμών να ενισχυθεί και να επεκταθεί. Το πρόγραμμα EU for Health λοιπόν ε, ως προτεραιότητα θα ασχοληθεί με τα διδάγματα που αποκομίσαμε από την πανδημία και με τη μακροχρόνια υποστήριξη έργων. Θα επικεντρωθεί και στην διαθεσιμότητα φαρμάκων, εμβολίων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων Ο περιορισμός ε, των ασθενειών ε, που σχετίζονται με την μικροβιακή αντίσταση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχουμε και το Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου. Όλα αυτά θα αποφασιστούν από την Κομισιόν στα τέλη του έτους. Η κρίση του κορονοϊού μας έδειξε με δύσκολο τρόπο ότι Πρέπει να επεκτείνουμε και τις ψηφιακές μας δυνατότητες ε, στην ιατρική. Ε, πρέπει να σταματήσει ο κατακρισματισμός των ιατρικών δεδομένων και να, βελτιωθεί, να βελτιωθούν τα ψηφιακά ιατρικά συστήματα. Έτσι λοιπόν, στο Συμβούλιο έχουμε συμπεράσματα για την οργάνωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ευρώπης για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου ε, δεδομένων υγείας υπήρξαν επίμαχες συζητήσεις για μια εφαρμογή σε πανευρωπαϊκή που θα μπορούσε να προστατεύει καλύτερα τους πολίτες. Και εκεί χρειαζόμαστε διάφορες βελτιώσεις, το ξέρετε όλοι, τόσο καλά όσο και εγώ. Εξίσου σημαντική είναι και η υπόδειξη ότι χρειάζονται και επενδύσεις και μέσω άλλων μέσων του πολιτικού δημοσιονομικού πλαισίου για την ιατρική. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κυρίε και κύριοι, ένα πράγμα είναι σαφές. Το θέμα της υγείας στο μέλλον θα αποτελέσει κεντρική δραστηριότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την άποψή μου αυτό δεν είναι κακό για τα κράτη-μέλη γιατί μας το έδειξε η πανδημία. Χρειαζόμαστε εδώ περισσότερη Ευρώπη, μια Ευρώπη πιο ικανή να δράσει και είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Και η πανδημία του COVID-19 μας έδωσε για την ευκαιρία να σκεφτούμε Ποια μέτρα χρειαζόμαστε για την καταπολέμηση της τρέχουσας πανδημίας και για μελλοντικών κινδύνων για την υγεία. Ενωμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να καταστήσει και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολόκληρο τον κόσμο έναν πιο ασφαλή τόπο. Πολλοί έχουν στραμμένο το βλέμμα προς εμάς για να δουν πώς ελεύθερες δημοκρατικές κοινωνίες μπορούν να αντιμετωπίσουν τόσο δύσκολες κρίσεις ε, που αποτελούν υπαρξιακή κρίση για πολλοί κόσμο και πότε το στόχος μας είναι να προστατεύουμε τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά να δείχνουμε και αλληλεγγύη σε παγκόσμιο επίπεδο. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Before... Uh, Ευχαριστούμε. Πρωτού συνεχίσουμε να σας δώσω τα αποτελέσματα της, ε, ε, του πρώτου γύρου ψηφοφορίας, τα οποία έχουν ως εξής ορισμός της Χέλκα Μπέρμπερ ως μέλος του ελεγκτικού συνεδρίου. Εγκρίνεται η πρόταση. Ορισμός του εκτελεστικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών εγκρίνεται. Έτοιμα για κατεπήγον. Προκειμένου να εγκριθεί η αντιμετώπιση του COVID-19 εγκρίνεται, διεξαγωγή κλινικών δοκιμών εγκρίνεται, μοναδικές ψηφοφορίες. Τροποποίηση του κανονισμού 1303 κάθετος 2013 εγκρίνεται. Τροποποίηση του κανονισμού 2017-2454 εγκρίνεται. Ψήφισμα για την απαγωγή παιδιών που γονείς στην Ιαπωνία εγκρίνεται. Δικαιώματα ατόμων με διανοητική αναπηρία εγκρίνεται. Ψηφοφορίες για αιτήματα επί της διαδικασίας. Άρθρο 67, παράγραφος 1. Για τις οδικέ μεταφορές απορρίπτεται. Επίσης, όσον αφορά τον χρόνο οδήγηση, απορρίπτεται. Επίσης, όσον αφορά το καποτάζ, το ψήφισμα για την απόρριψη απορρίπτεται τροποποίηση των οδηγιών 2017-2455 και 2019-1995 η πρόταση για απόρριψη της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απορρίπτεται. Τροπολογίες της υπεύθυνη Επιτροπής με ε, μία ψηφοφορία 1 έως 9 εγκρίνονται. Οικονομικέ δραστηριότητε τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ετήσια έκθεση 2019. Απορρίπτεται η 4, η 15 εγκρίνεται. η 5 απορρίπτεται, η 6 απορρίπτεται. Παράγραφος 32, αρχικό κύμα, κειμένο πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 32, αρχικό κείμενο, παράγραφος 2 εγκρίνεται. Παράγραφος 35, αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Τροπολογία 1, εγκρίνεται. Παράγραφος 38, αρχικό κείμενο, πρώτο τμήμα, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, εγκρίνεται. Παράγραφος 41, αρχικό κείμενο, παράγραφος 1, ε, εγκρίνεται. 2, ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 3, πρώτο τμήμα, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, εγκρίνεται. Παράγραφος 55, αρχικό κείμενο, εγκρίνεται. Τροπολογία 7 απορρίπτεται. Τροπολογία 8 απορρίπτεται. Τροπολογία 9 απορρίπτεται. Παράγραφος 72 αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Τροπολογία 10 απορρίπτεται. Τροπολογία 11 απορρίπτεται. Τροπολογία 12 απορρίπτεται. Τροπολογία 13 απορρίπτεται. Τροπολογία 16 εγκρίνεται. 14 απορρίπτεται. 2 εγκρίνεται. Έλεγχο των οικονομικών δραστηριοτήτων τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ετήσια έκθεση 2018. Τροπολογία 7 απορρίπτεται. Παράγραφο 9. Αρχικό κείμενο. Πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφο 11. Ε, τροπολογία 1 απορρίπτεται. Παράγραφο 12. Αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Παράγραφο 15. Αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Παράγραφο 16. Αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Παράγραφος 19. Αρχικό κείμενο εγκρίνεται. Παράγραφος 20. Αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. 8 εγκρίνεται. Παράγραφος 24 αρχικό κείμενο πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα εγκρίνεται. Τροπολογία 10 απορρίπτεται. 11 απορρίπτεται. Τροπολογία 9 εγκρίνεται. 12 απορρίπτεται. Παράγραφος 36. Αρχικό κείμενο. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13 απορρίπτεται. 3 απορρίπτεται. 4 εγκρίνεται. 14 εγκρίνεται. 15 απορρίπτεται. 5 απορρίπτεται. 6 απορρίπτηκε. Τώρα, συνεχίζουμε με τη συζήτηση και θα δώσω το λόγο στην κυρία Κυριακίδη, εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Η συζήτηση αυτή ε, γίνεται μια κρίσιμη στιγμή στα πλαίσια μιας ε, πάρα πολύ σοβαρής, σοβαρότερης ε, κρίσης υγείας που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες. Με περιορισμούς στη μετακίνηση, στα ταξίδια, με δυσκολίες να αναπνεύσει η οικονομία μας μετά από μήνες εγκλισμού. Αλλά το άνοιγμα αυτό έρχεται συνοδευόμενο από κινδύνου. Γιατί κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση τις επόμενες εβδομάδες ή μήνες και είναι πάρα πολύ νωρί για να μιλήσουμε για τη ζωή μετά το COVID-19. Σίγουρα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή για να προβληματιστούμε και πρέπει να προβληματιστούμε από τα δύσκολα μαθήματα που παίρνουμε. Να προβληματιστούμε για το τι πρέπει να βελτιώσουμε, και να ενισχύσουμε τις δράσεις μας ώστε να προστατευτεί η Ευρώπη από μελλοντικέ αντίστοιχε κρίσει. Και πρέπει επίση να καθίσουμε και να σκεφτούμε ποιο μπορεί να είναι ο ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέματα υγεία και ποιε είναι οι ευθύνε των χωρών μελών. Σύμφωνα με τις συνθήκες. Την επόμενη εβδομάδα στις 15 Ιουλίου θα παρουσιάσουμε ένα πρόγραμμα δράσης το οποίο θέτει διάφορες ιδέες για να βοηθήσουμε τις χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν ε, καλύτερα και να διαχειριστούν καλύτερα οποιοδήποτε νέο ξέσπασμα του COVID-19. Και εδώ θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Ένα δεύτερο κύμα δυστυχώς δεν είναι αναπόφευκτο. Όμως εξαρτάται από μας να το ελέγξουμε και να προετοιμαστούμε γι' αυτό. Και ακόμα όταν έρθει και αν έρθει πρέπει να επικεντρωθούμε στο πώς θα ανακουφίσουμε τα συστήματα υγείας μας κυρίως όταν θα έρθει το φθινόπωρο και θα έχουμε και ε, γρήπη. Είναι σαφές ότι πρέπει η προσέγγιση μας να είναι μια προσέγγιση που την έχουμε όλοι μαζί ενιαία και να προστατεύσουμε όσο γίνεται καλύτερα ε, τους πιο ευάλωτους. Ε, πολλοί ακόμα και ευρωβουλευτές και πολίτες έχουν ζητήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει να παίξει πιο σημαντικό ρόλο όσον αφορά την υγεία. Και εγώ συμφωνώ βεβαίως και είμαι έτοιμη να συνεργαστώ μαζί σας προς αυτό το σκοπό. Και ως πρώτο βήμα θα πρέπει να ενισχύσουμε τη δυνατότητα που έχουμε να στηρίξουμε τις χώρες μέλη. Κάτι το οποίο απαιτεί έναν πιο ισχυρό ακόμα οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στους επόμενους μήνες θα ε, προτείνουμε να ενισχυθεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Ασθενειών και όσον αφορά την ικανότητά του και όσον αφορά την εντολή που έχει να αντιμετωπίσει τέτοιες κρίσεις. Και θα προτείνουμε επίσης να ενισχυθεί και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ώστε να μπορεί να συντονίσει τη δράση μας και να αποφεύγει την έλλειψη φαρμάκων. Πρέπει να δούμε πώς θα ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό πλαίσιο επίσης όσον αφορά τα διασυνοριακά θέματα υγείας. Μία από τις προτεραιότητες είναι τώρα να συζητήσουμε και το θέμα της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δημόσιας υγείας και τα όρια του. Έχω πει ήδη από την αρχή ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης ε, προσφέρει ένα πάρα πολύ καλό φόρουμ για να συζητήσουμε αυτό ακριβώς το θέμα και να δούμε τι είναι αυτό το οποίο μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα ε, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ξέρουμε ότι κάποια πράγματα δεν έχουν σύνορα. Ακόμα βέβαια και στην πιο δύσκολη κρίση πρέπει κανείς να βλέπει ευκαιρίες, γιατί υπάρχουν. Και υπάρχουν ευκαιρίες από αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα. Να ενισχυθεί η αυτονομία των δικών μας συστημάτων υγείας και φαρμάκων. Είναι ένα από τα κύρια μαθήματα που πήραμε. Γι' αυτό λοιπόν και προτείνουμε το πρόγραμμα αυτό για την ε, υγεία με 9,4 δισεκατομμύρια πρικοδότηση, κάτι το οποίο αποτελεί προτεραιότητα για την ανάκαμψή μας. Έχουμε ακούσει τους ε, πολίτες που λένε ότι πρέπει να είμαστε έτοιμοι, πρέπει να επενδύσουμε ε, στα συστήματα υγείας μας για το μέλλον. Χρειάζεται λοιπόν στενή συνεργασία και χρειάζεται και συμφωνία ανάμεσα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τις επόμενες εβδομάδες και μήνες για να έχουμε αποτελέσματα. Εγώ θα στηρίξω τις φιλοδοξίες αυτές. Συγχρόνως, και γνωρίζω πάρα πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό το θέμα, χρειάζεται και μία νέα στρατηγική για τα φάρμακα ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη στρατηγική αυτονομία του φαρμακευτικού μας τομέα και να φροντίσουμε να υπάρχει πρόσβαση σε φάρμακα, σε προσιτές τιμές από τους πολίτες μας. Σε συνεργασία λοιπόν με τους ενδιαφερόμενους για αυτή την ε, στρατηγική έχουμε προχωρήσει στις προτάσεις μας. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, οι επόμενοι έξι μήνε είναι κρίσιμη σημασία. Δεν είναι τώρα η στιγμή να επαναπαυθούμε η κατάσταση παραμένει πάρα πολύ εύθραυστη και αυτό το βλέπουμε σε πολλές χώρες μέλη. Αλλάζουν τα νούμερα από στιγμή σε στιγμή. Χρειάζεται λοιπόν ένα ασφαλές ε, εμβόλιο γιατί από ό,τι φαίνεται είναι η μόνη αποτελεσματική λύση για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Χρειαζόμαστε όμως ακόμα χρόνο γι' αυτό. Αποκοινούμε τις χώρες μέλη. Εμείς ε, κάνουμε διαπραγματεύσεις με τους ε, κατασκευαστές εμβολίων για να δούμε πότε θα μπορούμε να το έχουμε στη διάθεσή μας. Και θα φροντίσουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο ώστε να ε, αναπτυχθούν εμβόλια που να είναι αποτελεσματικά και προσιτά ε, για όλους, χωρίς να ξεχνάμε κανέναν πρέπει να συνεχίσουμε να στηρίζουμε και χώρες και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορέσουμε να προστατεύσουμε όλο τον κόσμο και μέσα και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως τους πιο ευάλωτους. Πρέπει να φροντίσουμε να σώζουμε ζωές. Από την αρχή της πανδημίας είχα 26, 28 συναντήσεις με όλους τους υπουργούς υγείας και είμαι σε συνεχή επαφή μαζί τους. Είναι ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε το συντονισμό που χρειαζόμαστε, τη συνένεση και τη συνεργασία μεταξύ μας για να έχουμε αποτελέσματα. Πρέπει να βάλουμε από κοινού τους πόρους που έχουμε στη διάθεσή μας και από κοινού να αντιμετωπίσουμε τα ζητήματα που είναι κοινά για όλους. Είναι το πρώτο μάθημα και το πιο σημαντικό που πήραμε από αυτή την κρίση, ότι πρέπει να ανταποκρινόμαστε στις προσδοκίες των πολίτων και Ευρωπαϊκή, των πολιτών και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει περισσότερο ισχυρό ρόλο από την αρχή. Γιατί τα θέματα υγείας δεν σταματούν στα εθνικά σύνορα και συλλογικά έχουμε χρέος και ευθύνη να το λάβουμε υπόψη μας αυτό. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστούμε κύριε ε, Επίτροπε. Και τώρα έχουμε τις αγορεύσεις των εκπροσώπων των πολιτικών ομάδων. Ξεκινούμε από το ΕΛΚ. 1,5 λεπτό, κύριο Λίζε. Αγαπητοί συνάδελφοι, το Μάρτιο, τον Απρίλιο στην αρχή της ε, πανδημίας ε, και εγώ όπως άλλοι στο ιατρικό επάγγελμα επέστρεψα στο ιατρείο μου και το πρώτο που διαπίστωσα όταν ρώτησα τους συναδέλφους δεν είχαμε μάσκες. Ε, επισκέπτες, ε, ε, είχα πελάτες και χρειαζόταν να προστατεύω το στόμα μου με το χέρι μου. Για πολλούς γιατρούς και νοσηλευτές στον Πέργαμο, στη Μαδρίτη, αυτό σημαίνει ότι μολύνθηκαν και σήμερα έχασαν τη ζωή τους. Αυτά είναι Έχουμε πολλά παραδείγματα ότι δεν πρέπει να εξαρτώμαστε σε τόσο μεγάλο βαθμό από την Κίνα και τους λοιπούς όταν πρόκειται για ζωτικά θέματα υγείας. Έτσι λοιπόν χαίρομαι που έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αυτό το ψήφισμα σήμερα. Ευχαριστώ τον Μάνφροντ Βέμπερ που το υποστήριξε αυτό να δεχθούμε αυτό το ψήφισμα και ευχαριστώ και τους συναδέλφους άνδρες και γυναίκες για την εξαιρετική συνεργασία ε, υποστηρίζουμε τις προτεραιότητες της Γερμανικής Προεδρίας του Συμβουλίου και τις προτάσεις της Επιτροπής. Τους επόμενους μήνες θέλουμε μαζί να επιτύχουμε πολλά, αλλά και μακροχρόνια, μακροπρόθεσμα θέλουμε μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δέσμευση για την υγεία. Στο παρελθόν τα κράτη-μέλη έβλεπαν με πρισκεψία τα θέματα υγείας, έλεγαν ότι είναι εθνικά. Ήταν λάθος μας το έδειξε τώρα αυτός ο ιός και άλλες απειλές ε, δεν σταματάνε στα σύνορα. Έτσι χρειαζόμαστε μια Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. Ευχαριστώ πολύ. Thank you on behalf of... ευχαριστούμε. Από τους σοσιαλδημοκράτες έχει το λόγο η κυρία Φριτσόν για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ένα είναι το σίγουρο ότι δεν σταματάνε τα σύνορα την ε, πανδημία και αυτή η κρίση μας δίδαξε πόσο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί κανένα κράτος μόνο του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ε, κρίση. Χρειάζεται περισσότερο συντονισμός, περισσότερη συνεργασία στην Ένωση και είναι ξεκάθαρο το εξής ότι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν την αρμοδιότητα για τον τομέα της υγείας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουν τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι σωστό να έχουμε μια ένωση υγείας. Έτσι θα έχουμε μάθει κάτι από αυτή την κρίση και θα τα καταφέρουμε καλύτερα στο μέλλον για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιε κατάσταση για να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό που χρειάζεται ο κόσμο όσον αφορά τα φάρμακα, όσον αφορά το προφυλακτικό, προστατευτικό υλικό και έτσι θα μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά χρειάζεται περισσότερη συνεργασία. Σα ευχαριστώ για τώρα για το Ρήνιο η κυρία Τριέλ Νουάρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να σα τα πω στα Γαλλικά, κύριε Επίτροπε, κυρία Επίτροπε. Περνούμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, μια γενομική κρίση. Πρόκειται περί μια τραγωδία, απώλεια ανθρωπίνων ζώων, αλλά επίση έτσι συνειδητοποιηθήκαμε. Οπότε α εκμεταλλευτούμε αυτή την μοναδική ευκαιρία και να αντλήσουμε κάποια συμπράσματα. Όλοι και διακομματικά είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε με τον ΠΟΗ να ετοιμάσουμε έναν μηχανισμό, έναν μηχανισμό απόκρισης στα υγειονομικά. Και χάρη σε εσά, αγαπητή Στέλλα, προχωράμε προς τα εκεί είναι μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τις αρμοδιότητες των ε, ευρωπαϊκών υπηρεσιών και οπότε να είναι περισσότερο αποτελεσματικές είναι μια ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε μια αποτελεσματική πρόληψη και αυτό μέσα από την παιδεία, την εκπαίδευση για την υγιεινή να σεβαστούμε το Green Deal όσον αφορά την διατροφή, την ε, μόλυνση, ρήπανση την ε, αλλαγή του κλίματος και οπότε θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν καλύτερες ε, υποδομές στον τομέα της υγείας με συγκεκριμένα κριτήρια και να μην γίνει Ευρωπαϊκή Ένωση ε, απλώς διανομέας ε, χρημάτων. Επίσης, όσον τα ιατρικά δεδομένα, τις σωστές πρακτικές, ε, να έχουμε ένα σημείο αναφορά στην Ευρώπη και έχουμε επίσης ευκαιρία να είμαστε ανεξάρτητοι αυτάρκες για τα φαρμακευτικά, για τα προϊόντα της υγείας και να υπάρχει προσβασιμότητα από όλους τις υπηρεσίες υγείας και έτσι να έχουμε την ευκαιρία να επιδείξουμε αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας, να λάβουμε υπόψη αυτού ε, αυτούς που έχουν πληγεί περισσότερο, δηλαδή τις περιοχές της Ευρώπης που χτυπήθηκαν περισσότερο, αλλά και τις πιο ευάλωτες τρίτες χώρες. Τέλος, σας προτείνω να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία για να δούμε πώς, ε, ε, πώς σχετίζεται η υγεία με όλες μας τις πολιτικές και έτσι θα ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των συμπολιτών και έτσι ε, όλοι μαζί θα προχωρήσουμε στο όραμα μιας Ευρώπης που προστατεύει με συγκεκριμένους τρόπους. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε εκ μέρους του ΑΕΔ η κυρία Σαρντόνα. Να ευχαριστώ Σήμερα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ότι υπάρχει πανδημία και απάντησε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα ψήφισμα για την υγειονομική στρατηγική της Ευρώπης μετά από τον COVID. Έχετε ανταποκριθεί ε, κακά και καθυστερημένα στην πανδημία. Το κλείσατε το πρόβλημα. Τελείωσε ο COVID. Πάμε στην επόμενη φάση. Αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί εδώ τα πράγματα. Σήμερα στο ψήφισμα καταφέρατε να βάλετε ένα σωρό πράγματα τη σύνδεση μεταξύ του COVID και τη κλιματική αλλαγή. Αναφορά στο γεγονό ότι οι εθνικέ μειονότητε επλήξαν περισσότερο, επλήξαν όλοι και ειδικότερα οι μεγάλοι άνθρωποι. Ε, αναφέρεστε στους ΛΟΑΤ και στην αντισύλληψη. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει να κάνει με τον κορονοϊό. Αλλά ένα πράγμα κάνετε πολύ καλά. Αυξάνετε τι ε, πολυθρόνε, τι καρέκλε. με την πανδημία ως αιτιολογία αυξάνεται τους οργανισμούς ε, και τις θέσεις που θα, και τον κόσμο που θα απασχοληθεί εκεί, την γραφειοκρατία. Το βλέπουν οι πολίτες. Θέλουμε απαντήσεις τώρα, όχι άχρηστη προπαγάνδα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέλου των Πρασίνων, έφα η κυρία Ντεσούτερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Λυπάμαι που χρειαζόταν μια παγκόσμια κρίση υγεία για να βάλουμε την υγεία ως προτεραιότητα στο ε, θεματολογιό μας. Αλλά ας κοιτάξουμε προ τα μπρος, ας μάθουμε από αυτή την κρίση και α βεβαιωθούμε ότι στο μέλλον η υγεία θα παραμένει ψηλά στην ατζέντα μας. Πέραν τη ε, ετοιμότητα που πρέπει να βελτιώσουμε, πρέπει να καταβάλουμε προσπάθειε για μια ολοκληρωμένη ε, πολιτική στον τομέα τη υγεία και να δούμε και άλλου θεμελιώδου τομεί. Πρέπει να εστιαστούμε στην πρόληψη είναι επωφελής και για τους πολίτες και για τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Δεύτερον, ας αναθεωρήσουμε το φαρμακευτικό μας σύστημα, να διασφαλίζουμε πρόσβαση σε φθηνά φάρμακα για όλους. Ε, και τρίτον, ας ενισχύσουμε τη μία προσέγγιση για την υγεία, την ενιαία προσπάθεια για την υγεία. Αλλιώ ε, όλε οι προσπάθειε ε, θα είναι καταδικασμένε. Πρέπει να δούμε την αλεξάρτηση μεταξύ τη δική μα υγεία και τη υγεία του πλανήτη. Ε, εξαρτάται από εμά. Θα θυμόμαστε τον COVID-19 ως τη χειρότερη υγειονομική κρίση της πρόσφατης ιστορίας παγκοσμίω ή θα την θυμόμαστε ως την αφετηρία μιας βελτιωμένης ε, δημόσιας πολιτικής υγεία στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Εκ μέρου του ECR η κυρία ε, Δελαπίσα Καριών. Καλησπέρα, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, Ήλπιζα το ψήφισμα αυτό για τη δημόσια υγεία να είναι ένα τεχνικό έγγραφο με λεπτομέρειες πώς να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Όχι όμως. Ακούμε για νέους οργανισμούς, για νέους θεσμούς, ε, προσπάθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να αυξήσει τελικά την εξουσία των Βρυξελών ε, πάνω στα έθνη. Πρόκειται για λέξεις ε, καινούριες περιεχομένου, η πράσινη συμφωνία, η ανθεκτικότητα, δεν ξέρω εγώ τι λέξεις για να καθησυχάζουν συνειδήσεις και τίποτα άλλο. Ενώ ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η κυρία Μέρκελ μας λέει πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Ενώ εδώ μιλάμε για κανονικότητα και για συμφέροντα τα οποία είναι υπερεθνικά. Οι ανάγκες μας όμως είναι διαφορετικές. Στην υγειονομική αυτή κρίση αυτό που χρειαζόμαστε είναι συγκεκριμένα πρωτόκολλα δράσης ε, με σαφήνεια, με ακρίβεια και που εφαρμόζονται αμέσως και να μας προστατεύουν πραγματικά από οποιαδήποτε νέα έξαρση ή νέους ιούς. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αντικαθιστά τα κράτη-έθνη, αλλά διευκολύνει την ελεύθερη συνεργασία σε θελοντική βάση και με λογική πάνω απ' όλα. Μόνο έτσι θα ενισχυθεί η Ευρώπη. Μόνο έτσι θα βγούμε από την κρίση αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. και τώρα να προχωρήσουμε στην δεύτερη ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε αυτά τα οποία βλέπετε στην ημερήσια διάταξη, αυτά τα οποία εγκρίθηκαν και θα αρχίσουμε στις 8.30 την ψηφοφορία και θα την ολοκληρώσουμε στις 9.40 με την ίδια διαδικασία όπως και στην προηγούμενη ψηφοφορία θα γίνουν όλες ονομαστικά και μπορείτε να επαληθεύσετε το τι ψηφίζατε, τα δύο αποτελέσματα μπορείτε να, τα δείτε από αυτά τα οποία θα ανεβάσουμε στο website. Τώρα έχουμε την έναρξη της ψηφοφορίας. Έρχεται μέχρι τις 9.45 να ψηφίσετε. Τα αποτελέσματα της δεύτερης ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν αύριο στις 9. Ε, ε, Η κυρία Κονέσουνα, έχετε δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδελφούς που συμμετέσχουν για την σύνταξη αυτού του κειμένου, αυτό το κοινό ψήφισμα το οποίο είναι μια ευρεία συνένεση διακομματική. Η κατάσταση αυτή είναι χωρίς προηγούμενο, άρα χρειάζονται και αντίστοιχες λύσεις. Το business as usual πια δεν αποδίδει. Χρειάζεται στροφή, αλλαγή πορείας. Θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία στην ευρωπαϊκή πολιτική και να δούμε τι ε, γίνεται πρώτα πρώτα με αυτούς που εργάζονται εδώ στο Κοινοβούλιο γιατί είδαμε ότι απέδειξε η πανδημία ότι δεν έχει Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τις αρμοδιότητες που έπρεπε για να αντιμετωπίσει την κρίση. Άρα χρειάζεται μια άλλη διαχείριση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων. Θα πρέπει να ελπίσουμε στην Γερμανική Προεδρία. Αλλά δεν είμαι και τόσο σίγουρη, γιατί εδώ και χρόνια αυτή η χώρα μπλοκάρει πάρα πολλές νομοθεσίες που θα βοηθούσαν. Να δούμε τι θα γίνει με τα φάρμακα των σπανίων ασθενειών, να δούμε τι θα γίνει με τα εμβόλια, τι γίνεται με το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί. Θα πρέπει να είναι διαθέσιμα τα φάρμακα και αποτελεσματικές θεραπείες. Οι φαρμακοβιομηχανίες σήμερα έχουν τα μέσα. Δεν θα πρέπει να είναι προς ζημίαν, αλλά υπέρ της υγείας του κόσμου. Θα πρέπει να υπάρχει προσβασιμότητα σε πάσα διάγνωση. Γι' αυτό και με τον συναδελφό Μποτέγκα και άλλους είπαμε ότι πρέπει να προχωρήσει το ψήφισμα Right to Cure και με μια τέτοια λύση να έχουμε καλύτερη μπούσουλα για το μέλλον. Τώρα, για τους μη εγγεγραμμένους η κυρία Ροντινίλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η πανδημία μας απέδειξε το ότι χρειάζεται περισσότερη συνεργασία, ολοκλήρωση και αλληλεγγύη στην δημοσία υγεία. Γιατί νομίζω ότι αυτή η ευρωπαϊκή στρατηγική είναι μη ρεαλιστική. Αυτό θα πρέπει να καλύψει ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο. Αλλά τώρα έχουμε business σε σχέση με την αναζήτηση του εμβολίου. Νέες στρατηγικές. Πρώτα-πρώτα όμως μία επιλογή. Να δούμε τι θα γίνει με τις επενδύσεις στην υγεία και την ε, έρευνα. Να δώσουμε τη σωστή απάντηση στον ε, κόσμο. Να υπάρχουν υψηλά στάνταρ στον τομέα των υγειονομικών, πέραν των ε, μακροοικονομικών μεταβλητών. Να φρενάρουμε το σύμφωνο σταθερότητας και να το καταργήσουμε μόλις ολοκληρωθεί η κρίση. Ο πραγματικός ιός είναι η λιτότητα, άρα να σταματήσει. Και έτσι να νικήσουμε το, την πανδημία και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις για την Ευρώπη. Και τώρα. Συνεχίζουμε με τους εκπροσώπους πολιτικών ομάδων, η κυρία Μονσεράτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Βρισκόμαστε στη μεγαλύτερη υγειονομική κρίση που έχουμε ζήσει ποτέ, με φοβερές επιπτώσεις και κοινωνικές και οικονομικές. Οφείλουμε λοιπόν να έχουμε καλύτερο συντονισμό και να ενισχύσουμε τα συστήματα υγείας μας για να αντιμετωπίζουμε τέτοιες απειλές. Εμείς ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας υπέρ της ευημερία των Ευρωπαίων, υπέρ της υγείας, έτσι ώστε να έχουν μεγαλύτερη προστασία. Και απέναντι σε αυτή την υγειονομική κρίση, αλλά και σε χρόνιες ασθένειες, αυτό ακριβώ πρέπει να κάνουμε. Θέλουμε μια Ευρώπη για την υγεία και η υγεία να ληφθεί υπόψη σε όλε τι πολιτικέ με περισσότερο προπολογισμό, με περισσότερα χρήματα, περισσότερε αρμοδιότητε επίσης και τη δυνατότητα να παίρνει αποφάσεις η Ευρώπη για αποτελεσματικές απαντήσει σε θέματα υγείας. Χρειάστηκε πρόληψη, αποτελεσματική, περισσότερη έρευνα για να έχουμε στη διάθεσή μας φάρμακα και θεραπείες που να είναι αποτελεσματικά, αλλά βέβαια και εμβόλια στα οποία να έχουν πρόσβαση όλοι Πρέπει λοιπόν να δούμε την παραγωγή και την υγεία γενικότερα, από την οποία μπορούν να δημιουργηθούν νέε θέσει απασχόλησης. Έχουμε τα καλύτερα συστήματα υγείας στον κόσμο, Ακριβώ γι' αυτό και αποτελούμε σημείο αναφορά για την υγεία παγκοσμίω. Αυτή λοιπόν είναι η Ευρώπη που υποστηρίζουμε, τη υγεία και των ανθρώπων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ τους ευρωβουλευτές να τηρούν το χρόνο τους. Για ένα λεπτό, ο κύριος Σουχέη. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί φίλοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να είναι δίκαια εάν εξαρτάται το κατά πόσο έχει πρόσβαση στην υγεία ή όχι από το που γεννήθηκες είναι δυνατόν να λέμε ότι δεν είναι στρατηγική σημασία. Ω Ούγγρο, ω ε, σοσιαλιστή, μέλο των σοσιαλδημοκρατών, εγώ δουλεύω για να δημιουργήσουμε ένα μέλλον για τα παιδιά μα εδώ στην Ευρώπη. Και ένα μέλλον που να περιλαμβάνει την Ευρώπη για την υγεία. Ώστε στη χώρα μου να μην μπορεί να υπάρχει κάποιος ο οποίος να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να πεθάνει επειδή βρίσκεται στην Ουγγαρία από ό,τι θα είχε αν ήταν στη Γερμανία και όταν ε, για τον ίδιο αριθμό ασθενών στην Ουγγαρία έχουμε τρεις-τέσσερις νοσηλευτικό προσωπικό ενώ το αντίστοιχο νούμερο στη Γερμανία είναι 12. Αν επ' αυτού πρόκειται να στηρίξω το πρόγραμμα το Ευρωπαϊκό για την Υγεία. Εμείς δεν θέλουμε να αφαιρέσουμε κάτι από τις χώρες μέλη, θέλουμε να τους δώσουμε κάτι, υγεία. Ευχαριστούμε. Στεφανιούτα. Κύριε Επίτροπε, η ευτυχία εξαρτάται από την ελευθερία και η ελευθερία εξαρτάται από το θάρρος. Έτσι έχει πει κάποιος ηγέτης. Σήμερα δεν είμαστε ευτυχείς επειδή δεν αισθανόμαστε την ελευθερία. Και θα ήθελα εδώ να έχουμε ε, και να ζητήσω ένα ισχυρό πρόγραμμα για την υγεία. 85% των χρημάτων για το πρόγραμμα αυτό έρχεται από το Next Generation Europe. Οι νομικές υπηρεσίες στο Συμβούλιο έχουν εκφράσει κάποιες ανησυχίες. Οπότε δεν ξέρω, όπως είπε και ο κύριος Χέλη, τελικά σε κάποιες χώρες ε, κατάσταση είναι διαφορετική από άλλες, διότι άλλες έχουν ε, δωμάτια στα νοσοκομεία πέντε αστέρων και άλλοι δεν έχουν καν πρόσβαση στο νοσοκομείο. Έχουμε όμως τώρα την ευκαιρία να συνεισφέρουμε στην ευτυχία των Ευρωπαίων πολιτών προσφέροντάς τους καλύτερη υγεία, την καλύτερη υγεία στον κόσμο, την ευρωπαϊκή υγεία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Μελά. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώ αποτελεί ανακρίκο συνεργασία για τα θέματα υγεία. Αλλά αν αποστεριώρει, δηλαδή έξι μήνε μετά από την πανδημία, να υιοθετήσουμε μια στρατηγική για την υγεία, ε, αυτό είναι η απόδειξη ότι έχει αποτύχει στην αποστολή τη η Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να προλαμβάνουμε. Κάτι το οποίο δεν έκανε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια, ένα ειδικό οργανισμό, ο Κέντρο Πρόληψη και Ελέγχου, αλλά δυστυχώ ο οργανισμό αυτό μόνο στι 22 Ιανουαρίου, ένα μήνα δηλαδή μετά την αρχή που άρχισαν να κυκλοφορούν οι επίσημε πληροφορίε, αντέδρασε. Έπειτα είναι το θέμα τη χρηματοδότηση. Οι χώρε ε, μέλη όταν ε, έχουν τόσο κακή οικονομική κατάσταση εξαιτία τη κρίση, τι έγινε η απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ασύντακτη τουλάχιστον. Σήμερα με το ψήφισμα αυτό ζητάμε περισσότερη Ευρώπη, να δημιουργηθεί μια Ευρώπη της υγείας. Για μένα αυτό πλήττει την επικουρικότητα, την ίδια την αρχή της επικουρικότητας. Νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά όργανα θα μπορούσαν να κάνουν καλύτερα πράγματα να σκεφτούν το άνοιγμα των συνόρων ε, στο χώρο Σέγγεν. Όμως ο ιός κυκλοφορεί και ο δικός και ο αέρα, από θάλασσα. Για ένα λεπτό η κυρία Μέτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Αυτή η κρίση το έδειξε πολύ σωστά. Για μια πιο δίκαιη Ευρώπη χρειαζόμαστε ποιοτική πρόσβαση στην υγεία για όλους. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια Ευρώπη της υγείας που θα μας επιτρέψει καλύτερο συντονισμό για να επενδύσουμε σε μια Ευρώπη που θα εξυπηρετεί τους πολίτες, άνδρες και γυναίκες. Να υπογραμμίσω δύο σημεία. Πρώτα απ' όλα η λιτότητα, η κρίση του COVID-19 εξάντλησαν τα δημόσια νοσοκομεία και τους ε, το προσωπικό του. Πρέπει να υποστηρίξει η Ευρώπη τι επενδύσει των κρατών μελών για τι υποδομέ δημοσία υγεία. Δεύτερον, η υγεία δεν ε, πρέπει να αφαιθεί μόνο στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να επενδύσει, να δημιουργήσει δημόσια εργαστήρια και κέντρα ερευνών, τα ευρήματα των οποίων θα ωφελήσουν όλου. θα βοηθήσουν να έχουμε λιγότερο ακριβές θεραπείες επίσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. 1,5 λεπτό ο κύριος Γκόκινγκ. Η πολιτική υγείας δεν είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Το έδειξα ε, και τα τελευταία χρόνια. Ο COVID-19 όμως έδειξε ότι είναι ευρωπαϊκή πολιτική. Ε, είδαμε πόσο αδύναμα είναι τα, και διαφορετικά τα συστήματα υγείας στην Ευρώπη. Εγώ έρχομαι από μια χώρα όπου είμαι ευγνώμων γιατί είναι πολύ καλό το σύστημα. Έχω τρία υγιή παιδιά και βλέπω τι γίνεται σε άλλες χώρες και λέω έχει έρθει η ώρα να δράσουμε. Από τον COVID-19 ήρθε η ώρα να μάθουμε τι θα κάνουμε με τη στρατηγική μετά τον COVID-19. Πρέπει λοιπόν να μάθουμε ότι όχι μόνο θα έχουμε σχέδια άμεσης αντιμετώπιση ε, οποιασδήποτε πανδημίας, αλλά πρέπει τα συστήματα υγείας στις επιμέρους χώρες να υφίστανται ε, σε συνθήκες κοινέ για την έρευνα για παράδειγμα για ε, πήγοντα περιστατικά ε, ώστε να αποφεύγουμε μέσω της προορής αναγνώρισης και εντοπισμού των περιστατικών. Βλέπουμε στην Ευρώπη και για την περιθέλψη των καρκινοπαθών Χρειαζόμαστε όλα αυτά, χρειαζόμαστε πρότυπα ποιοτικά, δεσμευτικά. Να υπάρχει δηλαδή ένα πλαίσιο και φυσικά να λαμβάνουμε υπόψη την επικουρικότητα Έχουμε πάρα πολλού ε, εδώ βουλευτέ που προέρχονται από το χώρο τη υγεία. Το Σεπτέμβριο στο Στρασβούργο θέλω να προσπαθήσουμε να του φέρουμε όλου γύρω από το ίδιο τραπέζι, ώστε στο μέλλον, ε, εδώ στο Κοινοβούλιο, να μπορούμε να ε, λάβουμε και αποφάσει για την, πολιτική, την πανευρωπαϊκή πολιτική για την υγεία. Ένα, μισή, ένα λεπτό η κυρία Πόλφιερ Ένα λεπτό η κυρία Ευχαριστώ. Δεν έχει ανάψει το μικρόφωνο του η Απόψε συνεδριάζουμε και συζητούμε, αλλά θα πρέπει να αντιλήσουμε συμπεράσματα από αυτή την κρίση που περνούμε. Θα πρέπει να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στο μέλλον. Και θέλω να σας πω κάτι σημαντικό για μένα. Είναι κάτι σε σχέση με την ε, πανδημία, κάτι που σχέση με την ε, μικροβιακή ε, αντοχή. Πέθαναν τόσες εκατοντάδες χιλιάδων και επομένως το σημαντικό είναι να μάθουμε πώς γίνεται αυτή η ανθεκτικότητά μας σε αντίστοιχα προβλήματα στο μέλλον. Ήταν σωστό να προωθήσουμε τέτοιο ψήφισμα, αλλά ας αρχίσουμε να σκεπτόμαστε και άλλα σχετικά. Να σκεφτούμε τις ευθύνες μας για τα αντιβιωτικά, για έρευνα περισσότερη που θα μας βοηθήσει για τέτοιες ε, απειλές, συνεργασία, νέες τεχνικές και άλλες προσπάθειες. Όλες οι πολιτικές ομάδες να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ένα λεπτό έχει το λόγο ο κύριος Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Η πανδημία μας υπενθύμησε ότι είναι δημόσιο αγαθό, παγκόσμιο η υγεία. Είναι κάτι που είναι προϋπόθεση για εθνική ασφάλεια. Οπότε δεν αρκεί όσο και χρειάζεται να έχουμε εθνικές αρχές ε, προσβάσιμες, αποτελεσματικέ κλπ. Αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση της Υγείας και να έχουμε έτσι κάποια ελάχιστα πρότυπα να υπάρχει ένα τεστ αντοχής των εθνικών συστημάτων υγείας, μηχανισμός ταχείας απόκρισης, να θωρακίσουμε το πώς θα μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική, μια αυτάρκεια στα φάρμακα εδώ για την Ευρώπη, για μας. Άρα περισσότεροι πορεία για την έρευνα στα φάρμακα και να υπάρχει και για τα ζώα και για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο δεν αρκεί να λέμε μπράβο στους εργαζόμενους ε, στην υγεία και να το κάνουμε και κάθε μέρα για αλλά εμείς τα θεσμικά όργανα έχουμε ευθύνη καθήκον να έχουν εργασιακές συνθήκες που αναλογούν στον ιορισμό που επέδειξαν τους τελευταίους μήνες σε όλη την Ευρώπη. Ε, αυτό θα πρέπει να κάνει η, Ευρωπαϊκή Ένωση Υγείας. One minute, Mrs. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαστε εγκλωβισμένοι σε ένα σύστημα όπου οι μέτοχοι από τις μεγάλες πολυεθνικές έχουν ε, συμφέρον να απολυθούν ε, τα φάρμακά τους. Και έχουμε να κάνουμε με έναν τεράστιο τομέα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τη φιλοδοξία να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματικά πρέπει να καταλάβει ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες ε, δεν φροντίζουν πάντα για το καλό, ότι έχουν φτιάξει το δικό τους ε, κρυστάλλινο πύργο. Το σύστημα αυτό πρέπει να αλλάξει. Και τώρα έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε τα πράγματα, να δημιουργήσουμε μια αλληλεγγύη με συνεργασία μεταξύ των χωρών μελών να αναγκάσουμε τις αγορές όταν παράγουν φάρμακα να υπάρχει διαφάνεια και να είναι προσιτά για τον κόσμο. Και δεν μπορεί να κερδοφορούν οι εταιρείε αυτές στην πλάτη των Ευρωπαίων πολιτών και της υγείας τους. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό η κυρία Τότ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ο κορονοϊός θα μας συνοδεύει στη ζωή μας για κάμπος ακόμα. Δεν ξέρω πότε θα βρούμε την κανονικότητά μας και πάλι. Πολύ επικρίνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση τους τελευταίους μήνες και είναι αλήθεια. Πρέπει να το πούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον στην αρχή δεν κατάφερε να δράσει αποτελεσματικά για να προστατεύσει τον κόσμο από τον κορονοϊό. Τα εθνικά μέτρα είναι αναγκαία, και η συνεργασία είναι αυτό το οποίο αποδείχτηκε ότι βοηθάει. Πρέπει τώρα να στραφούμε προς το μέλλον. Έχουμε μπροστά μας ένα έγγραφο με στόχο να καθορίσει τη στρατηγική μας μετά τον κορονοϊό για τη δημόσια υγεία. Και από αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή σας στο εξή. Κατά τη γνώμη μου, δεν πρόκειται για ένα ελάχιστο σύστημα υγείας ε, που χρειαζόμαστε, όχι, αλλά χρειαζόμαστε τη μέγιστη προστασία της υγείας των ε, πολιτών. Πρέπει να υπάρχει συνεργασία με τις χώρες μέλη και να δούμε πόσο καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και το θέμα των εμβολίων. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό, ο κύριος Σεχήμ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αυτή η κρίση μας έμαθε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη συνεργασία στα θέματα της υγείας. Αυτό χρειάζεται, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τέτοιε κρίσει για να έχουμε αρκετέ μάσκες, για να έχουμε εξοπλισμό, για να έχουμε φάρμακα. Ενωμένοι είμαστε περισσότερο δυνατοί. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε και δεν πρέπει να αφήνουμε να εξαρτώμεστε από τον έξω κόσμο εκτό Ευρώπη. Όχι. Η υγεία Βέβαια, είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών, αλλά είδαμε ότι η συνεργασία μπορεί να μας προστατεύσει, γι' αυτό και καλωσορίζουμε το νέο αυτό πρόγραμμα για την υγεία. Πρέπει επίσης να φροντίζουμε την υγεία των εργαζομένων. Οι κανόνες να είναι τέτοιοι που να προστατεύουν τους εργαζόμενους και ε, στους χώρους εργασίας τους από προβλήματα υγείας που μπορεί να υπάρχουν εκεί. Συχνά εργάζεται ο κόσμος χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. Και αυτό είναι ντροπή. Πρέπει να σταματήσει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Το λόγο τώρα έχει η Επίτροπος, η κυρία Κυριακίδη, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, κύριε Επίτροπε. Everybody. Η Επίτροπος. Άκουσα προσεκτικά όλους και πρέπει να σας πω ότι είπατε πολλά που ως επιτοπλίστων με βρίσκουν σύμφωνοι. Ο Πίτερ Λίζερ. Είπα ότι δεν σταματούν στα σύνορα οι απειλές για την υγεία. Ε, γίναμε όλοι μάρτυρες σε τούτο. Και επίσης ε, θυμάμαι σε σχέση με το ΕΛΚ ε, που είχατε επισημάνει τις ελλείψεις και στο EU for Help βάλαμε ως τμήμα των προβλεπωμένων παρεμβάσεων το να έχουμε στρατηγικά αποθέματα Συγγνώμη, όχι μόνο όχι για το ΕΛΚ. Δεν λέει για το ΕΛΚ, λέει για το προστατευτικό υλικό. Χρειάζεται προστατευτικό υλικό, επομένω, λέει η Επίτροπο, ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για περαιτέρω κρίση. Δεν θα είναι μόνη αυτή η κρίση. Πολλοί από εσά είπατε ότι κανεί δεν μπορεί μόνο του να αντιμετωπίσει την κρίση. Ε, αυτό όντω το διαπιστώσαμε. Επίσης αναφέρατε και το θέμα τη επικουρικότητας, οπότε θα πρέπει σχετικά με αυτό να είμαστε σαφείς, γιατί και στο ισχύον άρθρο 168 ε, τα λέει, αλλά πάλι και στα πλαίσια του άρθρου πολλά μπορούμε να κάνουμε και έχουμε ένα σωρό ε, δράσεις στα πλαίσια του 168. Άρα έχουμε πολλά περιθώρια και ε, σίγουρα έτσι μπορεί να γίνει μεγάλη σημαντική στροφή στον τομέα της υγείας. Ε, είπατε τη λέξη τραγωδία, ε, κυρία Και όντως συμφωνώ μαζί σας, ε, γιατί το τελευταίο πεντάμινο, ε, Λενουάρ, για μένα το θέμα δεν ήταν μόνο τα νούμερα. Κάθε μέρα ξύπναγα, ε, άκουγα τα κρούσματα, άκουγα τους θανάτους, ε, και ήξερα ότι πίσω από τα νούμερα υπάρχουν ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες ιστορίες και ένα σωρό τέτοιες ιστορίες παρήλασαν ε, ήρθαν στο επίκεντρο τα, τους τελευταίους μήνες και βέβαια αναφέραμε το ότι έχουμε όραμα, έχουμε φιλοδοξία ε, σε σχέση με το πώς θα ενισχύσουμε ε, τον, τον φορέα για τις επιδημίες το ECDC και γενικότερα τα θεσμικά όργανα. Κυρία Ντεσούτερ, τα, είπατε, χρειάζεται η πρόληψη, ε, ενιαίος φορέ, ενιαία πολιτική υγείας, να δούμε τι γίνεται και με τις μη ε, μεταδιδόμενες νόσους και επίσης να δούμε πώς θα αναβαθμιστούμε και θα έχουμε πιο θωρακισμένα συστήματα υγείας. Ε, αυτά είναι σίγουρα οι στόχοι μας στον τομέα της υγείας και επίσης Κάποιος... Α, η κυρία Κονιέτσκα, ανέφερε ότι αυτή η κατάσταση χωρίς προηγούμενο, ε, βέβαια, γι' αυτό χρειαζόμαστε και λύσεις χωρίς προηγούμενο. Αυτό είναι το EU for Health. Είναι μια πρόταση φιλόδοξη που θα μπορούσε να φέρει την επιθυμητή στροφή στην πολιτική μας επίσης κυρία Ροντινέλη ότι παρά είμαστε αισιόδοξοι και δεν είμαστε ρεαλιστές. Ναι, είμαστε φιλόδοξοι, έχετε δίκιο, αλλά είμαστε ρεαλιστές από την άλλη και αν θέλουμε να κάνουμε τη διαφορά θα πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα για την επόμενη επταετία. Επίσης μας είπατε για περισσότερο συντονισμό που χρειάζεται σε κάθε επίπεδο. Ε, βέβαια, θα πρέπει με συνεργασία να καταφέρουμε να είμαστε η πιο υγιής περιοχή του κόσμου. Έτσι θα πρέπει να δούμε το θέμα να προστατεύσουμε βέβαια και τα δικαιώματα των ασθενών. Επίσης μας είπατε και τι γίνεται με τον προϋπολογισμό. Βεβαίως και εκεί υπάρχουν ζητήματα, τα διερευνούμε με τους νομικούς και να δούμε τι θα γίνει με το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο για να σημειώσουμε κάποια πρόοδο. Μα μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε αυτά τα καινοτόμα προγράμματα. Και τέλος, τέλος αλλά σημαντικό, ο κύριος Λόπεθ ανέφερε το τι γίνεται με την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας. Και εδώ παίζει και εδώ έχει σχέση το EU for Health. Θα ε, σας δώσουμε μία ανακοίνωση τις επόμενες εβδομάδες. Όλοι, όλοι θίξατε ζητήματα που στο πρόγραμμά μας, στη δουλειά μας τα καλύπτουμε και συνεργαζόμαστε ε, να βρούμε μία στρατηγική ευρωπαϊκή για το εμβόλιο. Ακόμα κυκλοφορεί ανάμεσά μας ε, ο ιός. Κανείς δεν είναι ασφαλής, αν δεν είναι όλοι ασφαλείς. Ευχαριστώ για τη συζήτηση και προσβλέπω στην συνεργασία σε όλα επίπεδα με το Κοινοβούλιο για να μπορέσουμε να φέρουμε την αλλαγή που χρειάζεται. Thank you very much, Commissioner. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Τώρα για το Συμβούλιο, τελευταίος ομιλητής, ο ε, Αναπολίτης Υπουργός, κύριε Ρότ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί κύριοι και κυρίες. Ευχαριστώ για την εμπνευσμένη αυτή συζήτηση δεν μπορώ παρά να σας υποστηρίξω και τονίζω ο ιός δεν έχει διαβατήριο και δεν σταματά στα εθνικά σύνορα. Ανεξαρτήτως ιδεολογικών συζητήσεων πρέπει να φροντίσουμε να καταλάβουμε ότι δεν κλέβουμε τίποτα από κανέναν. Όλοι έχουμε το καθήκον να μεριμνήσουμε για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων. σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να οργανωθούμε ώστε σε αυτό τον παγκοσμιοποιημένο κόσμο μια πανδημία να μπορεί να αντιμετωπιστεί στο, από το δικό μας επίπεδο δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα κράτη και γιατί με απασχολεί τόσο πολύ βλέπω ότι εδώ συμφωνούμε σε πολλά θέματα πρώτον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει μια ποιοτική αρχή υγείας και να βοηθήσει για να έχουμε συστήματα υγείας αποτελεσματικά. Δεύτερον, χρειαζόμαστε φάρμακα και ε, ε, αγαθά που σχετίζονται με την υγεία περισσότερη ανεξαρτησία της Ευρώπης, λιγότερη εξαρτησία από τρίτα κράτη. Τρίτον, χρειαζόμαστε περισσότερη συζήτηση και συντονισμό και ανταλλαγή απόψεων. Για τι φοβηθήκαμε τόσο πολύ στην αρχή. Ε, έχουμε να μάθουμε ένας από τον άλλο και Φυσικά είναι σημαντικό και τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλουν ένα σαφές μήνυμα προς τους πολίτες ότι η υγιεινή και οι κανόνες αποστάσεων πρέπει να τηρούνται. Ναι, αγωνιζόμαστε για μια ελεύθερη Ευρώπη χωρίς σύνορα. Και αυτή η εποχή είναι εποχή διακοπών όπου πολλοί κόσμος ταξιδεύει και έτσι είναι σημαντικότερο από ποτέ να δώσουμε ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να όχι να φοβάστε αλλά να προσέχετε. Το εμβόλιο το οποίο ελπίζουμε να βρεθεί ελπίζουμε να βρει σύντομα η επιστήμη, η έρευνα, ελπίζουμε να το διαθέσουμε σε όλους. Δεν θέλουμε να αποκλείσουμε κανέναν. Και επίσης στόχος είναι να δείξουμε την ευθύνη μας, ε, να σταθούμε στο ύψος της ευθύνης μας και στον κόσμο και ε, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους γείτονες. Ανέκαθεν πίστευαν όλοι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ικανή να δράσει. Μόνο στα Δυτικά Βαλκάνια δώσαμε 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ για υποστήριξη της αντιμετώπισης της πανδημίας αποφασιστικά και εκτενώς. Εδώ μιλάμε για αλληλογγύη όχι μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και με τους γειτονές μας. Θα χαιρόμουν ιδιαίτερα αν καταφέρναμε να συμφωνήσουμε σύντομα η γερμανική ε, Προεδρία του Συμβουλίου είναι διαθέσιμη γι' αυτό, είναι έτοιμη γι' αυτό. Ε, χαίρομαι που θα συνεργαστούμε και που υπάρχουν σαφή σημάδια αλληλεγγύης για αυτό το σημαντικό θέμα που απασχολεί όλους τους ανθρώπους, ε, όλους τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και που έχει, ε, μας έχει θέσει περισσότερες απαιτήσει από ποτέ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Η συζήτηση κλείνει. Η ψηφοφορία για τις τροπολογίες θα λάβει χώρα αύριο και η τελική ψηφοφορία την Παρασκευή. Θα ολοκληρώσουμε στις 9.45 μετά από το τέλος της ε, ε, τελικής ε, ψηφοφορίας και θα ξαναρχίσουμε αύριο στις 9. Η ημερησία δεξιά έχει δημοσιευτεί και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.